Good afternoon, colleagues. I'm going to make... Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θα αρχίσω, διότι έχουμε δύο πολύ σημαντικά θέματα μετά από τα έξυπνα σύνορα και έχουμε καθυστερήσει. Ο εισηγητής θα είναι σε λίγο μαζί μας. Εάν λοιπόν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για την ημερήσια διάταξη, εγκρίνεται. Σημείο 1. Σημείο 2. Γλωσσικό καθεστώς. Υπάρχει διερμηνία στα γαλλικά, γερμανικά, ολλανδικά, αγγλικά, ελληνικά, σουηδικά, ισπανικά, ουγγρικά, πολωνικά, βουλγαρικά και ρουμάνικα. Οι συντονιστές ε, συμφώνησαν την επόμενη 5η 17 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο να προσθεθεί μια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας στο Στρασβούργο από τι 9.30 μέχρι τις 10 το πρωί έτσι ώστε να ψηφίσουμε το ε, κείμενο για τον ε, κανονισμό για τα δεδομένα. Οι συστάσεις των συντονιστών της 23ης Νοεμβρίου συμπεριλαμβάνονται στα έγγραφα της συνεδρίασης. Εγκρίνεται λοιπόν τις ανακοινώσεις. Περνάμε στο σημείο 3. Βρίσκεται ο συγγητής εδώ ή έρχεται τουλάχιστον. Τότε ας αρχίσουμε με την παρουσίαση του κυρίου Γκάρκοφ. Και αγαπητοί συνάδελφοι, κατά τη διάρκεια της τελευταίας νομοθετικής ε, περίοδου, οι συζητήσεις για τα έξυπνα σύνορα οδήγησαν στην απόφαση να ζητήσουμε μία μελέτη για τις τεχνικές ε, δυνατότητες που έχουμε για το έργο. Η μελέτη τελείωσε το 2014 και ένα πιλωτικό πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί το 2015. Αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ε, υπηρεσία Γιουλίσα και τώρα ο διευθυντής της κύριος Γκάρκοφ θα μας παρουσιάσει την έκθεση. Μαζί του θα είναι ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κύριο Ρόζενμπουργκ. Θα δώσουμε πρώτα το λόγο στον κύριο Γκάρκοφ, μετά στον κύριο Ρόζενμπουργκ και έπειτα στον εισηγητή, στην εισηγήτρια μάλλον, κυρία Φαγιόν, διότι ο κύριος Ντίας Δεμέρας δεν μπορεί να έρθει σήμερα. Κύριε Κάρκοφ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε έτσι ώστε να παρουσιάσω ενώπιόν σας τα τελικά αποτελέσματα του πιλωτικού προγράμματος της Γιουλίζα για τα εφή σύνορα. Πρέπει να σας πω ότι ε, Πραγματικά έχουμε καταβάλει προσπάθειες και αυτή η έρευνα βρίσκεται στα πλαίσια των, της προσπάθειας δημιουργίας ευφυών συνόρων. Ευελπιστούμε δε ότι αυτό το πολιτικό πρόγραμμα θα παρουσιάσει ε, μαρτυρίες αποτελεσματικές και αξιόπιστες σχετικά με την δυνατότητα χρήσης τεχνολογιών όσον αφορά ε, τους ταξιδιώτες που περνούν τα σύνορα. Θέλω να υπογραμμίσω ότι ε, πιστεύω στο πρόγραμμα αυτό ε, γιατί τα ε, επιτεύγματα στα οποία καταλήξαμε μέσω του πιλωτικού προγράμματος μας αφήνουν να ευελπιστούμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά έστω και αν αφορούν ε, όλα τα ε, σύνορα ε, και αφορούν βεβαίως και την διαχείριση των σύνορων και περαιτέρω γνώση των ταξιδιωτών. Μίσω τους στόχους του πιλωτικού προγράμματος. Πρώτον, να μελετηθούν μελετικές επιλογές βάσει μετρησίμων κριτηρίων και βάσει των στοιχείων που θα συλλέγονται να ε, βρεθούν, να διατυπωθούν οι πιο σωστές τεχνικές λύσεις οι οποίες θα διευκολύνουν τις διαδικασίες ε, ελέγχου των συνόρων και βεβαίως ε, όλα αυτά με διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων. Το ίδιο το πιλωτικό πρόγραμμα είναι ένα ιδιαίτερα περίπλοκο πρόγραμμα. Η ιδέα περιπλοκότητά του αποδεικνύεται και από το πεδίο εφαρμογής το οποίο βασίστηκε στην μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2014 ε, και σε 13 υποθέσεις εργασίας, έστω και αν ε, πρέπει να θεωρήσουμε ότι 78 ήταν στην ουσία οι υποθέσεις εργασίας γιατί έγιναν ε, σε πολλαπλά σημεία διέλευσης. Περισσότερες από 109 ερωτήσεις ε, απαντήθηκαν μέσω αυτής ε, της ε, έρευνας και μέσω δοκιμών επιτόπου. Οι 7 μήνες διήρκεσε η προσπάθεια με 12 κράτη-μέλη και 18 διαφορετικά σημεία περάσματος των συμμόρων πέρα πάνω από 350 συνοριοφύλακες άμεσα ενεπλάκησαν ε, στην διαδικασία των δοκιμών. Ε, ελέγξαμε περισσότερο από 58.000 τραξιδιώτες από 110 εθνικότητες σε εθελοντική βάση το ίδιο το πιλωτικό πρόγραμμα αναφέρθηκε σε δύο κεντρικά στοιχεία, ε, δύο μετρικά στοιχεία, δηλαδή ε, ε, τις δυνατότητες που υπάρχουν όσον αφορά την τεχνολογία για τις διαδικασίες μετρήσεων των συνόρων και είδαμε και τους λεγόμενους process accelerators, τους επιταχυντές δηλαδή, δηλαδή θηρίδες ABC και κιόσκια στο πιλωτικό πρόγραμμα η αντίληψη των ε, συμμετεχόντων των ταξιδιωτών ελήφθη βεβαίως υπόψη. Ε, ας δούμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις ε, δοκιμές οι οποίες σχετίζονται με τα βιομετρικά στοιχεία. Πρέπει να σας πω ότι ε, αναπτύχθηκαν σε σχεδόν όλα τα ε, ε, συνοριακά περάσματα, είτε χερσαία είτε θαλάσσια και με διάφορες εναλλαγές δηλαδή μιλήσαμε, είχαμε τέσσερα δακτυλικά αποτυπώματα, οχτώ, δέκα, απεικόνιση του προσώπου, καθώς επίσης και απεικόνηση της ήριδος. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι όλα τα βιομετρικά στοιχεία ε, ταυτοποιήθηκαν ε, ταυτόχρονα σε όλα τα ε, σύνορα. και αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ορισμένα ευφύη σύνορα θα πρέπει να ε, εναρμονίσουν όλα τα νέα στοιχεία της τεχνολογίας. Και στα τρία είδη συνόρων ε, μελετήσαμε την δυνατότητα χρήσης των ε, ABC gates καθώς επίσης και των κιοσκιών ε, θα επαναλάβω και εδώ ότι όσον αφορά την υπηρεσία μας, τα αποτελέσματα ε, του πιλωτικού προγράμματος είναι αρκετά ικανοποιητικά ε, και έχουν τη δυνατότητα να μας δώσουν μια συνοπτική συνολική εικόνα όσον αφορά στην δυνατότητα χρήσης νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση των συνόρων. Ας δούμε τώρα μερικές λεπτομέρειες. Πρώτα απ' όλα τα γενικά στοιχεία τα οποία προκύπτουν από το πιλωτικό πρόγραμμα. Από τη δική μας άποψη είναι πολύ σημαντικό αυτό, αφορά δηλαδή τον υψηλό βαθμό αποδοχής σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του πιλωτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες στον έλεγχο εκλήθησαν να δώσουν και την άποψή τους στο σχετικό feedback για το πώς αντελήφθησαν αυτήν την διαδικασία. Σε γενικές γραμμές λοιπόν η αντίδραση ήταν θετική. Ε, ήρθαν σε επαφή με πολύ ικανοποιητικό τρόπο με την νέα τεχνολογία. Ε, επίσης και από την πλευρά των σύνοριοφυλάκων ε, είχαμε θετική αντίδραση. Η γενική θέση ήταν ότι μπορεί να διευκολυνθεί αυξηθεί αποτελεσματικότητα και να υπάρξει προστιθέμενη αξία και από πλευράς των συνοριοφυλάκων. Άλλα ευρήματα όσον αφορά ε, την χρήση νέων τεχνολογιών που είναι πολύ ενθαρρυντικά είναι τα εξής ε, μεγαλύτερη ορατότητα, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη χρήση των βιομετρικών ταυτοποιητών ε, και μεγαλύτερη ευκολία στη διαδικασία περάσματος των συνόρων έχει επιβεβαιωθεί. Το πιλωτικό πρόγραμμα ταυτοποιήθηκαν επίσης και κάποια, κάποιες γενικές ε, προκλήσεις ε, σχετικά με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν. Πρώτον, ε, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχουν ε, συγκεκριμένα πρότυπα και ε, ε, αποδεκτά όρια όσον αφορά τα, τους βιομετρικούς ταυτοποιητές. Δεύτερον, ότι υπήρξαν διαφορές στην απόδοση των μηχανημάτων ε, δηλαδή σε μία περίπτωση το μηχάνημα μπορούσε να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά σε, ε, ε, σε σύνορα εναέρια, ενώ σε χερσαία σύνορα ανάμεσα ας πούμε στη Ρωσία και την Φιλανδία δεν λειτουργούσε πλέον, δεν είχε την ίδια καλή απόδοση. Όσον αφορά τώρα την εμπειρία πολιτών τρίτων χωρών, και εδώ διαπιστώσαμε ε, λήψεις όσον αφορά την ανταλλαγή στοιχείων και προτύπων, ε, κυρίως όταν μιλάμε για τα ε, στοιχεία των διαβατηρίων. Είχαμε ιδιαίτερες δυσκολίες να περάσουν από Gates ABC οι κάτοχοι διαβατηρίων Κίνας και Βραζιλίας. Όσον αφορά τα, τις ε, βιομετρικές ε, συσκευές, ε, βρήκαμε ότι δεν υπάρχουν κοινά πρότυπα ποιότητας όσον αφορά την απόδοση και το αποτέλεσμα στο οποίο θα πρέπει να φτάνουν αυτές οι συσκευές. Ανάλογα δηλαδή με το είδος των συνόρων και στους σαρωτές είδαμε διαφορές ε, ενδεχομένως λοιπόν μπορεί να υπάρξουν κάποιες ε, διαφορές ε, όσον αφορά την απόδοση των σαρωτών αλλά βεβαίως αυτό δεν μπορεί να επηρεάσει συνολικά την προσπάθεια. Ας βούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τις, τα συμπεράσματα για τα βιομητρικά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά τα δακτυλικά αποτυπώματα ευρέθη ότι είναι δυνατόν να έχουμε καλά, καλής ποιότητας αποτελέσματα για σειρές 4, 8 ή 10 δακτυλικών αποτυπωμάτων και στα τρία είδη των συνόρων. Ωστόσο πρέπει να αναφέρουμε ότι ε, για τις περιπτώσεις σε 8 και 10 ε, ε, δακτυλικών αποτυπωμάτων μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες και βεβαίως ε, χρειάζεται επιπλέον χρόνος έτσι ώστε να έχουμε σειρές 8 ή 10 δακτυλικών αποτυπωμάτων. Ας πούμε για 8 δακτυλικά αποτελέσματα σε σχέση με σετ 4 χρειάζεται διπλός χρόνος, ενώ για σειρές 10 ε, δακτυλικών αποτυπωμάτων χρειάζεται τριπλός χρόνος από ό,τι για σειρές 4. Επίσης, όσον αφορά την οριμότητα της τεχνολογίας και των συσκευών, οι συσκευές ε, που χρησιμοποιούνται για σειρέ τεσσάρων αποτυπωμάτων φαίνεται να είναι σε καλύτερο βαθμό οριμότητα από τις άλλες. Όσον αφορά τώρα την ε, ε, εικόνα του προσώπου και σε σχέση με την ταυτοποίηση των φωτογραφιών στα διαβατήρια, η διαδικασία είναι εύκολη και γρήγορη. Η ίδια η τεχνολογία είναι όριμη και διαθέσιμη. Ας πούμε, ε, με απλές ε, ε, web κάμερες είχαμε την δυνατότητα να έχουμε καλά αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ήδη η τεχνολογία, είναι αρκετά καλή, είναι σε ικανοποιητικό βαθμό προχωρημένη. Όσον αφορά τώρα το, τη σάρωση της Ήριδας, έχει αποδειχθεί στο πιλωτικό πρόγραμμα ότι είναι δυνατή από πλευράς τεχνολογίας. Ωστόσο υπάρχει μεγάλη διαφορά των και τις απόδοσής τους ανάλογα με το περιβάλλον και τις συνθήκες στις οποίες καλούνται να λειτουργήσουν. Από την πλευρά μας λοιπόν συμπεραίνομαι ότι αυτή η τεχνολογία δεν είναι αρκετά ε, προχωρημένη και αρκετά όρημη έτσι ώστε να δώσει τα ίδια αποτελέσματα σε όλα τα σύνορα. Όσον αφορά τώρα το χρονικό περιθώριο για την σάρωση της ήρωδος ε, είναι περίπου ίδια, ίδιο χρονικό διάστημα με τις άλλες δύο περιπτώσεις ελέγχου. Όσον αφορά τώρα τους process accelerators, τους επιταχυντές διαδικασίας, η χρήση ε, των ε, ABC gates για την έξοδο είναι δυνατή. Όσον αφορά τώρα τους ε, ABC Gates, λέω ότι τεχνικά, από τεχνικής απόψεως, είναι δυνατή η χρήση αυτών των ε, εξόδων και έχουν λειτουργήσει και μπορούν να λειτουργήσουν για όλους τους ε, πολίτες ή για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το feedback που είχαμε και από τους ταξιδιώτες και από τους συνοριοφύλακες που συμμετείχαν σε αυτήν την πιλωτική διαδικασία είναι θετική. και επίσης ε, ε, τεχνικά είναι δυνατό να ελέγξουμε ε, όλα τα στοιχεία τα οποία περιέχονται στο τσίπ του διαβατηρίου. Ε, απ' την άλλη πλευρά βεβαίως, μόνο εάν υπάρχει σωστή ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων από αυτά που βρίσκονται μέσα στο διαβατήριο μπορούμε να προχωρήσουμε. Όσον αφορά τα κιόσκια τώρα, για την ε, καταγραφή βιομετρικών στοιχείων και αυτό είναι ε, δυνατό από τεχνικής ε, απόψεως. Χρησιμοποιήθηκε και ελέγχθηκε στο πιλωτικό πρόγραμμα. Όσον αφορά τώρα την, τον χρόνο με χρήση των κιόσκς, σύμφωνα με την, ε, με την πιλωτική μας ε, μελέτη φαίνεται ότι μπορούν να, υπάρχουν, να υπάρξουν ε, βελτιώσεις χρονικά της διαδικασίας με τη χρήση αυτού. Επίσης είναι σαφές και προκύπτει από το πιλωτικό πρόγραμμα ότι ενδεχομένως στη διάρκεια της διαδικασίας οι ταξιδιώτες θα χρησιμοποιήσουν, θα, θα χρειαστούν βοήθεια. Just, just to, Και για να ολοκληρώσω μπορώ να σας πω ότι ε, οι δυνατότητες, η ασφάλεια και η αξιοπιστία των τεχνικών μεθόδων έχουν επιβεβαιωθεί. Η χρήση των βιομετρικών ταυτοποιητών για την επαλήθευση της ταυτότητας των ταξιδιωτών και την ταυτοποίηση των ταξιδιωτών που δεν έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα είναι ικανοποιητική. Βεβαίως υπάρχουν ε, ε, ε, προβλήματα ας πούμε σε περίπτωση χρήσης κινητών διαδικασιών ας πούμε χρήση μετρητών βιομετρικών στοιχείων του προσώπου μέσα σε τρένα αλλά εν πάση περιπτώσει σε γενικές γραμμές το συμπέρασμα είναι θετικό και καταλήγουμε ότι υπάρχει τεχνική δυνατότητα. Ε, Επίση, με τον ίδιο τρόπο επιβεβαιώνεται και η χρήση των επιταχυντών. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο αντίκτυπος στο πέρασμα των ε, συνόρων έχει καθοριστεί και είναι, σε, ε, είναι θετικό βάσει μετρήσιμων μεθόδων. Και ε, ε, ε, σύμφωνα με το πιλωτικό πρόγραμμα κάτω από 30 δεύτερα διαρκεί ή ο έλεγχος και θεωρούμε ότι αυτή είναι μια καλή διαδικασία και μια καλή επίδοση για, την, για το πέρασμα των συνόρων. Δύο σημαντικά στοιχεία δύο σημαντικά ευρήματα. Πρώτον, είναι πολύ σημαντικό, τα τεχνικά, είναι πολύ σημαντική η τεχνική ε, παρουσίαση των ε, μηχανημάτων ε, και για τα βιομετρικά στοιχεία ε, είναι σημαντικό να έχουμε ε, δυνατότητα γρήγορης, ε, γρήγορης και επίσης και από πλευράς των συνοριοφυλάκων έχουμε πολύ θετικά στοιχεία, θεωρούν ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία και ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν με ικανοποιητικό τρόπο αυτές τις δυνατότητες. τώρα, ο συνδυασμός των βιομετρικών στοιχείων ε, έχει ταυτοποιηθεί και έχει ελεγχθεί ως επιτεύξιμος και ε, ε, δυνάμει αποτελεσματικός, έτσι ώστε να επιτευχθούν τα μέγιστα, τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα και να υπάρχει η μέγιστη αποτελεσματικότητα στη διαδικασία διέλευσης των συνόρων. Θα αναφέρω... Θα αναφέρω κάτι σημαντικό όσον αφορά τα πιλωτικά σχέδια είναι σημαντικό να αναφέρουμε εδώ ότι με το EU Visa έχουμε και εργασία υπό τα πιλωτικά υπό ένα άλλο πρίσμα της τεχνολογίας σε σχέση με την πιθανή επίπτωση αυτών των μεθόδων και υπάρχουν αρκετά ευρήματα ως αφορά τους στόχους. Στόχος ήταν η μελέτη παράλληλα με το έργο στο πιλωτικό επίπεδο για να εκτιμήσουμε τη στάση και την πείρα από πλευράς χρήσης βιομετρικών στοιχείων και τεχνολογίας όσον αφορά και το πόσο, κατά πόσο συνάδουν με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και βλέπουμε εδώ ότι έχουμε περίπου 1234 στις ε, παληθεύσεις με τους σταθμούς που καλύφθηκαν 50% άνδρες γυναίκες ισόρροπη λοιπόν σύνθεση όσον αφορά τους ταξιδιώτες και τους πολίτες. Αποτελέσματα, κύρια συμπεράσματα, η λεπτομερής έκθεση που θα αποτελεί τμήμα και είναι τμήμα της συνολικής έκθεσης πιλωτικής ε, ε, εμπειρίας. Η χρήση των βιομετρικών στοιχείων δείχνει ότι Υπάρχουν κάποιοι συμβιβασμοί που πρέπει να επιτυγχάνονται και η δακτυλοσκόπηση θεωρείται λιγότερο παρεμβατική μέθοδος σε σχέση με την, ε, την ε, αποτύπωση της ήριδας ε, για παράδειγμα και ναι φυσικά έχετε δίκιο τελευταία διαφάνεια και έτσι ολοκληρώνω την παρέμβασή μου και πάλι να τονίσω ότι σε σχέση με τους φορείς και τα όργανα έχουμε σημαντικό input για τα ΕΦΗ σύνορα σε σχέση με τη διαχείρισή τους με βάση αυτή την πρόταση. Και σε σχέση με τη μελέτη που συντάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρυσι παρέχονται αρκετά στοιχεία για το κατά πόσον είναι εφικτά τεχνολογικά αυτά τα, στόχη Είναι εφικτή. Σας ευχαριστούμε. Πρωτού περάσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέγει ο Πρόεδρος, να δούμε σε σχέση με το αν υπάρχουν μέλη ευρωβουλευτές που θα ήθελαν να παρέμβουν. Μάλιστα. Τρεις. Λοιπόν, εσείς οι τρεις. Άλλοι. Άλλοι. Κανείς άλλος δεν ζητεί να παρέμβει. Τρία μέλη, τρεις ευρω... τέσσερις ευρωβουλευτές. Άλλοι πάνω από τέσσερις, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτό το σημείο στις και 45. Τέσσερις ευρωβουλευτές, ευρωβουλευτές, κανείς άλλος δεν ζητεί να παρέμβει. Λοιπόν, συνάδελφοι, να είσαστε λογικοί και να είσαστε σύντομοι ώστε να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε και με τον κύριο Ρόζενμπεργκ φυσικά από την Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα είμαι πράγματι σύντομος να υπενθυμίσω ότι αυτό το πιλωτικό σχέδιο ήταν μια προσέγγιση που ξεκίνησε το 2014 σαν αντίδραση σε ερωτήσεις και αμφιβολίες που υπήρχαν και στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για κάποιες πτυχές της πρότασης του 2013 για τα ευφυή σύνορα. Ο στόχος ε, του συνολικού εγχειρήματο ήταν να υπάρξει έλεγχος και να υπάρξει επανεξέταση κάποιων από τα στοιχεία που βρίσκονται σε αυτή, βρισκόντουσαν σε αυτές τις προτάσεις. Πρώτο προϊόν, πρώτο αποτέλεσμα ήταν αυτή η μελέτη όπως προαναφέρθηκε Οκτωβρίου πέρυσι και δεύτερο προϊόν, υποπροϊόν ή τελευταίο προϊόν είναι αυτή η έκθεση για την φάση των δοκιμών. Η φάση δοκιμών με βάση τη συμφωνία που υπήρξε μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Ιουλίσα με την ε, έκθεση που ε, ετέθησε στη διάθεσή σας την προηγούμενη εβδομάδα με την εξέταση που έγινε ήταν μια πολύ καλή μελέτη μπορούμε να πούμε σε σχέση με την συμφωνία Μπορούμε να συγχαρούμε λοιπόν την Ιουλίζα για αυτή την πολύ επιτυχή μελέτη και έκβαση, την χωρίς προηγούμενο δηλαδή αυτή δοκιμασία και σε σχέση με τα κράτη-μέλη και τη συνεισφορά που υπήρξε ιδιαίτερες ευχαριστίες και όσον αφορά την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Οργανισμό για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο εντάχθηκε στη συζήτηση των νέων προτάσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει τα συμπεράσματα και τις παρατηρήσεις ε, της έκθεσης που ε, καλώς τεκμηριωμένες ε, οι τοποθετήσεις δίνουν μια πιστική απάντηση, μια πιστική συνεισφορά στα όσα τεκταίνονται μεταξύ του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Πρέπει να υπογραμμίσουμε όμως ότι αυτή η έκθεση φυσικά είναι μια αυστηρά τεχνικού χαρακτήρα έκθεση. Δεν μπορούσε να απαιτήσει κανείς κάτι παραπάνω. Τεχνικού χαρακτήρα έκθεση. Καταδεικνύει τι είναι εφικτό, τι μπορεί να λειτουργήσει και τι όχι. Τι είναι εποφελές και χρήσιμο <coughs> Δεν είναι όμως ε, ένα πρότυπο ως πρόταση για το πώς τα σύνορα θα έπρεπε να τα διαχειριζόμαστε μελλοντικά. Για να συμπληρωθεί αυτή η τεχνικού χαρακτήρα ανάλυση πρέπει να προσθεθούν άλλα στοιχεία νομικού χαρακτήρα, οικονομικού, πολιτικού, και πρέπει επίσης να σημειώσουμε και άλλες ε, πτυχές όπως την αρχιτεκτονική δομή του συστήματος ε, και την αποθήκευση δεδομένων και την πιθανή ακριβώς πρόσβαση που θα έχουν οι υπηρεσίες, ε, οι διοκτικές αρχές, αστυνομικές αρχές σε όλα αυτά τα στοιχεία. Συντάσσουμε λοιπόν για την αναθεωρημένη αυτή μορφή προτάσεων θα υπάρξει η σύνοψη αυτή, μια συνολική σύνθεση για την διαχείριση ευφυή διαχείριση των συνόρων υπό όλε αυτέ τι πτυχέ. Όπω προαναγγέλθηκε από πλευρά Επιτροπή, νο, ε, αναθεωρημένε νομικέ προτάσει στι αρχέ του 2016 πιθανότατα κατά το Μάρτιο θα σα διανεμηθούν. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε που είσαστε τόσο σύντομο. Τάνια Φαζόν. Και από πλευρά σα ως εισηγήτρια ίσως θα μπορούσατε να παρέμβετε και μας πείτε κάτι. Ευχαριστώ Πρόεδρε και φυσικά ευχαριστούμε και τον ε, εκπρόσωπο της Ιουλίζα για την επεξήγηση και μάλιστα με εξειδίκευση και εξειδικευμένο τρόπο για τα πιλωτικά αυτά προγράμματα και τα αποτελέσματά τους. Κάποιες ερωτήσεις θα είχα. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι είναι πολύ θετικό ότι έχουμε αυτό, όχι μόνο αυτή τη μελέτη κατά την έναρξη του έτους, αλλά και θα έχουμε και την ε, ε, αξιολόγηση διότι τα αποτελέσματα σαφώς καταδεικνύουν ότι οι αρχικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για παράδειγμα για τη δακτυλοσκόπηση δημιουργούσαν ε, προβλήματα αρχικά. Τώρα είναι μια πολύ σημαντική φάση απόφασης αυτή για την επίλεξη των στόχων του προγράμματος και για την επιλογή των βιομετρικών στοιχείων. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα για τη δακτυλοσκόπηση, τα δακτυλικά αποτυπώματα. Θα ήθελα να μας δίνατε κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Έχουμε σε σχέση με τα αποτελέσματα αυτού του πιλωτικού εγχειρήματος, το εξή. Ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία δακτυλοσκόπησης ε, είναι χρονοβόρα αυτή η φάση είναι πολύ, θα έλεγα, συντομότερη η πρώτη φάση από τη δακτυλοσκόπηση. Η διάρκεια σε σχέση με την δακτυλοσκόπηση είναι κάτω από 30 δευτερόλεπτα. Σε διάφορα σενάρια είχαμε και παραπάνω από 30 δευτερόλεπτα. Εσείς όμως προτείνετε και το συνδυασμό αμφωτέρων. Η ανησυχία είναι ότι θα έπαιρνε περισσότερο χρόνο στα σύνορα αυτή η διαδικασία αντί του στόχου που είναι ένας από τους στόχους της πρότασης των ευφυών σύνορων να διευκολύνουμε μια διαδικασία που θα δίνει τη δυνατότητα σε ταξιδιώτες να περνούν τα σύνορα σε μικρότερο χρονικό διάστημα, ταχύτερα δηλαδή Ποια ήταν ε, τα βιώματά σας ε, σε σχέση με ε, όσους είχατε συνεργαστεί με αυτούς. Από ό,τι γνωρίζω πολλοί θεωρούν ότι η δακτυλοσκόπηση είναι μια ιδιαίτερα παρεμβατική μέθοδος που μ, ίσως παρισφρέει στον ιδιωτικό ακριβώς χώρο ε, της ζωής των πολιτών και τι μπορεί να γίνει και τι θα μπορούσε να συμβεί αν απαιτήμα διότι για τους επιβάτες στα σύνορα δεν έχουν κάποια δικαιώματα να δράσουν ή να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Υπάρχει και γλωσσικός φραγμός. Ε, ε, αν δεν υπάρξει αναγνώριση αυτών των στοιχείων δεν θα μπορούν να περάσουν τα σύνορα και δεν θα έχουν κάποια δικαιώματα τα οποία θα έπρεπε να διασφαλίζονται για αυτούς. Έχοντας κάποια πιλωτικά τέτοια προγράμματα στην Φιλανδία και αλλού, είδαμε ότι είναι πολύ δύσκολο σε σχέση με τις τεχνολογίες, τεχνολογικές δυνατότητες δεν πάνε όλα τόσο στρωτά και γρήγορα όπως θα έπρεπε. Βέβαια στην πρώτη φάση υπάρχουν τέτοιες καθυστερήσεις, αλλά αν κάτι αποτύχει και δεν πάει καλά, αν πάει κάτι στραβά, τι γίνεται. Πολλές ανησυχίες υπάρχουν για το τι θα συνέβαινε σε σχέση με τέτοιους επιβάτες, με τέτοιους ταξιδιώτες. Αυτή θα ήταν η πρώτη μου ερώτηση ή παρατήρηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Τάνια. Κυρία Χολμάιρε, το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ντεκάρκοφ για αυτήν την εξαιρετικά καλή και λεπτομερή έκθεση. Μου φαίνεται πως είναι σαφές πως η εμπειρία σας αποτελείται κυρίως από, από τα αναγνωριστικά στοιχεία του προσώπου και είχατε την ευκαιρία να τα δοκιμάσετε σε πολλές ε, περιπτώσεις. Από ό,τι όμως ε, καταλαβαίνω και από αυτά που είπε και η Τάνια Φαγιόν, το σημείο, ε, το δύσκολο σημείο είναι όταν θα μου ζητούν οι αρχές να δείχνω το διαβατήριό μου αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ίσως ε, σίγουρα το έχετε ε, ζήσει και εσείς όταν δοκιμαζόταν αυτό το σύστημα, όμως... Ε, Έχω παρατηρήσει και εγώ καθυστερήσεις γενικότερα, δυσκολίες στην ε, συσκευή να διαβάσει τα στοιχεία. Σε αντίθεση με, άλλες, ε, με άλλα κιόσια όπου μου ζητήθηκε η ταυτότητά μου και μετά έπρεπε να ε, την κοιτάξουν και να δουν αν είμαι εγώ κτλ. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα είναι κάτι τεχνικό. Θεωρείται ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα μπορούν να ακολουθήσουν τις εξελίξεις της ε, τεχνολογίας. Αν ας πούμε εφαρμοζόταν αύριο και όλα σε το σύστημα των ε, έξυπνων ε, συνόρων μπορεί να επιταχυνθεί κάπως η διαδικασία και στα χερσαία σύνορα. Πώς λειτουργεί ακριβώς αυτό το σύστημα με τα δακτυλικά αποτυπώματα. Οι επιβάτες δηλαδή τι θα κάνουν, θα πρέπει να βγαίνουν από το όχημα, να σταματούν, ποιο είναι το σύστημα ε, το οποίο σας έδωσε τα καλύτερα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια των δοκιμών σας και σε σχέση με ε, την εφαρμογή. Μια ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είδαμε ε, μετά τα πρόσφατα γεγονότα στο Παρίσι ότι ακόμα και με την ταυτοποίηση των δακτυλικών αποτυπωμάτων οι τρομοκράτες δεν εντοπίστηκαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι προτίθεται να κάνει γι' αυτό, πώς θα το χειριστεί, γιατί είδαμε πόσο και η Eurodac δεν είχε μεγάλες ε, επιτυχίες, είχε και κάποιες δυσκολίες. Ακόμα και όταν τα δακτυλικά λοιπόν αποτυπώματα κάποιου είναι γνωστά, ενδέχεται αυτός να διαφύγει από τις αρχές. Πώς μπορούμε δηλαδή να αποτρέψουμε τέτοιες ε, περιπτώσεις. Αυτή η ερώτηση ήταν για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση και σχετικά με την ίδια του ματιού. Είναι εφικτή η τεχνολογία αυτή, τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο, διότι έχω την εντύπωση πως τα αποτελέσματα στα χερσαία σύνορα ήταν κάπως προβληματικά. Θα μπορούσατε ίσως ε, να ε, μου πείτε κάτι παραπάνω για την τεχνολογική διάσταση του θέματος αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Γκάρκοφ για την παρουσίασή του. Και μου έκανε εντύπωση μάλιστα το πόσο ενθουσιασμό δείξατε για αυτό το σύστημα των ευθειών συνόρων. Πρέπει να πω ότι για μένα και την πολιτική μου ομάδα υπάρχουν κάποιες ε, δυσκολίες στο να αποδεχτούμε αυτό το σύστημα, παρότι γνωρίζουμε ότι η κατάσταση δείχνει πως πρέπει να βελτιώσουμε την διαχείριση των εξωτερικών μας συνόρων. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να γίνει εις βάρος των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω ε, για το ότι συμπεριλάβατε την ε, μελέτη της Υπηρεσίας ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και με χαρά άκουσα πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη τα ευρήματα της υπηρεσίας. Και εδώ έχω και μία ερώτηση. Εκφράστηκε ο φόβος σε αυτό το άρθρο που διαβάζω σχετικά με την διόρθωση των προσωπικών δεδομένων. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν είναι κάτι που μπορούμε να επιλέξουμε... που μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Είναι θεμελιώδες δικαίωμα, είναι αδιαπραγμάτευτο. Και υπάρχει λοιπόν αυτός ο φόβος ότι δεν θα μπορούν να γίνουν διορθώσεις ή τροποποιήσεις στα προσωπικά δεδομένα των πολιτών εάν χρειάζεται. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Βαρζιά έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Κορπούς επανειλημμένα ε, έχω ακούσει παρουσιάσεις ε, των συμπερασμάτων της ε, μελέτης και μου φαίνονται πολύ λογικά αυτά που λέει. Είναι όντως πρόκειται για μια τεχνική μελέτη και την παρουσιάσετε με αρκετά ισορροπημένο τρόπο, έστω και αν έχετε δείξει μάλλον υπερβολική αισιοδοξία στο τέλος. Ε, ε, είναι γεγονός ότι ε, υπάρχει δυσκολία όσον αφορά ειδικά τα πολλαπλά σετ δακτυλικών αποτυπωμάτων. Αναρωτιέμαι όμως εάν ορισμένα στοιχεία της ανάλυσής όταν μας λέτε ότι ε, χρειάζεται διπλός χρόνος για σετ τεσσάρων δακτυλικών αποτυπωμάτων ε, σε σχέση με τέσσερα ε, μου φαίνεται λογικό, δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να γίνει μελέτη για να διαπιστώσουμε κάτι τέτοιο. Επίσης προβληματίζομαι λίγο όσον αφορά την διαφορά ανάμεσα στον χρόνο χρήσης Ε, μάλλον τον χρόνο ανάπτυξης και τον χρόνο κατά τον οποίο θα είναι πλήρως λειτουργικό το σύστημα. Επίσης, στρεφόμενοι κυρίως προς την Κομισιόν και όχι σε εσά, ε, προβληματίζομαι λίγο σε σχέση με την διασύνδεση με άλλους υφιστάμενους τρόπους ελέγχους, ελέγχων των συνόρων. Η κυρία Χολμάγερ, ε, δεν ξέρω γιατί αναφέρθηκε στους τρομοκράτες του Παρισιού, δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει με τα e σύνορα και κάποιες άλλες ε, ερωτήσεις. Ε, η μελέτη σας έγινε σε εθελοντική βάση, δηλαδή όλοι όσοι συμμετείχαν και έδωσαν την άποψή τους ήταν ε, εθελοντές. Μελετήσατε την άποψη που, αυτών που δεν θέλησαν να συμμετάσχουν και γιατί δεν θέλησαν να συμμετάσχουν. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναρωτηθούμε γιατί αρνήθηκαν κάποιοι να συμμετάσχουν. Επίσης, μας λέτε ότι σε γενικές γραμμές ε, οι πολίτες τρίτων χωρών δεν αντιτίθενται στο σύστημα όταν ε, ερωτώνται. Έχουμε ταξιδέψει πολύ σε τρίτες χώρες και ξέρουμε ότι και αντίστοιχα συστήματα υπάρχουν σε αυτές τις χώρες. Κάνατε μελέτη αναεθνικότητα γιατί υπάρχουν εθνικότητες που γνωρίζουν ήδη αυτά τα συστήματα και άλλες που ενδεχομένως δεν τα γνωρίζουν. Αυτό θα ήταν ενδιαφέρον γιατί εδώ έχουμε μία ανάλυση η οποία δεν είναι πολύ σαφής κατά την άποψή μου. Ερωτώ λοιπόν σε σχέση με ε, τους ανθρώπους που ερωτήσατε ε, κάνατε μία κατανομή αναεθνικότητα γιατί ενδεχομένως εκεί ε, θα είχαμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Ευχαριστώ. E, Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω θερμά για αυτή την εισήγηση, την παρουσίαση του κύριου Γκάρκοφ. Από ό,τι κατανόησα, το σύστημα της διαχείρισης, FES σύστημα διαχείρισης συνόρων, σε αυτή τη φάση, δοκιμαστική φάση, ουσιαστικά δεν σκοπεύει, δεν στοχεύει στο να δυσχεράνει τη ζωή των ταξιδιωτών, δεν πρόκειται για πιο χρονοβόρα διάβαση σύνορων, ούτε και πρόκειται να δημιουργηθούν προβλήματα με ε, δημιουργία δυσκολιών. Το αντίθετο, αυτό το σύστημα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά πρώτο λόγο για την ταυτοποίηση προσώπων, ατόμων, που υπάρχει υποψία ότι μπορεί να εμπλέκονται σε ποινικέ πράξεις και πρόκειται και για τους υπόπτους ε, τρομοκρατίας ή τρομοκρατικών πράξεων για την αποκάλυψή τους. Πρόκειται λοιπόν όπως αναφέρθηκε από την κυρία Χόλμα για αυτή την ε, ειδική χρήση κατά πολέμηση της τρομοκρατίας. Έχω την εντύπωση ότι οι, ε, οι δυσκολίες που δημιουργούνται για τους ταξιδιώτες είναι κάτι το αποδεκτό και μπορούν να το δεχθούν όταν πιστούν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δημιουργηθεί μεγαλύτερη ασφάλεια για αυτούς τους ίδιους. Τώρα έχω μία ερώτηση που θα ήθελα να διατυπώσω. Είπατε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι σήμερα δεν υπάρχει μια ενιαία ποιοτική προδιαγραφή όσον αφορά πιθανές συσκευές ε, που χρησιμοποιούνται για τη δακτυλοσκόπηση ή για φωτογραφικές μηχανές που ε, λαμβάνουν, κάνουν τις φωτογραφίσεις ε, δεν υπάρχει κάποια ενιαία, ένα ενιαίο πλαίσιο για συσκευές ή για την ποιότητα με βάση την οποία λειτουργούν αυτές οι συσκευές. Άρα λοιπόν είναι δύσκολο να αποφανθεί κανείς για, το, για τα πιστοποιητικά αυτά. Μία ερώτηση λοιπόν, όταν υπάρχουν τέτοιου είδους τεχνικού χαρακτήρες, τεχνικές διαδικασίες, είσαστε σε θέση να εκπονήσετε κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές που θα μπορούν και θα πρέπει να τηρούνται όσον αφορά την ποιότητα των στοιχείων που θα συλλέγονται μέσω αυτών των διαδικασιών. Αυτή είναι η ερώτηση. Ευχαριστώ διότι φυσικά θα μπορούσε υστερότερα στη στο έργο των περαιτέρω διατάξεων και κανονιστικών ρυθμίσεων να διαμορφώνεται ένα τέτοιο πλαίσιο. Τα όσα μας αναφέρατε είναι πολύ χρήσιμα και επικοδομητικά βέβαια, αλλά αυτό που αποκόμισα εγώ από την δική σας εισήγηση, από την δική σας έκθεση είναι ότι ουσιαστικά σήμερα ήδη τέσσερα αποτυπώματα ή και μία φωτογράφηση για την καλύτερη αποτύπωση της, ε, του προσώπου του χρήστη όπου οι συσκευές αυτή τη στιγμή δεν είναι ακριβώς οι πιο μ, τεχνικά όριμες ή αποτελεσματικές. Θα μπορούσατε για τη δακτυλοσκόπηση, για τα δακτυλικά αποτυπώματα και τις φωτογραφίες να μας πείτε ότι υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εκπονηθεί που θα μπορούν να ικανοποιούνται και να καλύπτονται ως προδιαγραφές σε όλα τα σύνορα ώστε να μπορεί να διευρυνθεί αυτό το πρόγραμμα και να τηρούνται αυτές οι προδιαγραφές μελλοντικά. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως ακούσαμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναμένουμε την έκθεση τον Μάρτιο του 2006 και σίγουρα θα συζητήσουμε διεξοδικά επ' αυτού. Ο κύριος Γκάρκοφ θα έρθει αρκετές φορές στην Επιτροπή μας, γι' αυτό λοιπόν αυτές τις ερωτήσεις θα έχουμε το χρόνο να τις απαντήσουμε αργότερα. Και σας λυπάμαι λιγάκι να πω, γιατί θα έχετε ένα σωρό ερωτήσεων να απαντήσετε. Επί της ουσίας, βέβαια, ε, δεν μας ε, φτάνει ο χρόνος και λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Γι' αυτό, λοιπόν, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να επιλέξετε μία ερώτηση, την οποία θέλετε να απαντήσετε και έχετε χρόνο ε, το πολύ τρία λεπτά για να την απαντήσετε. Δεν φταίτε εσείς, βέβαια, αλλά δεν προλαβαίνουμε μπορείτε να απαντήσετε. Κύριε Γκάρκοφ, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω με λίγα λόγια όλες τις ερωτήσεις μέσα σε αυτά τα τρία λεπτά. Τώρα, ε, σχετικά με την δακτυλοσκόπηση σε σχέση με την αναγνώριση προσώπου, γιατί το ένα και όχι το άλλο. Ε, η κυρία Χολμάιερ νομίζω έκανε μια σχετική ερώτηση. Ε, έχουμε την τεχνολογία. Και αυτή η τεχνολογία για βιομετρική αναγνώριση μας παρέχει περισσότερες δυνατότητες. Για παράδειγμα, κάποιο πρόσωπο που δεν μπορούμε να εντοπίσουμε μέσω των δακτυλικών αποτυπωμάτων, να τον αναγνωρίσουμε, με τη... τα βιομετρικά στοιχεία θα μπορέσουμε να το κάνουμε και θα αποφύγουμε τα λάθη στα σύνορα. Ε, τώρα, τι θα γίνει αν αποτύχει το σύστημα. Στα πλαίσια του πιλωτικού προγράμματος είχαμε μια ε, ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις εναλλακτικέ που έχουμε. Όχι μόνο για τα τεχνικά μέτρα ε, και όχι μόνο τι μπορούμε να κάνουμε για να συνεχίσει να λειτουργεί το σύστημα, αλλά και για άλλα προβλήματα επιτόπου στα σύνορα. Το, τα χερσαία σύνορα που μας έδωσαν και τα καλύτερα αποτελέσματα, μας έδειξαν ότι η τεχνολογία λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Το ερώτημα βέβαια είναι ποιες είναι οι συγκεκριμένες τεχνικές ελίξεις που θα εφαρμόσουμε στα χερσαία σύνορα, έτσι ώστε να διευκολύνουμε τους ταξιδιώτες να μην κάνουμε τη ζωή τους ε, δύσκολη. Σίγουρα δεν είναι όλα τα σύνορα τα ίδια. Τα σύνορα Φιλανδίας-Ρωσίας, ας πούμε, θα αντιμετωπίσουν περισσότερες δυσκολίες. Τώρα, αυτόματη διασταύρωση στοιχείων από διαφορετικέ βάσει δεδομένων. Θα ήθελα να σα καταστήσω σαφέ ότι το θέμα δεν είναι τεχνικό. Τεχνικά όλα γίνονται. Είναι πολιτικό το ζήτημα. Είναι κάτι που θέλει πολιτική βούληση και τη δημιουργία μέσων που θα διευκολύνουν την εφαρμογή των αποφάσεων. Ε, σάρωση της θηρίδας του ματιού. Δεν έχει οριμάσει ακόμα αυτό το σύστημα. Βρήκαμε πράγματι αρκετές δυσκολίε ιδιαίτερα από τους, ε, σε σχέση με τους ταξιδιώτες από την Ασία λόγω του σχήματος του οφθαλμού. Ε, είναι λοιπόν ε, κάτι το οποίο πρέπει να ε, μελετήσουμε παραπάνω και να περιμένουμε τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Τώρα, διόρθωση δεδομένων και πώς επηρεάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Δεν υπάρχει τεχνικά, επαναλαμβάνω, πρόβλημα. Το θέμα είναι ε, πώς η πρόταση κανονισμού για τα έξυπνα σύνορα θα το αντιμετωπίσει. Δεν βλέπω να υπάρχει τεχνικά κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα και φυσικά σέβομαι απόλυτα το δικαίωμα του κάθε πολίτη να ζητήσει διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων. Τώρα, επίκοη τρίτων χωρών και εθνικότητα. Ηθαγένεια. Όπως σας είπα από την αρχή, ένα από τα, ένας από τους στόχους του προγράμματος ήταν να εφαρμοστεί ε, πλήρως σεβόμενο απόλυτα ε, τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτικότητα του πολίτη. Γι' αυτό λοιπόν δεν συλλέξαμε στοιχεία όπως η υπηκότητα. Ωστόσο υπάρχει μια συμπληρωματική μελέτη η οποία παρέχει πληροφορίες ε, που αφορούν ακριβώς αυτό το θέμα. Θα επανέλθω λοιπόν σε αυτό. Τέλος, τα πρότυπα. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν πρότυπα για το βιομετρικό εξοπλισμό. Υπάρχουν και τα πρότυπα αυτά έχουν αναπτυχθεί κυρίως από τις Ηνωμένε Πολιτείες και οι συσκευές, τα σκάνερ, ε, οι σαρωτές της ίδιας ε, των βιομετρικών στοιχείων έχουν πιστοποιηθεί από τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα χρησιμοποιεί και το FBI, για παράδειγμα. Η προσωπική μου άποψη είναι ε, ότι ε, τα βιομετρικά στοιχεία και οι συσκευές αναγνώρισης βιομετρικών στοιχείων γίνονται ολαιόνα και σημαντικότερες ε, στον έλεγχο των συνόρων. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά στην Ευρώπη και πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι θα διαθέτουμε τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό. Αυτά και σε αυτά τα τρία λεπτά προσπάθησα να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ε, κύριε Γκάρκοφ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία μας είπατε και για τις απαντήσεις που δώσατε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν ξεκινήσουμε το επόμενο θέμα, ε, ε βλέπω ότι είναι πάρα πολύ οι όρθιοι στο πίσω μέρος της αιθούσης. Παρακαλώ λοιπόν να προσπαθήσετε να βρείτε κάποια θέση, να καθίσετε έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. if you're not sure where to sit down, then just, just seek some guidance and... Uh... αν δεν ξέρετε πού πρέπει να καθίσετε, παρακαλώ ζητήστε βοήθεια. So colleagues, please take your seats and we're going to start. Okay. So colleagues, one of the um, central... Αγαπητοί συνάδελφοι, ένας, ε, ο κεντρικ... ένας από τους ε, κεντρικούς ε, στόχους της και προθέσεις της σημερινής μας συνάντησης ήταν ε, το να μελετήσουμε την εφαρμογή του hot spots στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τα μέλη, ε, μερικά εκ των οποίων παρίστανται, ε, που ζήτησαν αυτήν την ενημέρωση και θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου τα οποία είναι παρόντα ε, και, που, ε, και όλους βεβαίως όσοι βρίσκονται εδώ για να μας βοηθήσουν να κάνουν τη δουλειά μας και να μας διαφωτίσουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ε, μαζί όλους τους κεντρικούς πρωταγωνιστές αυτών των σημείων, τους συντονιστές των hot spots, εκπροσώπους των μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με τα θέματα που σχετίζονται με τα hot spots. Πρώτα απ' όλα θα δούμε το θέμα των hot spots στην Ελλάδα και μετά στην Ιταλία. Ελπίζω πράγματι ότι αυτή η συνεδρίαση δεν θα είναι ε, μοναδική, ότι θα υπάρξουν ε, τακτικές ε, συνεδριάσεις παρακολούθησης της υλοποίησης των hot spots. Και βεβαίω, ε, μια και είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε, θα μεριμνήσω έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να έχουν την δυνατότητα να ε, μιλήσουν και επίσης να του υποβάλουμε ερωτήσεις και να έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν. Γι' αυτό παρακαλώ πολύ να είστε προσεκτικοί όλοι με το χρόνο σας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο τμήμα, το οποίο αφορά την Ελλάδα και θα δώσω ε, τον λόγο στον ε, ε, Μάρτιν Μπέρουε, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Home της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να σας μιλήσουμε για αυτό το σημαντικό θέμα. Απλώς για να αποσαφηνίσω τον ρόλο μου μέσα στο πλαίσιο αυτό που πριν από δύο μήνες ζητήθηκε από τον πρόεδρο να ηγηθώ του ρόλου του, των αρμοδιοτήτων από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα κομβικά σημεία υποδοχή, hotspots και όλα τα άλλα θέματα μετανάστευση στην Ελλάδα. Πρέπει να σα διορθώσω σε ένα θέμα. Δεν είμαι μέρο ε, υπάλληλο τη Γενική Διεύθυνση Home. Ωστόσο, εργάζομαι, συνεργάζομαι σε πάρα πολύ στενή σχέση με τους συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών GD Home μπορώ να πω ότι οι όροι και προϋποθέσεις υπό τους οποίους εργαζόμαστε στην Ελλάδα είναι προκλητικοί, είναι μια πρόκληση μπορεί κανείς να πει. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός αφήξεων επιπλέον σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες οικονομικές που βιώνει η χώρα και αν ένα τρίτο στοιχείο κάνει κανείς λόγο για το σύστημα διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών που υπήρχε στην Ελλάδα μπορεί κανείς να πει ότι δεν, είχε, δεν ήταν ιδιαίτερα προηγμένο ο συνδυασμός του μεγάλου αριθμού και λοιπόν και του παροχημένου συστήματος δημιουργούν τεράστιες προκλήσεις που πρέπει να υπερβούμε, να αντιμετωπίσουμε. Σε σχέση με τη συνεργασία και συζητήσεις με τις ελληνικές αρχές έχουμε επικεντρωθεί σε πέντε τομείς κυρίως όπου θεωρούμε ότι πρέπει να επιτευχθεί, να σημειωθεί πρόοδος πρώτον στον ρόλο των hotspots, δεύτερο το σύστημα επανεγκατάστασης πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί. Τρίτον, να μπορέσουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των επιστροφών για την βελτίωση της διαχείρισης συνόρων και φυσικά για να υπάρξουν και βελτιώσεις στο δυναμικό υποδοχής και ε, ποιοτικά και αριθμητικά. Θα ήθελα να σας δώσω πολύ σύντομα κάποια στοιχεία των κυριότερων εξελίξεων κατά τους τελευταίους δύο μήνες για τα hot spots πρώτον. Όπως γνωρίζετε πέντε νησιά έχουν καθοριστεί από τις ελληνικές αρχές για την τοποθέτηση ως αυτών των hot spots Λέρος, Κος, Λέσβος, Χίος, Σάμος και πρέπει να πούμε ότι από πλευράς λειτουργικής ε, η ε, δυνατότητα αυτής ε, της λειτουργίας hotspots σε άλλα σημεία γίνεται καταχώρηση αλλά δεν υπάρχει δομημένη αυτή η προσέγγιση που θα, θέλαμε εμείς να δούμε ότι θα μπορούσε να λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Οι ελληνικές αρχές αυτή τη στιγμή σχεδιάζουν, προγραμματίζουν να ξεκινήσουν οι εργασίες σε τρεις από αυτές τις πέντε νήσους Ακόμα αυτή την εβδομάδα θα υπάρξει επιβεβαίωση, επαλήθευση ότι στην ΚΟ, Λέσβο και Λέρο θα, θα λειτουργούν τα κέντρα αυτά και στόχος είναι να ακολουθήσει γοργά τον Ιανουάριο η Χίος και η Σάμος στην συνέχεια όπου πρέπει να αποσαφινιστούν κάποια πράγματα. Συνεργαζόμαστε με τις ελληνικές αρχές ώστε να βελτιστοποιηθούν οι ε, διαδικασίες για τη διαδικασία καταγραφής και της καταχώρησης ε, αυτών των ε, ατόμων των προσφύγων εκεί και από κοινού καταβάλουμε προσπάθειες με τους οργανισμούς σε ομάδες εργασίας επιτόπου ώστε συλλογικά να μπορέσουμε με τις προσπάθειές μας να βελτιώσουμε τα πράγματα για την επανεγκατάσταση σύντομα από ε, την Ελλάδα θα αναμέναμε αναμένουμε να αυξηθούν οι αριθμοί τις επόμενες εβδομάδες ε, των ε, όσων θα μετεγκατασταθούν. Υπάρχουν όμως στη στενοπή όσον αφορά τις, τη διάθεση, την προώθηση των διαδικασιών. Περισσότερα πρέπει και μπορούν να γίνουν και για την δυνατότητα επανεγκατάστασης ε, αναμένουμε με τα μέτρα τα οποία θα ακολουθήσουν στη συνέχεια να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Υπάρχει όμως ε, και <clears throat> πρόβλημα όσον αφορά τις, ε, το δυναμικό και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις επιστροφές ατόμων επιστροφές ατόμων που συναρτώνται επίσης και με τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές αρχές. Η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα παρέχοντας μεγαλύτερη συνδρομή στις ελληνικές αρχές ώστε με τη βάση αυτή να μπορέσει το πρόγραμμα να συνεχίσει να αναπτύσσεται. Βλέπουμε ότι υπάρχουν στενοποί όμως όσον αφορά τρίτες χώρες που σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι καθόλου πρόθυμες ε, να δεχθούν τους ε, ε, όσους επιστρέφουν ή όσους θα μετεγκατασταθούν πρέπει να γίνουν δεκτοί από τις χώρες αυτές. Κατά την τελευταία εβδομάδα είχαμε αξιωματούχους που είχαν αναπτύξει τις δραστηριότητές τους και που με άλλες εκατοντάδες θα αυξηθούν κατά τον Ιανουάριο οι ελληνικές αρχές έχουν καταλήξει σε μια συμφωνία με την Frontex για την πρόσθετη ε, δράση στα βόρεια σύνορα των αξιωματούχων αυτών ώστε να μπορέσει να υπάρξει καταγραφή των ε, ε, μεταναστών και προσφύγων στα βόρεια σύνορα καθώς επίσης και να υπάρξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Τώρα για την υποδοχή υπάρχουν κάποιες σημαντικές εξελίξεις ε, σε σχέση με αυτό το σκέλος. Έχουμε καταλήξει ουσιαστικά σε μια συμφωνία με την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες ώστε 20.000 θέσεις υποδοχής να μπορέσουν να αναπτυχθούν στην ε, χώρα αυτός ο αριθμός επιπλέον στις 4.500 θέσεις που έχουν προγραμματιστεί για τα τρία hot spots που προανέφερα και που κατά τα τέλη του έτους θα μπορούν να προσθεθούν στον αριθμό θέσεων για τα άτομα αυτά και έχουν ε, προγραμματιστεί ξεχνώ το όνομα της ε, τράπεζας ε, που θα ε, συνέδραμε. Βλέπουμε όμως 25.000 επιπλέον θέσεις θα δημιουργηθούν. Ολοκληρώνω εδώ την παρέμβασή μου και σας ευχαριστώ Πρόεδρος. Θα ήθελα να τηρείτε το χρονικό όριο γιατί θα υπάρξουν ερωτήσεις στη συνέχεια και θα πρέπει να μπορέσουμε οι ευρωβουλευτές να θέσουν τις ερωτήσεις τους. Από πλευράς του συντονιστή για τις hot spots η κυρία Καραγγελή παρακαλώ. Έχετε τον... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Hotspot λοιπόν στην Ελλάδα και ειδικά στη Λέσβο ή στη Μόρια όπως οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εσά θα το έχετε ακούσει. Ε, θα προσπαθήσω να είμαι αρκετά περιεκτική και σύντομη και στόχο είναι περισσότερο να δώσω το ένασμα για μια πολύ καλή κουβέντα που εγώ τουλάχιστον θα ένιωθα την ανάγκη ότι θέλω να κάνω μαζί σα. Πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ λιγάκι στι διασώσει και στι επιχειρήσει διάσωση πριν έρθουν οι άνθρωποι στη Μόρια ε, να περιγράψουμε λιγάκι το τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στο hot spot, ε, ποιες ακριβώς διαδικασίες είναι αυτές που ε, είναι στο στάδιο του improvement από μέρους της Ελλάδας, λίγες σκηνές και λίγες εικόνες για τη ζωή μέσα στο hot spot και κάποια ζητήματα τα οποία εγώ θεωρώ πολύ βασικά και θα ήθελα πάρα πολύ να τα συζητήσουμε. Ξεκινάω λοιπόν λέγοντα ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έρχονται ξαφνικά στο hot spot τη Μόρια. Έρχονται όπω βλέπετε στο χάρτη από τι ακτέ τη Τουρκία. Ε, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω πάρα πολλά κόκκινα βέλη για να δείξω σε ποια σημεία του νησιού έχουμε αφήξει προσφύγων και μεταναστών. Είναι όλη η βορειοανατολική έω και το κάτω μέρο του νησιού, νοτιοανατολική πλευρά. Και αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί έρχονται σε πάρα πολλά σημεία και πρέπει να μεταφερθούν στο hot spot τη Μόρια που βρίσκεται μέσα στο κίτρινο κύκλο, όπω όπως βλέπετε το χάρτη. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολλά σημεία εισόδου τα οποία εναλλάσσονται διαρκώς, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν πάρα πολλές ανάγκες για την ε, έρευνα και τη διάσωση, γεγονός που επιβαρύνει πολύ το ε, ελληνικό λιμενικό σώμα. Έρχονται λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί μέσα σε βάρκες που βλέπετε στην οθόνη. Ε, οι βάρκε είναι ε, πολύ συγκεκριμένε σε τύπο, είναι αυτού του τύπου, δεν έχουμε δει αλλού τύπου βάρκε στην Ελλάδα, με ελάχιστες Ε, είναι μέσα 40, 50, πολλέ φορέ και 60 άνθρωποι, γυναίκε, μωρά, παιδιά, ε, μεικτοί πληθυσμοί. Και εδώ είναι το δύσκολο σημείο για μα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε διαχωρισμό προσφύγων και μεταναστών όταν οι συνθήκε εισόδου των ανθρώπων είναι τέτοιε, όπω βλέπετε, είναι μέσα στη θάλασσα. Ε, και υπάρχει ο κίνδυνος ναυαγίου ακόμα και στα 10 μέτρα πολλές φορές ή 15 από την ακτή χωρίς υπερβολή. Το έχω ζήσει και μπορώ να σας το περιγράψω πάρα πολύ ε, ε με μπελανά σημεία αυτό το ε, σημείο γιατί βλέπετε είναι παιδιά τα οποία πολλές φορές είναι η πρώτη φορά που βλέπουν θάλασσα. Είναι άνθρωποι που πρώτη φορά βλέπουν θάλασσα και αυτό τους επιβαρύνει, τους φοβίζει και πανικοβάλλονται. Και επιπλέον, και εδώ θα τελειώσω με το κομμάτι της διάσωσης, οι άνθρωποι αυτοί έρχονται σε ε, όπου είναι δυσπρόσιτες. Είναι πολύ δύσκολο να έχουμε τη δυνατότητα είτε να έχουμε γιατρούς, είτε να έχουμε ασθενοφόρια ή ακόμα και λεωφορεία για τη δική τους μεταφορά. Πολλές φορές είναι αναγκασμένοι να περπατήσουν ολόκληρες πλαγιές. Είναι η γεωγραφία του νησιού τέτοια. Πολλές και πολλοί από εσάς νομίζω ότι έχετε επισκεφθεί το νησί και γνωρίζετε για το τι ακριβώς μιλάω. Πάρα αυτά όμως οι άνθρωποι εξακολουθούν να έρχονται. Και η Ελλάδα, ε, δεν ξέρω γιατί εδώ δεν φαίνονται τα νούμερα στη διαφάνεια, ε, ε, η Λέσβος με το κόκκινο χρώμα είναι αυτή που σηκώνει το βάρος των αφήξεων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ολόκληρη. Ε, δεν ξέρω γιατί δεν φαίνεται στη διαφάνεια τη που βλέπετε, ε, το νούμερο το οποίο είναι κυκλωμένο είναι 135.021 αφήξεις στη Λέσβο μόνο για το μήνα Οκτώβριο, αν μπορείτε να διακρίνετε. Και το θεωρώ πολύ σημαντικό γιατί είναι και ο μήνα που ξεκίνησαν πάρα πολλέ ή κορυφώθηκαν, για να είμαι πιο ακριβή, οι εργασίε μέσα, μέσα στο χώρο τη Μόρια. Για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα improvement στο accommodation κυρίω, διότι οι διαδικασίε καταγραφή οφείλω να πω ότι ήταν αυτέ που και τώρα με τι προδιαγραφέ των hotspot χρησιμοποιούμε. Τα νούμερα νομίζω ότι μιλάνε πολλές φορές καλύτερα από μόνα τους. Ε, είναι τα νούμερα τα συνολικά με τις αφήξεις στην Ελλάδα και είναι και τα νούμερα από κάτω με τη Λέσβο που φαίνεται ότι σηκώνει το βάρος αυτή τη στιγμή. Και εδώ είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από τη Λέσβο στο λιμάνι του Πειραιά και έχουν καταγραφεί ήδη. Τα ποσοστά τα οποία βλέπετε και εύχομαι να μπορείτε να διακρίνετε αυτή τη φορά είναι αναδιήμερο και αφορούν σε ανθρώπους που έχουν ταυτοποιηθεί με τις διαδικασίες ε, που προβλέπονται, ε, έχουν περάσει από όλες ε, τις διαδικασίες όπου και η Ελληνική Αστυνομία και η Frontex σε συνεργασία έχουν δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε να γίνονται και εδώ θα μου επιτρέψετε, όσο μπερδεμένο και να φαίνεται το σχεδιάγραμμα, να πω ότι είναι οι συνολικές καταγραφές που γίνονται στην Ελλάδα και οι συνολικές καταγραφές που γίνονται στη Λέσβο, που θα δείτε ότι σχεδόν αγγίζει το συνολικό ποσοστό. Και το λέω αυτό γιατί είναι αρκετά δύσκολο ε, και θεωρώ ότι είναι και αρκετά σπουδαίο ε, άνθρωποι οι οποίοι έρχονται με τον τρόπο που είδατε λίγο πριν να υπόκειται στη διαδικασία φυσικά της πρώτης υποδοχής, όπου η η για τους πρόσφυγες σε αυτό το σημείο δεν δίνει μια βαρύτητα στις ευάλωτες ομάδες και με τη βοήθεια και άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων για να ακολουθήσει η διαδικασία του screening και του debriefing σε συνεργασία με τη Frontex ε, η ελληνική αστυνομία της λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων με το σύστημα του Eurodac, η φωτογράφηση και φυσικά όλες οι απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες θα μπορέσουν ε, να οδηγήσουν στη χορήγηση του διοικητικού εγγράφου που είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε στη συνέχεια να μιλάμε για άσυλο και relocation, τη διαδικασία του ασύλου και του relocation, την οποία θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική και ίσως ότι έχουμε και πολλά να πούμε. Ε, ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολο να διακρίνεται αυτό το σχεδιάγραμμα είναι αυτό το οποίο ε, είναι ξεκάθαρη η διαδικασία για μας στην Ελλάδα που πρέπει να ακολουθεί για το relocation, αλλά επίσης νομίζω ότι είναι και αρκετά τα ζητήματα που καλό είναι να βελτιωθούν και να τα συζητήσουμε όλοι μαζί. Οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες και μπορώ να τα δώσω στα mail σας αν επιθυμείτε. Θα ήθελα όμω λιγάκι να δούμε τη διαδικασία των δακτυλικών αποτυπωμάτων με τα Eurodac μηχανήματα, γιατί όπω άκουσα και πριν, είναι μια διαδικασία που πράγματα απαιτεί χρόνο. Και σκεφτείτε ότι η ελληνική αστυνομία δουλεύει 24 ώρε το 24ωρο για να μπορεί να καταγράφει γρήγορα ανθρώπου, με όλες τις νόμιμες διαδικασίες να ε, γίνεται η λήψη των φωτογραφιών, να περνούν στο σύστημα του Eurodac και να έχουμε την τελική έκδοση των διοικητικών εγγράφων. Αυτό είναι κάτι που απαιτεί πάρα πολλές ώρες εργασίας και παρά ε, τους λίγους ανθρώπινους πόρους ή τους πολλούς που έχουμε προσπαθήσει το τελευταίο καιρό να έχουμε στα νησιά, καταλαβαίνετε ότι το φόρτο εργασία είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ε, τι προσπαθούμε αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη βελτιώσει, τουλάχιστον στο hot spot της Μόριας, τις θέσεις ε, για την ε, προσωρινή φιλοξενία. Ε, αυτή τη στιγμή μιλάμε για 1.000 με 1.100 θέσεις φιλοξενίας μέσα στο hotspot της Μόριας και αυτό το οποίο ε, προσπαθούμε είναι να δημιουργήσουμε δύο νέους σταθμούς ε, registration station ε, όπως τους ονομάζουμε, καταγραφής για να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα περισσότεροι άνθρωποι να περνούν και να καταγράφονται ε, την ίδια μέρα. Ε, το σχέδιο είναι για να δούμε λιγάκι τη μορφολογία μέσα της Μόριας οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή καταγράφονται σε δύο σταθμούς, τον πάνω αριστερά και τον κάτω δεξιά και μέσα στο τέλος της εβδομάδας θα έχει τελειώσει και η δημιουργία δύο νέων ε, σταθμών. Λίγες εικόνες από τα έργα τα οποία γινόντουσαν την προηγούμενη εβδομάδα και ολοκληρώνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται εργασίες μέσα στο χώρο. Ε, είναι ο χώρος για τους καινούριου σταθμούς ε, καταγραφής. Είναι σκηνές από τις προσπάθειες που γίναν για να βελτιωθούν οι συνθήκες ε, ε, και ο αριθμός του accommodation σε συνεργασία με την υπατερμοστία. Ε, φτάνουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυξημένες ανάγκες, θα έλεγα, όχι μόνο ε, σε επίπεδο ε, ρούχων που μπορεί να φανταστείτε, φανταστείτε αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και είναι βρεγμένοι και καλούμαστε εκείνη την ώρα να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση, αλλά έχουμε και ανθρώπους με αναπηρίες, με κινητικά προβλήματα, πολύ μωρά παιδιά, βρέφη που μπορεί να γεννήθηκαν λίγες ώρες πριν, ε, και σας το λέω με πλήρη ειλικρίνεια, έχω δει μωρό να γεννιέται στη βάρκα και να είμαι στην αυτή την ώρα που φτάνει και πολύ περισσότερο ανθρώπους θύματα βασανιστήριων με σημάδια πολλές φορές ζωγραφισμένα στο πρόσωπο. Ε, Παρά αυτά προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να δημιουργήσουμε και έχουμε δημιουργήσει τις συνθήκες για τη στήριξη ευάλωτων ε, κοινωνικά ομάδων όπως είναι γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες με τα παιδιά ή παιδιά ε, για χώρους δημιουργικής απασχόλησης μέσα ε, στη Μόρια για τον καιρό που θα φιλοξενηθούν. Και εδώ θα ήθελα να δώσουμε λίγο έμφαση κυνηγώντα το χρόνο ε, τίθονται κάποια ζητήματα. Ε, εύχομαι να πήραμε όλη μια ιδέα το τι γίνεται αυτή τη στιγμή μέσα στη Μόρια. Είναι όμως πολύ βασικό να πω ότι ε, προς το τέλος της εβδομάδας θα θέλαμε να έχουμε την ενίσχυση με τα Eurodac μηχανήματα που έχουμε ζητήσει, ε, όπως επίσης και κάποιο πρόσθετο προσωπικό από την Frontex. Και οφείλω να πω εδώ ότι και με τον ΕΑΣΟ έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Είναι, ε, ανταποκρίθηκε άμεσα στο έτοιμά μας για ε, στήριξη στις διαδικασίες του relocation αλλά παραμένει και για μένα και θα το μεταφέρω σαν άνθρωπο του πεδίου, παραμένει ένα ανοιχτό ζήτημα το οποίο έχω την αίσθηση ότι η γραφειοκρατία των Βρυξελών και η γραφειοκρατία της Ελλάδας μερικές φορές δεν βοηθάει και θα πρέπει λιγάκι να βοηθήσουμε ο καθένας από τη θέση του, έτσι ώστε ξέρω και άκουσα τι υπόθηκε λίγο πριν για τα χρήματα και για τις χρηματοδοτήσεις. Η Ελλάδα ξεκίνησε και ο μηχανισμός έχει ξεκινήσει να απορροφά κονδύλια. Παρ' όλα αυτά μένουν πολλά ζητήματα τα οποία νομίζω ότι είναι, ε, έχουν δυσκολίες και χρειαζόμαστε τη στήριξη, όπως είναι οι διερμηνείς, ε, και χαίρομαι που βλέπω και τον Ιταλό συνάδελφό μου γιατί πρόσφατα στη Μόρια μιλούσαμε και λέγαμε ότι μέσα στα hot spot ε, και 100 διερμηνεί να έχει πολλές φορές δεν σε φτάνουν για να μπορέσεις να κάνεις αποτελεσματικά τη δουλειά σου ε, και θα κλείσω γιατί βλέπω το χρόνο να περνάει λέγοντας ότι σαν άνθρωπος που θεωρώ ότι πολλές φορές είμαστε στην πρώτη γραμμή, δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε ε, τη λειτουργία αυτού του συστήματος που θέλουμε όλοι να δούμε, λειτουργεί του relocation, του ασύλου και όλες αυτές τις υποδομές των hot spots, χωρίς να λάβουμε υπόψη μας ότι η πόρτα ε, της Ευρώπης δεν είναι η Ελλάδα για αυτούς τους ανθρώπους. Η πόρτα βρίσκεται στην Τουρκία και άρα χρειάζεται να κάνουμε κάποιες συντονισμένες κινήσεις όλοι μαζί σαν ευρωπαϊκή οικογένεια ε, απέναντι σε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την υπομονή και το χρόνο που καταχράστηκα νομίζω κύριε Πρόεδρε. Okay, next is... Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριο Έμπρη από την ΕΑΣΟ τώρα θα λάβει το λόγο, θα μιλήσει για τρία λεπτά και σας παρακαλώ να κρατήσετε το ε, χρονοδιάγραμμα. Θα έχετε το χρόνο για απαντήσεις αργότερα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη μου χαρά ξαναβρίσκομαι εδώ ενώπιόν σα και θα είμαι σύντομο. Θα ήθελα να αναφέρω ορισμένα σημεία τα οποία αναφέρα και την περασμένη εβδομάδα που ήρθα εδώ για να σα ενημερώσω. Ε, είχαμε ζητήσει την γνώμη 274 επιπυρογνωμόνων και το λάβαμε απαντήσει από τους 176. Έχουμε λοιπόν μία ε, κατάσταση που θα σας παρουσιάσω αμέσως. Στην Ελλάδα έχουμε κάποια σχέδια επιχειρήσεων. Ένα από αυτά έχει υπογραφεί ήδη με την ελληνική κυβέρνηση και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διαδικασία αναθεώρησης έτσι ώστε να είμαστε πιο ευέλικτοι και να δούμε τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εστιάζουμε σε τρεις τομείς. Καταρχάς παροχή πληροφοριών για τα σημεία αποβίβασης όπου παρέχονται πληροφορίες για τη διαδικασία ε, ασύλου και μεταγκατάστασης. Έπειτα ε, επεξεργασία των ε, αιτήσεων και των κατάλληλων κρατών μελών που θα ε, δεχτούν την μεταγκατάσταση και, κατά τη και την διαδικασία καταγραφής. Αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούμαστε στην Ελέσβο. Έχουμε περίπου ε, 7 ε, υπαλλήλου που ε, βοηθούν στην παροχή πληροφοριών. Επίσης, τις προσεχείς ημέρες θα είμαστε στον Πειραιά και όσον αφορά την ε, διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων θα είμαστε έτοιμοι στις αρχές του 2016. Ο αριθμός του προσωπικού μας ενδεχομένως να αυξηθεί στους 20. Σχετικά με τα ταξιδιωτικά έγγραφα έχουμε δύο ε, εμπειρογνώμονες υπαλλήλους που εργάζονται για αυτόν τον σκοπό. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε στην ε, δημιουργία των άλλων hot και μία από τις εδράσεις που έχουμε αναλάβει με αυτόν τον σκοπό είναι η παροχή κινητών ε, γραφείων. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να παρέχουμε αυτές τις κινητές μονάδες έτσι ώστε να διευκολύνουμε την καταγραφή αλλά και την δημιουργία των ε, νέων hotspot. Η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε είναι η χωρητικότητα, ε, είναι η διαδικασία καταγραφής των ε, ετούντων άσυλο. Η ΕΑΣΟ έχει επαναλάβει την πρόθεσή της να βοηθήσει τις ελληνικές αρχές στη διαδικασία καταγραφής και αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με τις ελληνικές αρχές έτσι ώστε να είναι λειτουργικό το σύστημα το στομότερο δυνατόν. Αυτή τη στιγμή επικοινωνούμε επίσης με τις ελληνικές ε, αρχές έτσι ώστε να οδηγηθούμε σύντομα σε ένα αναθεωρημένο και επικαιροποιημένο σχέδιο αντιμετώπισης ετών hot spot. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Διευθυντής Επιχειρήσεων τη Frontex, Κλάου Ρόσλερ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο έργο της Frontex. Υποστηρίζει απόλυτα η Frontex την προσέγγιση με hotspots ως ε, αναπόσπαστο τμήμα των ε, δράσεών μας. Αυτή τη στιγμή 114 ε, αξιωματούχοι δρούν στη Λέσβο πάνω από 40 στοιχείο, 32 στη Σάμο, 44 στη Λέρο και στο Αγαθονήσι και 33 στην Κό. Είναι αναγκαίο λοιπόν να κάνει κανείς λόγο όχι μόνο για τους ρόλους αλλά και για τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και τα θέματα ασφάλειας που αντιμετωπίζουμε όταν συνεπικουρούμε την διαδικασία υποδοχής μεταναστών από πλευρά των ελληνικών αρχών ως Frontex το περιορισμένο δυναμικό στέγασης και υποδοχής μεταναστών. Οι περιορισμένες δυνατότητες καταγραφής ε, αυτοί είναι οι παράγοντες που αποτελούν προκλήσεις ε, και πρέπει συστηματικά να μπορέσουμε να προβούμε στην καταχώρηση, καταγραφή ως τμήμα της υποδοχής και διαχείρισης ε, των ροών μεταναστών στη χώρα. Υπάρχει ανάγκη μια στρατηγική αντιμετώπισης κρίσεων να λειτουργήσει με πλήρη στοχοθέτηση την κατάσταση όσον αφορά τους μετανάστες. Υπάρχει έλλειψη δυναμικού και πόρων για την ε, επαρκή υποδοχή των μεταναστών. Επίσης ε, κενά που υπάρχουν όσον αφορά το δυναμικό, ανθρώπινο δυναμικό από πλευράς ε, των ελληνικών αστυνομικών αρχών θέματα ασφάλειας ε, όσον αφορά την εθνικότητα ή ε, την, ε, τις εναλλασσόμενες, την εναλλασσόμενη υπηκότητα ατόμων που προέρχονται από το Αφγανιστάν, τη Συρία, το Ιράν. Υπάρχουν εδώ θέματα ασφάλειας με την έλλειψη, απουσία ταξιδιωτικών εγγράφων. Δεν υπάρχει ένα πλαίσιο ασφάλειας και μπορούν πολύ εύκολα να χακευθούν, να υπάρχει πλαστογράφηση των ταξιδιωτικών εγγράφων. Υπάρχει και το θέμα της σταδιακής ε, ενίσχυσης ε, της κοινή ε, δράσης Ποσειδών, Ποσάιντων. Ωστόσο όλα αυτά θα εξαρτώνται από, αυστηρά από το δυναμικό υποδοχής της χώρας υποδοχής για τα θέματα καταγραφής, καταχώρησης, δημιουργίας μητρών, φωτογράφησης, δακτυλοσκόπησης Υπάρχει λοιπόν το πρότυπο αυτό από πλευράς Frontex που θα επεκταθεί στην Ελλάδα όχι μόνο στη Λέσβο αλλά και στα άλλα τέσσερα νησιά που προαναφέραμε και είμαστε έτοιμοι να, συνδράμουμε ε, αυτή την ε, περιφερειακή μονάδα European Task Force στον Πειραιά από κοινού με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για το Άσυλο καθώς επίσης και την EU lisa και την Ευρωπόλ. Σε αυτή τη φάση αναλύει τα αιτήματα για την γοργή άμεση δράση και αντίδραση από πλευρά της Frontex ε, με στοιχεία τα οποία έχουν κατατεθεί, έχουν υποβληθεί από πλευρά πλευράς των ελληνικών αρχών και στις ελληνικές αρχές ε, και που θα μπορέσουν να αναλυθούν για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και πριν ε, ε ολοκληρώσουμε ε, θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον εκπρόσωπο της IRC που έχει αρκετό κόσμο στην Ελλάδα. Ράνη παρακαλώ δώσε μας την άποψή σου. Ευχαριστώ πολύ. Λέγομαι Ελένη Φόργερ και είμαι ε, υπεύθυνη της χώρας, ε, υπεύθυνη χώρας για τα προγράμματα ε, στην Ελλάδα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί μας δώσατε την ευκαιρία σήμερα να δώσουμε την άποψή μας σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα. Ε, δημιουργηθήκαμε πριν από πάρα πολλά χρόνια και τώρα δουλεύουμε με 40 ε, ε, χώρες και έχουμε συμμετάσχει στην αντιμετώπιση μερικών από τις περισσότερες ανθρωπιστικές κρίσεις. Είμαστε ε, η μοναδική μη κυβερνητική οργάνωση η οποία ε, ασχολείται με κάθε είδους ε, κρίσης. Τον Ιούνιο ξεκινήσαμε την ανταπόκρισή μας στη Λέσβο και δεν φύγαμε ποτέ από το νησί έκτοτε έχουμε ε, περισσότερους από 100 ε, ε, επαγγελματίες που δουλεύουν εξ ονόματος της IRC και όσον αφορά την πρόσβαση σε πόσιμο νερό αλλά και όσον αφορά την μετακίνηση και τις μετατοπίες μετακινήσεις και μεταφορές. αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληρώσει πάνω από 2.000 ευρώ ο καθένας σε διακινητές έτσι ώστε να περάσουν σε αυτά τα νησιά στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για πρόσφυγες που προσπαθούν να ξεφύγουν από πολέμους στη Συρία ή αλλού και από επισφαλείς καταστάσεις. Περισσότεροι από τους μισούς μπορεί και να έχουν πεθάνει στη διάρκεια του ταξιδιού. Από τον Αύγουστο ε, μέχρι τον Σεπτέμβριο, εκεί που η Ανθή μας έδειξε ε, που <coughs> φτάσανε, πεθάνουν οι περισσότεροι ε, είναι άντρες, γυναίκες και παιδιά που φτάνουν εκεί και περπατούν ε, πάνω από 70 χιλιόμετρα μέσα από δύσβατες περιοχές και επικίνδυνους ε, δρόμους. Εμείς παρέχουμε νερό, και προσπαθούμε να παράσχουμε και ιατρική βοήθεια γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα, ζουν, στη, κοιμούνται στις άκρες του δρόμου ε, και ε, ακόμα και αν μπορέσουν να βρουν κάπου να κοιμηθούν ε, πίνουν από δημόσιες βρύσες, δεν έχουν δυνατότητα για υγιεινή κτλ. Είναι η χειρότερη κατάσταση που έχουμε βρει ήδη τον Αύγουστο, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, ακόμα και τον Νοέμβριο οι αφήξεις παραμένουν υψηλές οι διαδικασίες πρώτης ε, υποδοχής στην ε, Μόρια ε, είναι ελλειπή σε γενικές γραμμές και επίσης η διαδικασία ταυτοποίησης αλλάζει από καιρούς καιρών και προκαλούνται εντάσεις και επικίνδυνες τριβές. Ε, αυτό έχει σαν ε, αποτέλεσμα να περιμένουν οι άνθρωποι αυτοί μέχρι να πάρουν τα διοικητικά τους έγγραφα αρκετό καιρό ε, και σε πολύ κακές συνθήκες. Ε, τους τελευταίους πέντε μήνες ε, έχουμε διαπιστώσει συχνές τριβές και εντάσεις ανάμεσα στους, στις ομάδες των προσφύγων. Λίγο έχει φτιάξει η κατάσταση από όταν ξεκίνησε η λειτουργία του hot spot στην Λέσβο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να οι, οι, άνθρωποι αυτοί, οι πρόσφυγες αυτοί να μπορέσουν με αξιοπρέπεια να προχωρήσουν το δρόμο τους και την πορεία τους προς τα εκεί που έχουν επιλέξει να πάνε. Αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι υπήρχε διαφορά ανάμεσα στην πραγματικότητα που αντιμετωπίζαμε εμείς επιτόπου και τις αποφάσεις που ελαμβάνονται σε υψηλότερο ε, επίπεδο. Ο φόβος μας ε, είναι ότι ε, η διαδικασία ταυτοποίησης θα εξακολουθήσει να είναι η πιο σημαντική διαδικασία ε, και όχι η ανταπόκριση στις βασικές ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Δεύτερον, υπήρξε ελλειπής πληροφόρηση όσον αφορά την εισαγωγή του hot spot. Στη Λέσβο ήταν δύσκολο να ε, εγκατασταθεί η διαδικασία και να στηριχτεί ο κόσμος. Οι διαβουλεύσεις με τους με τις ε, ε, οργανώσεις οι οποίες δρούν επί στο μέλλον θα μπορούσε ε, να διευκολύνει την κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, το, τα τελευταία χρόνια είχαμε περίπου 66.000 ε, ανθρώπους να φεύγουν από την Ελλάδα ενώ έχει αυξηθεί υπερβολικά ο αριθμός ε, το τελευταίο καιρό. Ε, γίνεται υπερβολική επικέντρωση στα ε, hot spots αλλά υπάρχουν και τις υπηρεσίες που παρέχονται αλλά υπάρχουν πάρα πολλές χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι επιλέξιμοι για αυτές τις υπηρεσίες και για αυτήν την αντιμετώπιση. Στην Λέσβο ήταν σαφές αυτό από την αρχή και δημιούργησε μεγάλες εντάσεις. Ωστόσο, ε, με την δημιουργία επιπλέον ε, hot spot φοβούμε ότι το μάθημα και η διδασκαλία της Λέσβου ε, δεν έχει γίνει γνωστή στους υπουργούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Θα πρέπει να μας πει η Επιτροπή τι έχει κάνει έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά και σε, σε όλα τα υπόλοιπα hot spots τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίστηκαν στη Λέσβο. Τι μπορεί να γίνει έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι η Τουρκία μπορεί πραγματικά να βοηθήσει και θα λειτουργήσει σωστά σε αυτή τη την διαδικασία. Ε, θα ήθελα να ασχοληθείτε με τα ερωτήματα αυτά. Και βεβαίως ε, είμαι στη διάθεσή σας ε, για οποιασδήποτε ερωτήσεις θα μπορούσατε ενδεχομένως να υποβάλετε. υποβάλλετε. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Και εσείς υποβάλλατε ερωτήματα και επομένως θα πρέπει η Κομισιόν να απαντήσει για να δούμε ακριβώς πώς θα προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας ε, γιατί οι ομιλητές δεν ξεπέρασαν το χρόνο ομιλίας τους και επομένως θα δώσω το χρόνο τώρα ε, στους, στη δυνατότητα τώρα στους βουλευτές να ρωτήσουν ή να θέσουν τις παρατηρήσεις τους. Η κυρία Χολμάγερ, παρακαλώ από το ΕΛΚ. Δύο λεπτά κυρία Χολμάγερ και οι αγαπητοί συνάδελφοι. Κανείς δεν ξεπεράσει τα δύο λεπτά. Άμεσα προς τις ερωτήσεις να περάσω. Πρώτη ερώτηση προς την Frontex και την EASO, ιδιαίτερα όσον αφορά την ελληνική πλευρά, πόσα άτομα θα χρειαζόντουσαν ώστε να μπορέσει να ελεγχθεί η κατάσταση όχι μόνο όσον αφορά την καταγραφή και καταχώρηση αλλά και υπό το πρίσμα ότι χρειάζονται και τροφή την σύντηση που πρέπει να διασφαλιστεί για αυτά τα άτομα και πράγμα το οποίο δεν μπορεί μόνο από την ευρωπαϊκή πλευρά να καλυφθεί αλλά και υπάρχουν υποχρεώσεις και του κράτους μέλους. Πώς βλέπετε τη δυνατότητα της Ελλάδας σε σχέση με τα στελέχη που χρειάζονται ώστε στις νήσους αυτές να διασφαλιστούν οι αναγκαίες συνθήκες διαβίωσης. Επίσης κατά πόσον ΜΚΟ, μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, που πολύ δύσκολες ε, συνθήκες αντιμετωπίζουν, ποιες προσδοκίε θα είχατε όσον αφορά την Ελλάδα για την υποστήριξη και συνδρομή των ΜΚΟ ε, εμείς στην Γερμανία έχουμε καλά, καλή πείρα με τη συνεργασία με ΜΚΟ γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να είχαμε αντιμετωπίσει τα προβλήματα των μεταναστών. Αναφέρατε ότι οι δακρυγόνα και τα λοιπά είχαν χρησιμοποιηθεί και στις εκπομπές των τηλεοπτικών δικτύων τα είχαμε δει αυτά. Κατά πόσον λοιπόν υπάρχουν επαρκή, υπάρχει επαρκή στελέχωση τι μπορεί να γίνει ώστε να καταρτιστεί και να επιμορφωθεί το προσωπικό, ώστε οι ομάδες ατόμων να μπορούν να διαχωρίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχουν τέτοιες εντάσεις ε, ή και οι εντάσεις ε, να μην δημιουργούνται λόγω εθνοτικής, ε, εθνοτικών αιτίων ή εθνικών αιτίων. Υπήρχε και συνοστισμός μεγάλος των ατόμων αυτών που ήταν ολέθριος και τα άτομα αυτά δεν άντεχαν πλέον και επιπλέον όσον αφορά την Frontex. Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε εμείς, υπάρχει πάρα πολύ ε, α, άτακτος ρυθμός μεταφοράς ε, των μεταναστών από τα νησιά κατά πόσον θα χρειαζόντουσαν ε, από πλευράς λιμενικού ή ακτοφυλακής ε, η αναγκαία, προς, η αναγκαία στελέχωση ώστε να πάψει να υπάρχει αυτό το λαθρεμπόριο και να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να προστατεύουν. προστατεύουν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Στη συνέχεια εσείς έχετε τον λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Μια εκ παρατήρηση θα ήθελα να κάνω. Ελπίζω ότι όλοι γνωρίζουν πλέον ότι εμείς όλοι ως Ευρωπαϊκό Θεσμικό Όργανο, ως Ευρωβουλή, αλλά και όλα τα κράτη-μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με μεγάλη καθυστέρηση αντιδράσαμε. Τώρα οι προκλήσεις είναι τεράστιες και δεν έχει ιδιαίτερο λόγο εδώ να κατηγορεί ο ένας τον άλλον πλέον, αλλά θα πρέπει από κοινού εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης όλοι να κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε τα πράγματα με βάση αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Συμφωνούμε επ' αυτού. Για τα επειδή παράλληλα με τα ανθρωπιστικά θέματα υπάρχουν διαφορετικές διάφορες φήμες που κυκλοφορούν. Κάποιες ερωτήσεις θέλω να θέσω. Είναι διαμφισβήτητο ότι η καταγραφή όλων των μεταναστών πρέπει να επιτευχθεί και εδώ χρειάζονται βελτιώσεις. Δεύτερο ερώτημα, δεύτερο ζήτημα που πρέπει να αποσαφινιστεί κάθε άτομο, κάθε πρόσφυγας ε, που ε, φτάνει, που ε, γίνεται δεκτός πρέπει να υπόκειται σε μια τέτοια διαδικασία. Όποιος δεν έχει όμως δικαίωμα να τύχει χορήγησης ασύλου πρέπει να επιστρέφει, να ε, μπορεί να επιστρέφει στη χώρα από την οποία προήλθε. Υπάρχουν όμως εδώ και θέματα ατόμων που ε, είναι πρόσφυγες ε, λόγω πολεμικών σειράξεων στις χώρες τους. Δεν είναι εύκολο αυτό να αποσαφινιστεί. Είναι αυτονόητο ότι όλοι οι πρόσφυγες λόγω πολεμικών σειράξεων έχουν δικαίωμα να εγκατασταθούν στις χώρες υποδοχής και δεν μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες από τις οποίες προήλθαν Τέλος, τέλος, ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα αποφασίζει, ποιος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να τύχει ασύλου και να αναγνωριστεί ως ε, ε, δικαιούχος ασύλου. Η Frontex, Ευρωπόλη, η ΕΑΣΟ θα συμμετέχουν στις δράσεις των ελληνικών αρχών και με ποιο τρόπο θα γίνεται αυτό. Τρίτη ερώτηση. Γίνεται πολλή λόγος και πρέπει να ολοκληρώσω τώρα με την παρέμβασή μου ότι πρέπει να διασφαλίζεται η καταγραφή όλων αυτών των ατόμων. Τι θα συμβαίνει όμως όταν όλοι αυτοί οι πρόσφυγες θα καταγράφονται στην Ελλάδα, κανένας δεν θα μπορεί παράτυπα ή παράνομα να μεταβεί αλλού και πώς όλα αυτά θα μπορούν να λειτουργήσουν σε σχέση με την ευρωπαϊκή μετεγκατάσταση το πρόγραμμα μεταγκατάσταση. Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει και το θέμα της έκφρασης τη Ευρωπαϊκή αλληλεγγύης απέναντί τη Και τελευταίο σημείο, ποιος είναι εκείνο ο οποίο είναι αρμόδιος για την καταγραφή των διαφορετικών ηλικιών των προσφύγων. Αν είναι κάποιοι κάτω από 16 ή πάνω από 16 ή 20 ετών. Και ποιο είναι εκείνο ο οποίο θα αποφασίζει σε σχέση με την Frontex ποιοι θα επιστρέφουν στη τις χώρες τους ε, και με βάση ποιες διαδικασίες για τη λήψη απόφασης. Σας ευχαριστώ. Εσείς από τους συντηρητικούς και μετα... μεταρρυθμιστές παρακαλώ. Thank you, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τις παρουσιάσεις για την Ελλάδα και επίσης έλαβα και πολλές πληροφορίες και από άλλους. Ε, τα hot spot φαίνεται πως λειτουργούν ε, σωστά διότι όλοι πρέπει να καταγραφούν. Και φαίνεται πως οι περισσότεροι καταγράφονται στα hot spot αυτά. Και αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, διότι το σκεπτικό πίσω από όλο αυτό ήταν ακριβώς ε, αυτό. Ταυτόχρονα, αν κατάλαβα καλά, το σκεπτικό των ε, hot spot ε, δεν οδηγεί ε, σε ένα λειτουργικό αποτέλεσμα, διότι εάν οι πληροφορίες μου είναι σωστές, μέσα σε 24 ώρες μετά την καταγραφή φεύγουν από το νησί. Αυτή λοιπόν η διαλογή σε πρώτο στάδιο δεν λειτουργεί. Εάν δηλαδή είσαι ελεύθερος να φύγεις το καταγραφείς, δεν έχει αποτέλεσμα. Θα μπορούσατε λοιπόν να μου εξηγήσετε πώς γίνεται αυτή η διαδικασία καταγραφής, εάν ελέγχεται, εάν προέρχονται όντως από τη χώρα που λένε πώς προέρχονται, εάν είναι από τη Συρία ή το Ιράκ. Εντάξει, αυτές οι χώρες εμαστίζονται από πολέμους, όμως όταν υπάρχει κάποιος με πλαστό διαβατήριο, πώς μπορείτε να το ελέγξετε αυτό σωστά διότι αν κατάλαβα καλά δεν είναι μια ε, πραγματική διαλογή, είναι μια καταγραφή σε χαρτί και μετά ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να φύγει. Δεν Καταλαβαίνω λοιπόν το πώς αυτό ακολουθεί το σκεπτικό του hot spot. Η ε, Αντζέλικα Μίλνερ για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες στο πάνελ, όλους τους εμπειρογνώμονες, διότι παρήχατε μία πάρα πολύ ε, σημαντική ε, βοήθεια στο να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Ε, μπορούμε να παρακολουθήσουμε όλη την ε, συζήτηση. Τις τελευταίες ημέρες η Ελλάδα μάλιστα δέχτηκε ε, την απειλή του να φύγει, να εκδιωχθεί από τον χώρο του Σέγγεν και συμφωνώ με την κυρία Ζίπελ η οποία είπε ότι είναι γενικά ευθύνη όλων μας το τι συμβαίνει στα εξωτερικά σύνορα. Τα εξωτερικά σύνορα λοιπόν διαχειρίζονται είτε ε, ανεπαρκώς είτε ε, λάθος. Αυτό ε, βέβαια δεν είναι φταίξιμο της Ελλάδας μόνο και η Τουρκία είναι ένα προβληματικό σημείο. Χρειάζεται λοιπόν να βρούμε μία κοινή λύση. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Στην έκθεση βλέπω την ισχύουσα κατάσταση ε, για τις 11 Οκτωβρίου και μόνο το 3% του εξοπλισμού που ζητήθηκε ε, εγκρίθηκε για την Ελλάδα. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω ε, τι γίνεται τώρα, ποιο είναι το ποσοστό του εξοπλισμού που λείπει, τι εξοπλισμός υπάρχει. Δεύτερη ερώτηση σχετικά με την κατάσταση αυτών των 30 ανθρώπων που είναι πραγματικά ένας πάρα πολύ μικρός αριθμός. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε ποια είναι τα μέτρα τα οποία οραματίζεστε εσείς σχετικά με το πώς θα γίνει ε, με επιτυχία αυτή η μετακατάσταση των ε, ανθρώπων. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Έρνστ για την ΕΓΚΟΕ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, ότι υπάρχει μια κατάσταση ε, που έχει πάρα πολλά προβλήματα με την διαδικασία ασύλου και τώρα προσπαθούμε ε, με κάθε τρόπο να ε, βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω τρεις ερωτήσεις. Καταρχάς, τα οικονομικά. Ε, γνωρίζουμε ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό η Ελλάδα δεν έλαβε ευρωπαϊκή οικονομική βοήθεια, ιδιαίτερα στον τομέα της μετανάστευσης. Όμως ακούσαμε ότι και η αρμοστία του ΟΗΕ έχει εκφράσει τις καταγγελίες της ότι υπάρχουν μεγάλα κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν καταβάλει επαρκής, ε, επαρκή οικονομική βοήθεια για τη δημιουργία αυτών των hotspot. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε πώς ε, συνεχίζεται η κατάσταση, πώς θα συνεχίσουμε. Έπειτα, ε, Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση για τις μη κυβερνητικέ οργανώσει και του χωρίς χωρί σύνολο θα την αργότερα. Δεύτερον, όταν λείπει η υπηκότητα κάποιου ανθρώπου, πολλέ μη κυβερνητικέ οργανώσεις μας έχουν πει ότι ε, υπάρχει συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο ότι είναι παράνομη η διαδικασία και ότι παραβιάζει την σύμβαση για τους πρόσφυγες. Τι συμβαίνει με τους ανθρώπους που πρέπει να ε, επιστραφούν. Μένουν πρώτων πυλών, τους ε, αφήνουν κάπου και δεν, ενδιαφέρει, δεν τους ενδιαφέρει τι γίνεται στη συνέχεια, τι γίνεται μετά την καταγραφή όταν διαπιστωθεί πως η υπηκότητα κάποιου δεν είναι ε, η επιθυμητή, ας πούμε, εντός εισαγωγικών. Και μετά, σχετικά με τον αριθμό των ε, ανθρώπων που μου μετακαταστάθηκαν, συγχαρητήρια. Και το λέω αυτό ηρωνικά φυσικά. Έπειτα, ποια είναι η άποψή σα για το σύστημα του Δουβλίνου. Χρειάζεται αλλαγή, χρειάζεται βελτίωση, κατάργηση, τι. Μπορούμε να διατηρήσουμε το σύστημα αυτό έτσι όπως ε, έχει. Ε, κάποιος από εσάς αναφέρθηκε σε αυτό και θα ήθελα να μάθω περισσότερε λεπτομέρειε για το πώς φαντάζεστε την εξέλιξή του. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει να μιλήσει εξ ονόματος των Πρασίνων, ε, γιατί η κυρία Σκάκελα δεν είναι εδώ. Αν όχι, Τότε να περάσουμε ε, στην Λάουρα Φεράρα, FTD. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα κάποιες αποσαφηνήσεις ε, όσον αφορά τις διαδικασίες ταυτοποίησης. Θα ήθελα να καταλάβω ποιες είναι οι δυσκολίες που ε, συγκεκριμένα αντιμετωπίζονται στις διαδικασίες ταυτοποίησης και επίσης ποιοι ε, ε, είναι, ε, οι πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι καταφέρνουν να διασχίσουν την Ελλάδα χωρίς να έχουν ταυτοποιηθεί και να φύγουν. όσον αφορά τώρα τους επαναπατρισμούς, ε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τύχουν της διεθνούς προστασίας τι γίνεται με αυτούς. Ε, δηλαδή υπάρχει δυνατότητα αυτά τα hot spots ε, τελικά να καταλήξουν κέντρα κράτησης ή υπάρχουν διαδικασίες ε, διαφορετικές. Επίσης, σε σχέση με πριν, ε, πώς έχει βελτιωθεί η κατάσταση σε σχέση με τα hot spots, δηλαδή ε, η ταχύτητα είναι μεγαλύτερη, ε, έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό ταυτοποίησης, γιατί όσον αφορά την ε, επανεισδοχή τα, οι αριθμοί είναι πάρα πολύ μικροί και επομένως καταλαβαίνουμε ότι σε αυτό το σημείο δεν έχουμε ε, κάποια βελτίωση ε, γιατί ξέρετε μας αναφέρουν τα hot spots σαν να είναι πανάκια ε, στην ε, μεταναστευτική αυτή κρίση. Επομένως θα ήθελα να ξέρω με συγκεκριμένο τρόπο πώς έχει αλλάξει η κατάσταση λόγω των hot spots και τι είδους βελτίωση έχουν επιφέρει. Ευχαριστώ. Ρομπέρτο Ματσόλα. Ρομπέρτα Ματσόλα. Θα είμαι σύντομη. Δυστυχώς ε, δεν θα είμαι εδώ για να ακούσω τις απαντήσεις σας, ε, γιατί πρέπει να είμαι σε μια άλλη επιτροπή, αλλά εν πάση περιπτώσει θα θέσω τα ερωτήματα. Ευχαριστούμε την ΕΑΣΟ ε, που ήρθε και επικαιροποίησε λίγο τη θέση της απέναντι στην δικιά μας κοινοβουλευτική επιτροπή. Κύριε Σκέμπρη, είπατε ότι ο αριθμός των των εμπειρογνωμόνων ε, ε, δεν σας, ικανοποιεί. Τι κάνει ακριβώς η ΕΑΣΟ, ε, τα, τα αιτήματά της τελικά τα απαντούν ας πούμε τα κράτη-μέλη με τις κινήσεις που κάνουν ή πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Και όταν αναφέρομαι σε κράτη-μέλη, αναφέρομαι σε όλα τα κράτη, όχι μόνο αυτά που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Επίσης, ποια είναι τα λεπτά σημεία ε, της ε, relocation. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το συζητάμε, το ξανασυζητάμε και βεβαίως... Ε, οποιαδήποτε επικαιροποιημένη πρόταση ή πληροφορία έχετε είναι σημαντική. Επίσης, ε, Frontex, ε, μιλάμε για την, Ιταλία, για την Ελλάδα τώρα, θα μιλήσουμε για την Ελλάδα, συγγνώμη, για την Ελλάδα τώρα, θα μιλήσουμε και για την Ιταλία μετά. αλλά ε, για την ώρα μόνο θα έχουμε τις δύο αυτές χώρες. Προφανώς θα πάει και αλλού η Frontex. Ε, σημείο εισόδου, μεταξύ του σημείου εισόδου και του σημείου εξόδου ε, των ανθρώπων αυτών, τι γίνεται, ποια είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα σημεία εξόδου, δηλαδή εκεί που φεύγουν. Όσον αφορά τώρα τα ψεύτικα διαβατήρια, τα πλαστά διαβατήρια, στα εξωτερικά σύνορα Σέγγεν ε, γίνεται κάποια έρευνα σχετικά με τα διαβατήρια. Ε, δεν θα πρέπει να συνεχίσουν οι έλεγχοι και εσωτερικά. Ε, γιατί θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι τα αριθμητικά στοιχεία τα οποία έχετε. Και αυτή είναι και ερώτηση προς την εκπρόσωπο της ελληνικής πολιτείας. Πόσα είναι αυτά τα διαβατήρια τα οποία έχετε βρει πλαστά στα σημεία εισόδου. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά πρέπει να πω ότι έφρυξα. Στη χώρα μου επί μήνες έλεγαν οι άνθρωποι γιατί δεν έρχονται οι πρόσφυγες, όλα είναι έτοιμα για αυτούς. Και η μεθοριακή υπηρεσία έλεγαν όχι, να μην έρθουν στην Πορτογαλία. Ο νέος Υπουργός ε, Εσωτερικών είπε, διόρθωσε, όχι επειδή ήταν βραδία διαδικασία όπως σε χώρες ε, στην Ιταλία και την Ελλάδα για τα hot spots ε, και πρέπει να γίνει κάποια δουλειά πιο πριν. Είναι όμως φρικτή αυτή η κατάσταση. Ποιος είναι ο υπεύθυνο. Γιατί σε σχέση με μια έκδηλη κρίση στην ΚΟ η πρωτοβουλία 70 μελών ευρωβουλευτών που έστειλαν μια επιστολή γιατί δεν ζήτησε τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας να λειτουργήσει άμεσα στην ΚΟ οι ελληνικές αρχές Έφρυξα με την απάντηση που ε, έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτό λέει είναι κάτι το οποίο μπορεί να απαντήσει ως ερώτημα μόνο η ελληνική κυβέρνηση. Και πραγματικά τι γίνεται εδώ. Έξι μήνες αργότερα τι έχει γίνει. Γιατί πήρε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ενώ ήταν πραγματικά κατεπίγουσα η κατάσταση. Κάτι δεν λειτουργήσε καλά και δεν λειτουργεί καλά. Ντρέπομαι. Έσχος είναι αυτό. Ως Ευρωπαία πρέπει να πω ότι ντρέπομαι για αυτή την κατάσταση δυστυχώς. Και έχω και κάποιες ερωτήσεις πράγματι εδώ και θα ήθελα να τις θέσω πραγματικά. Εσείς κύριε αναφέρατε και είπατε ότι δεν υπάρχουν αρκετές επιστροφές. Ποιοι επιστρέφουν και ποιος αποφασίζει για αυτές τις επιστροφές. Ο στόχος είναι αφεαυτού στόχος η επιστροφή, η, ε, η επανεισδοχή, η επιστροφή αυτών των ατόμων. Και ποιος αποφασίζει, τι γίνεται. Και προς την Ελληνίδα εκπρόσωπο να σας ρωτήσω, τι πιστεύετε ότι είναι το πρόβλημα όπως ανέφερε η συνάδελφος ότι δεν υπάρχει η συνδρομή, χρήματα η συνδρομή, γιατί πήρε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα η ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει να λειτουργήσει ο μηχανισμός ε, ε, πολιτικής προστασίας και η ερώτησή μου προς εμάς επίσης και σας ευχαριστώ για το υπενθυμίσατε αυτό ότι η Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης αναφερόταν αρχικά σε πρόσφυγες από την Ευρώπη που έπρεπε να διασωθούν και το ξεχνάμε αυτό. Μια και τόσες πολλές γυναίκες και παιδιά ιδιαίτερα μη συνοδευόμενα παιδιά ανήλικοι συμμετέχουν πρέπει να εξεταστεί η κατάστασή τους ξεχωριστά. Εσείς θα προσέθετε ώστε να παρουσιαστεί αυτή η πτυχή και να επαναληθεί. Ευχαριστώ. Εσύ Ζεράρ, παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ζερά, Ντεπρέ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, μου, λίγο αφηρημένος. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές γιατί μας έδωσαν σημαντικές πληροφορίες. Έχω μερικές ερωτήσεις όμως. διάβασα σε κάποιες εφημερίδες που έλεγαν ότι ορισμένοι πρόσφυγες προσπαθούσαν να μην ταυτοποιηθούν. Αληθεύει? Ε, άκουσα ότι υπήρχε συνοστισμός ε, και σύγχυση. Ε, ε, υπάρχουν λοιπόν όντως ε, άνθρωποι οι οποίοι δεν ταυτοποιούνται. Επίσης ακούσαμε για τη Λέσβο. Εκεί που δεν υπάρχουν οργανωμένα hot spots, τι γίνεται, έχετε πληροφορίες. Εδώ εκπροσωπούνται επίσης διάφοροι οργανώσεις, φορείς κτλ. Αλλά ποιος κάνει τι. Ποιος κάνει τι, με ποιο τρόπο οργανώνεται πραγματικά ε, η συνεργασία με τις ελληνικές αρχές και μετά με τις ιταλικές. Μια ερώτηση η οποία αφορά περίπου τα hot spots κυρίως αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να μπουν και θέλουν να ταυτοποιηθούν, να καταχωριστούν. Έχετε μία ιδέα ποιο είναι το ποσοστό των πραγματικών προσφύγων ε, οι οποίοι ε, είναι πιθανό να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες ε, σε αντιπαράθεση με τους οικονομικούς μετανάστες. Τους ξεχωρίζετε, εάν τους ξεχωρίζετε τους βάζετε κάπου αλλού, τους αφήνετε να φύγουν, τι συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν κατάλαβα πολύ καλά τι γίνεται σε καμία από τις παρεμβάσεις που άκουσα. Και μία τελευταία ερώτηση μεταξύ των προσφύγων. Έχετε μια ιδέα ποιο είναι το ποσοστό αυτών που εμπίπτουν στην κατηγορία του 77% δηλαδή, ε, έτσι τους λέω εγώ, ε, αυτοί δηλαδή που αυτόματα θα τους αναγνωριστεί το δικαίωμα το, του, του καθεστώτος του προσφύγου και θα μπουν επομένως στο σύστημα κατανομής. Και τι γίνεται με αυτού του ανθρώπου που εμπίπτουν δηλαδή στο 77% ε, την χάνουν μια ειδική μεταχείρισης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, έχουμε ακόμα τρεις ομιλητές. Τρεις ομιλητές και δεν έχει ζητήσει κάποιο... Α, και εσύ. Ωραία, ναι, ναι, ήσουν στον κατάλογο τρεις ε, δεν έχουν ζητήσει άλλη το λόγο και επομένως ε, θα ε, κλείσει ο κατάλογος. Η κυρία Βερζιά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να υποβάλω κάποια ερωτήματα σε όλους σας ε, για την ανάλυση ε, των ε, ροών προς την Ελλάδα και από την Ελλάδα, προς την Ελλάδα μάλλον, γιατί θα έπρεπε να καταλάβουμε για ποιο λόγο η Ελλάδα βρέθηκε να υποδέχεται τόσους πρόσφυγες. Συμφωνώ με αυτά που ακούστηκαν για την Τουρκία, γιατί και σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες που μαθαίνουμε φαίνεται ότι περιέργως, περιέργως ε, είναι όλο και λιγότεροι οι Σύροι οι οποίοι φτάνουν και βεβαίως εγώ δεν θέλω καθόλου να αμφισβητήσω τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία, αλλά θα ήθελα να μου πείτε τι διαπιστώνετε εσείς. Επίσης λέτε ότι έχετε δυσκολία με τον έλεγχο των διαβατηρίων. Όταν υπάρχουν προβλήματα λοιπόν με τα διαβατήρια, τι γίνεται με τους ανθρώπους που έχουν αυτά τα προβληματικά διαβατήρια. Επίση, θα συμφωνήσω με τον κύριο Ντεπρέ, ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό ε, κάποια στιγμή μπορεί να λειτουργήσει, ακόμα δεν λειτουργεί, αλλά εν πάση περιπτώσει αφορά τους 75-77% αυτοί δηλαδή οι οποίοι θα μπουν σε αυτό το σύστημα. Για τους ε, υπόλοιπους, ε, τι γίνεται, υπάρχουν ε, στους υπόλοιπους άνθρωποι που μπορούν να ζητήσουν άσυλο και Πώς ξεχωρίζετε λοιπόν αυτούς τους καλούς πρόσφυγες που θα μπουν στο σύστημα κατανομής και τους άλλους ε, κακούς πρόσφυγες. Ε, γιατί να μην λησμονούμε ότι όλα τα ευρωπαϊκά, όλες οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχουν προσυπογράψει τη συνθήκη της Γενέβης. Επίσης, τι γίνεται με την πολιτική επαναπατρισμού και εγώ θα ήθελα συγκεκριμένες πληροφορίες γι' αυτό πόσα είναι τα άτομα που αυτή η πολιτική αφορά, πόσοι είναι αυτοί που είναι στην Ελλάδα τώρα και πρόκειται να φύγουν, πόσους έχει διώξει. Επίσης, τι γίνεται με τη δράση της Frontex στα σύνορα της Φύρομ. Γιατί ε, μιλήσατε για τα νησιά, αλλά εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε και για την άλλη πλευρά. Ε, τι γίνεται στα χερσαία σύνορα. Ε, γιατί ε, ε, φαίνεται ότι έχουμε εκεί διπλές, τριπλές καταχωρήσεις, οι πληθυσμοί δεν αντέχουν πλέον. Τι γίνεται εκεί. Ο κύριος Κρυκόπ, παρακαλώ τώρα. Και να γνωρίζετε. Εσείς κύριε Κύρκο, έχετε τον λόγο. Θα μιλήσω ελληνικά, Πρόεδρε. Τον υπεύθυνο της Κομισιόν, αν και η ενημέρωση ήταν παντελώς ασαφής. Υποτίθεται πω τέλο Οκτωβρίου θα ήταν έτοιμα τουλάχιστον ένα ή θα ήταν έτοιμα τα hot spots όπω μα είχαν πει. Σήμερα ενημερωθήκαμε πω θα υλοποιηθούν τα hot spots και το hot spot τη Αθήνα που θα είναι και το μεγαλύτερο δεν είπαμε τίποτα, δεν έχει καν γίνει οριοθέτηση. Θα γίνουν θέσει φιλοξενία, κάτι αναφέρθηκε ο ΙΕ, θα, είμαστε σε ένα μέλλον. Θα εγκατασταθεί η Frontex σε κάποια σημεία. Βλέπουμε δηλαδή πω βρισκόμαστε σε ένα πολύ μεγάλο θα. Εδώ και μήνε ε, σα ενημερώναμε πω θα έρθει αυτή η στιγμή, πω δεν προχωράνε τα πράγματα, Πώ έχουν φρακάρει τα πάντα. Τι μάθημα πήρατε από την ενημέρωση που μα κάνετε εδώ και δύο μήνε και 45 μέρε και ένα μήνα και 15 μέρε κάθε φορά σα λέγαμε δεν προχωράει και κάθε φορά μα λέγατε θα. Έχετε πάρει ένα μήνυμα που θα να κάνουμε να ελπίζουμε λίγο. Και το δεύτερο, 5.000 τη μέρα φτάναν στη Μυτιλίνη, φτάναν στη Λέσβο. 150 έχουν μεταφερθεί με το relocation. Πού πάνε οι άλλοι η, ανάπτυξη της Frontex στα σύνορα με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας δείχνει ότι πολλοί φτάνουν εκεί χωρίς καν να έχουν ελεγχθεί. Δεν είναι λογικό πως αν οι πρόσφυγες απλώς παίρνουν το δρόμο του Δυτικών Βαλκανίων, πολύ σύντομα θα κλείσουν τα σύνορα της Ευρώπης. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε κάποιον έλεγχο σε αυτά. Ελέγχονται άνθρωποι και μετά εξαφανίζονται πάλι, όπως γινόταν και το καλοκαίρι. Για την κυρία Καραγγελή, θέλω να επιβεβαιώσω και εγώ και για τη δική της την προσφορά και για την προσφορά όλων των ανθρώπων που είναι στο πεδίο. Πραγματικά δουλεύουν με εκπληκτική αυτοθυσία. Όμω, όπω θυμάται και ο πρόεδρο Μωράε, από τον Ιούνιο προσπαθούσαμε να δούμε αυτόν τον καταραμένο μηχανισμό πολιτική προστασία. Τότε ήταν η παλαβή, μία, πάντων, μία περίεργη αριστερά, η οποία δεν ήθελε να κάνει τίποτα. Άφηνε του πρόσφυγε απλώ να εξαφανίζονται. Τώρα έχουμε έναν άλλον υπουργό, έχει αλλάξει η πολιτική, αλλά πάλι φτάσαμε προχθέ να ζητήσουμε ανάπτυξη του μηχανισμού. Δεν έχετε καταλάβει ότι εδώ είμαστε σύμμαχοι. Και ένα δεύτερο, για τι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Είναι αλήθεια ότι η αριστερά αντιμετωπίζει με κάποια φοβία αυτέ τι οργανώσει. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να μιλάει για το ποιοι βοήθησαν το καλοκαίρι στου πρόσφυγε και αυτό που είπε ήταν οι δημοτικέ αρχέ και η Εκκλησία. Δεν έφερε καθόλου την τρομακτική δουλειά που κάνουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Να πάμε λοιπόν όχι μόνο να μην έχει αυτή τη φοβία, αλλά ελπίζουμε από εσά να δημιουργηθεί ένα κάλεσμα προ τι ΜΚΟ και τι ελληνικέ, αλλά κυρίω τι ευρωπαϊκέ, γιατί μόνο αυτό είναι ο τρόπο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα νησιά. Ευχαριστώ. very Σας ευχαριστούμε, συμφωνούμε και αυτό που είπε η κυρία Χολμάιρ ήταν πολύ σημαντικό. Εσείς ε, τελευταία. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ και θα είμαι σύντομη. Είναι ντροπή επαναλαμβάνοντας ε, τα όσα ανέφερε συνάδελφος. Ντροπή είναι το ότι δεν καταφέρνουμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά, να δημιουργηθούν αυτά τα hot spots και υπάρχουν κατηγορίες. Επί μήνες ε, διεξάγονται συζητήσεις και λείπουν τόσα πολλά στοιχεία που η εικόνα ποτέ δεν θα είναι πλήρης δυστυχώς. Με ανησυχεί αυτό το οποίο συμβαίνει και υπάρχουν εναλλακτικέ ιδέες ε, που κυκλοφορούν. Αν αποτύχει η Ελλάδα με τα hot spots, αν δημιουργηθούν μόνο τρία hot spots από τα πέντε και δεν υπάρχει και βεβαιότητα θα λειτουργήσουν και σωστά, τι θα γίνει σε σχέση με τη διαδρομή των Δυτικών Βαλκανίων και τις χώρες αυτές. Αλλού θα προγραμματιστούν τέτοια hot spots και μέχρι πού θα φτάσουμε, ποια θα είναι η τελευταία διαχωριστική γραμμή, το τελευταίο σύνορο και από της τεχνικής πλευράς ακούγοντα ότι και η καταγραφή στην Ελλάδα των ατόμων αυτών δεν γινόταν με τον σωστότερο τρόπο και άλλο συνάδελφος το ανέφερε και για την επιστροφή τους ποιος θα επιληφθεί αυτής της επιστροφής και αυτό θα είναι μείζον θέμα και δεν είναι δυνατόν να σταματήσουν αυτοί οι άνθρωποι, να τους σταματήσει κανείς. Θέλουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους παραπέρα. Το βλέπει αυτό κανείς και στη διαδρομή των Δυτικών Βαλκανίων προς τις βόρειες χώρες της κεντροδυτικής Ευρώπης. Και ερώτηση εδώ, παρέμβαση. Βλέπουμε αποτυχία, μια νέα αποτυχία της πολιτικής μετανάστευσης μας. Όταν λέμε ότι υπάρχει μια ένας μηχανισμός μεταεγκατάστασης χωρίς αποτελέσματα και τώρα υπάρχει η ιδέα των hot και πάλι χωρίς αποτελέσματα Χάνουμε την αξιοπιστία μας δηλαδή εδώ και πολλά διακυβεύονται. Απευθύνω έκκληση λοιπόν να εγγράψουμε αυτό το θέμα ιδιαίτερα υψηλά στην ημερήσια διάταξη να δούμε τι μπορεί να γίνει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν τόσο ακριβείς στην ερώτησή σας. Θα ήθελα και εγώ να κάνω μία ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το IRC. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω κάτι που πιστεύω αφορά όλους μας. Πολλά κράτη-μέλη δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους ε, σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν παρά λοιπόν τις ανάγκες που υπάρχουν. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τι συμβαίνει με αυτόν τον μηχανισμό. Στην ε, παρουσίασή σας μας ε, είπατε πως έχετε δει και άλλες περιπτώσεις τι αναπτυσσόμενες χώρες και πως εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είμαστε προετοιμασμένοι για μια κρίση σε τόσο υψηλά ε, επίπεδα και πως δεν είμαστε καλά προετοιμασμένοι ε, στην Ελλάδα και ε, αλλού. Δεν υπάρχει κάποιος συντονιστής και η κυρία Γκόμες ερώτησε ποιος είναι υπεύθυνο. Κανείς δεν είναι υπεύθυνο, δεν υπάρχει ένας αρμόδιος για να συντονίσει όλους τους υπόλοιπους. Δεν μπορούμε λοιπόν ε, να ε, μιλήσουμε με κάποιον γιατί δεν ξέρουμε με ποιον να μιλήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω, ε, θα συνεχίσουμε με τον εφιστάμενο μηχανισμό ή εμείς ως Ευρωβουλευτές θα έπρεπε να απαιτήσουμε τη δημιουργία ενός νέου πρωτού επιδεινωθεί τόσο άσχημα η κατάσταση που δεν μπορούμε να την διαχειριστούμε καθόλου. Και αναφέρομαι στην διαπαθή των hotspot και όχι τόσο στις συνθήκες υποδοχής διότι πιστεύω πως ε, με τον υφιστάμενο μηχανισμό θα υπάρχει έλλειψη λογοδοσίας, έλλειψη ανάληψης ευθυνών. Αυτή λοιπόν την ερώτηση έχω στην Κομισιόν και στην ε, IRC. Θα αρχίσουμε λοιπόν ε, τον κύκλο των απαντήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις ερωτήσεις σας και τα σχόλιά σας. Δεν είναι δυνατόν φυσικά όλα αυτά να τα απαντήσω γιατί υπάρχουν και πολλές ερωτήσεις που έχουν στραφεί προς άλλους. Αλλά στον πρώτο γύρο αυτό θα κάνουμε αυτή την προσπάθεια, θα δούμε τι απομένει και θα επιστρέψουμε μετά στη συνέχεια αν χρειαστεί. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα απ' όλα να πω δύο λόγια <clears throat> για την χρηματοδότηση. Υπήρξαν αρκετές ερωτήσεις ε, για τη χρηματοδότηση. Τι γίνεται, ποια είναι η κατάσταση. Σύντομα, εν συντομία, ήδη υπό τα διάφορα εθνικά προγράμματα η Ελλάδα έχει περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ από πλευρά κονδυλίων. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι είναι πολύ δύσκολο στην Ελλάδα να έχει πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια λόγω διοικητικών διαδικασιών που πρέπει να λειτουργήσουν και που είναι χρονοβόρες και που όλα αυτά απαιτούν χρόνο. Προγράμματα που πρέπει να αναθεωρηθούν και να επαναξεταστούν για να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία. Λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε μια κατεπίγουσα σύνδρομη βοήθεια σε διαφορετικούς τομείς. Μέχρι στιγμής 50 εκατομμύρια κατεπίγουσας τέτοια σύνδρομης ε, έχουν ε, καταβληθεί στην Ελλάδα και με βάση αυτά μπορούν να καλυφθούν οι πρώτες δαπάνες από την Ελλάδα. Επιπλέον αναμένουμε ότι πολύ γρήγορα θα έχουμε μια ε, μεγάλη συμφωνία μεταξύ ημών και Ηνωμένων Εθνών και είπα της αρμοσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες που επιπρόσθετα θα δώσει τη δυνατότητα διεύρυνσης αυτών των δυνατοτήτων και θα φτάσουν τα κονδύλια για την κατεπίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια σε 130 εκατομμύρια ευρώ. Και πάλι απομένουν ανάγκες που δεν καλύπτονται όλες. Θα υπάρχουν νέα αιτήματα που θα κατατεθούν από τις ε, ελληνικές αρχές, από την ελληνική κυβέρνηση και θα εξετάσουμε να δούμε τι μπορεί να γίνει για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα αυτά, για να κινητοποιηθούν κονδύλια. Αλλά για αυτή τη χρονική στιγμή, για την κατεπίγουσα αυτή φάση, κάλυψη κατεπιγουσών αναγκών, καλύπτονται αυτές με αυτά τα κονδύλια που προανέφερα. Η στέγαση, η δυνατότητα υποδοχής μπορεί να λειτουργήσει, τα προγράμματα μετεγκατάστασης μπορούν να ξεκινήσουν να λειτουργούν και θα υπάρξουν και χρήματα για τις επιστροφές κονδύλια για τις επιστροφές. Αυτή είναι η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί επιτόπου στην Ελλάδα για αυτό το θέμα. Υπήρξαν και αρκετές ερωτήσεις για τις επιστροφές. Γιατί αφενός πώς γίνεται αυτό και αφετέρου πόσοι είναι εκείνοι που θα επιστρέψουν και πού, σε ποιες χώρες. Τώρα, γιατί δεν είναι μόνο η θέση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά είναι και τη ΥΠΑ των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες αυτή είναι ο τρόπος όπου συγκλίνουν όλοι όσοι συνεργάζονται σε αυτό το πεδίο δεδομένων των τεράστιων αριθμών αν θέλουμε να προστατέψουμε εκείνους που πραγματικά έχουν απόλυτη ανάγκη διεθνούς προστασίας ε, τότε αυτό το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν εκείνοι οι οποίοι δεν δικαιούνται και δεν βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση άμεσης ανάγκης θα επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους. Δύο τρόποι υπάρχουν για αυτές τις επιστροφές η εθελοντική επιστροφή, εθελοντικού χαρακτήρα, εθελούσιες επιστροφές και υποχρεωτικές επιστροφές. Οι εθελούσιες μέσα στο πλαίσιο των, το εθελοντικό πρόγραμμα μέχρι σήμερα περίπου 3.500 είναι εκείνοι που επέστρεψαν εθελοντικά. Αυτό ε, επιβραδύνθηκε κατά το μήνα Ιούλιο σε σχέση με τους περιορισμούς άμεσης χρηματοδότησης που υπήρχαν αλλά με την εξέβρεση χρηματοδοτικών λύσεων μπορεί τώρα να επιταχυνθούν οι διεργασίες και πάλι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να σας δώσω ένα παράδειγμα πώς λειτουργούν τα πράγματα. Μια και μπορεί να ακούσατε, να μάθατε ότι μια κατάσταση εξελίσσεται κοντά στα, ε, στα σύνορα της ε, πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Φάιρομ, κατά το τελευταίο διάστημα, που ήταν πολύ δύσκολο για μετανάστες από χώρες όπου δεν υπήρχαν πολεμικές σειράξεις ε, να μπορέσουν να περάσουν τα σύνορα της χώρας αυτής και να συνεχίσουν το ταξίδι τους περαιτέρω. Και αυτοί έμεναν, παρέμειναν στην Ελλάδα. Υπάρχουν από εκείνους ε, κάποιοι οι οποίοι θα μπορούσαν να επιστραφούν και θα πρέπει να δούμε πόσο, κατά πόσο αυτό το πρόγραμμα επιστροφών μπορεί να λειτουργήσει για αυτούς. Αυτό εξετάζουμε τώρα. Το άλλο είναι οι υποχρεωτικές επιστροφές. Και μέχρι σήμερα αυτά βασίζονται σε στατιστικά στοιχεία που έχουμε από τις ελληνικές αρχές, από τους Έλληνες συναδέλφους. 16.131 σε φέτος είναι εκείνοι που ναι, βρέθηκαν υπό διαδικασία επιστροφής. Ο μεγαλύτερος αριθμός σε σχέση με την Αλβανία που βρίσκεται κοντά στη, δίπλα στην Ελλάδα και για τρίτες χώρες πιο απομακρυσμένες, ιδιαίτερα Πακιστάν, Μπαγκλαντές, η κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη. Είναι πολύ πιο δύσκολο να επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί με αυτές τις διεργασίες και αυτό είναι κάτι που βρίσκεται υπό εξέταση και συζήτηση και βρίσκεται στο επίπεδο, ανώτατο επίπεδο διαβουλεύσεων να δούμε τι μπορεί να γίνει σε σχέση με αυτούς. Στην συνέχεια υπήρξαν και ερωτήσεις που τέθηκαν για τη μετεγκατάσταση και αναφέρθηκε αυτό γιατί λέει είναι δύσκολη η μετεγκατάσταση. Δεν είναι η δυσκολία η χρηματοδότηση. Τα κονδύλια υπάρχουν. Μπορεί να λειτουργήσει η μετεγκατάσταση αλλά υπήρξε περιορισμένη ζήτηση παρότι σε σχέση με τα όσα είχαμε στην αρχή υπάρχει κάπως μεγαλύτερη ζήτηση σήμερα από ό,τι κατά το παρελθόν. Και πάλι βλέπουμε εδώ ότι τίθεται το ζήτημα του να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα προβλήματα, τις διάφορες στενοπούς. Παράδειγμα, ζήτηση. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα προς ενημέρωση το ένα ή το άλλο πρέπει να αυξήσουμε το επίπεδο εμπλοκής και προσπάθειας που καταβάλλεται για να τα καταφέρουμε. Ένα άλλο θέμα τώρα είναι η στέγαση, οι δυνατότητες στέγασης. Αν θέλει κανείς να υποβάλει αίτηση για μετεγκατάσταση πρέπει για το διάστημα προς το, που θα μεσολαβήσει μέχρι ότου μετεγκατασταθεί πρέπει να στεγαστεί και πρέπει να μπορέσει να στεγαστεί και να συστηθεί. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν αυτή η προσπάθεια διασφάλισης αυτής της στέγασης με την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών. Και ένα τελευταίο ζήτημα εδώ. Υπάρχουν και τα άλλα κράτη-μέλη. Υπάρχουν υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερης εμπλοκής ε, και συμμετοχής των κρατών μελών. Αλλά πρώτον χρειαζόμαστε πολύ ταχύτερες διαδικασίες ε, για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών. Άτομα που θα ζητήσουν να μετεγκατασταθούν να γνωρίζουν ότι σε άμεσο μικρό χρονικό διάστημα θα μπορέσουν να μετεγκατασταθούν. Ενώ σήμερα αυτές είναι ε, χρονοβόρες διαδικασίες. Για οποιαδήποτε άλλα θέματα μπορούμε να επιστρέψουμε στη συνέχεια, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα δούμε λοιπόν αν ε, έχουμε χρόνο στο τέλος γι' αυτό. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις. Η κυρία Καραγγέλη τώρα έχει το λόγο. Σας παρακαλώ προσπαθήστε να κρατήσετε τα τρία λεπτά. Πολύ. Έχω πάρα πολλέ ερωτήσει, τι οποίε καλούμε να απαντήσω. Θα φροντίσω και εγώ να είμαι λιγάκι περιεκτική σε αυτά που θα πω και ελπίζω σε ένα δεύτερο γύρο. Ε, έχω κρατήσει τις πολλές απορίες σχετικά με τις επιστροφές. Θέλω να συμπληρώσω σε αυτά που υπόθηκαν λίγο πριν, ότι έγινε προσπάθεια επιστροφής, νομίζω ότι είναι γνωστό το περιστατικό, 2 Δεκεμβρίου με την πρεσβεία του Πακιστάν. Ε, και εδώ δεν είναι θέμα μόνο ελληνικό, είναι θέμα και ευρωπαϊκό, έχω την αίσθηση. Ε, από τους ανθρώπους που είχε συμφωνηθεί να επιστραφούν στο Πακιστάν, το Πακιστάν δεν τους έκανε δεκτούς την πρώτη φορά καθόλου και τη δεύτερη φορά που είχε συμφωνηθεί 2 Δεκεμβρίου έκανε δεκτούς τους μισούς. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε όλοι μαζί αυτό. Ε, τι είναι τα hot spots, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να ε, απαντήσω λιγάκι στο τι είναι τα hot spots, ε, αφού το άκουσα τόσες πολλές απορίες για το πώς λειτουργούν και τι κάνουν. Ε, να ξεκινήσω λέγοντας και υπογραμμίζοντας ότι οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης στην Ελλάδα γίνονταν έτσι ακριβώς όπως έχει οριστεί αυτή τη στιγμή να γίνονται μέσα στα hotspots. Αυτό το οποίο αφορά στην Ελλάδα για τη δημιουργία των hot έχει περισσότερο να κάνει με το accommodation. Πράγματι, υπήρχαν σκηνέ για τι οποίε δεν νιώθουμε περήφανοι, ούτε σαν Έλληνε ούτε σαν Ευρωπαίοι. Να μην ξεχνάμε όμω ότι είναι μια χώρα εν μέσω κρίση που ούτε στου δικού τη ανθρώπου πολλέ φορέ δεν μπορεί να προσφέρει τα απαραίτητα. Και καλεστήκαμε στην καρδιά του καλοκαιριού και σε συνέχεια τώρα να ανταποκριθούμε σε μια πολύ μεγάλη ανθρωπιστική κρίση που ήρθε μέσα σε μια δική μα εσωτερική ανθρωπιστική κρίση. Ε, σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις δεν θέλω να αναφερθώ γιατί θεωρώ ότι έχει απαντηθεί αυτό το σκέλος. Ε, το Δουβλίνο, ναι, θεωρώ ότι χρειάζεται ε, διορθώσεις, όχι γιατί το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι άνθρωποι που θέλουν να υποβάλουν αιτήματα ασύλου ή relocation, αλλά φοβούνται πάρα πολύ τις καθυστερήσεις που μπορεί να υπάρχουν σε αυτές τις διαδικασίες και στα σίγουρα ε, υπάρχουν ε, καθυστερήσεις οποίες πρέπει όλοι μαζί να δούμε πώς θα διορθώσουμε και πώς θα γίνουν ταχύτερες οι, ε, ε οι γραφειοκρατικές ε, διαδικασίες. Ε, τα κέντρα, τα hot spots σίγουρα δεν θα δημιουργηθούν και δεν θα γίνουν κέντρα κράτησης. Υπόθηκε, δεν θυμάμαι από ποιον, αλλά δεν έχει κανένα στο μυαλό της πολιτική να γίνουν κέντρα κράτησης. Ακόμα και οι άνθρωποι που πρέπει να επιστραφούν για τους λόγους που αναφέρθηκαν πριν, ε, νομίζω ότι είναι πολιτική απόφαση της Ελλάδος και το έχει επανειλημμένα τονίσει για γρήγορες επιστροφές δεν υπάρχει πρόθεση αυτοί οι άνθρωποι και άλλωστε νομίζω ότι η νομοθεσία τη χώρα μου τη γνωρίζει την τέτοια που δεν επιτρέπει στην κράτηση αυτών των ανθρώπων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουμε. Και εδώ πάλι έχω την αίσθηση ότι είναι κοινή η προσπάθεια και όχι μόνο από την πλευρά τη Ελλάδο για τον αριθμό των διαβατηρίων των πλαστών που υπόθηκε για τις διαδικασίες αυτές νομίζω ότι ε, δεν έχω αυτή τη στιγμή στοιχεία να σας δώσω. Καταλαβαίνετε ότι είναι εύλογο να μην έχω στοιχεία να σας δώσω αυτή τη στιγμή. Ε, δεν ξέρω συνάδελφος ότι τη Φρόντοξα μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. να πω για την πολιτική προστασία που άκουσα πάρα πολλά και καλούμε να απαντήσω. Ε, δεν υπήρχε ίσως ο μηχανισμός για τη σωστή το βάζω συσταγωγικά, κατανομή όλων αυτών. Όταν καλείσαι να αντιμετωπίσει σχεδόν 500.000 ανθρώπους μέσα σε ένα τρίμηνο, καλείσαι πρώτα να αντιμετωπίσει το άμεσο και στη συνέχεια να καταγράψει και οργανωμένα να μπορέσει να ζητήσει τη βοήθεια την οποία τώρα ζητάμε και μπορούμε να κατευθύνουμε στα σωστά σημεία. Ε, καταλαβαίνετε ότι στην καρδιά του καλοκαιριού και έκτοτε, και αναφέρομαι και στον Οκτώβριο γιατί έτυχε να τον ζω από κοντά στην ε, σχεδόν, ε, αυτό που περιγράψατε πριν ως συνοστισμός ε, ήταν συνοστισμός λόγω του ότι ερχόντουσαν 10.000 άνθρωποι στο νησί που έπρεπε να καλυφθούν ανάγκες και καταγραφής αλλά ταυτόχρονα και σύντησης. Και όλο αυτό έχει μια δυσκολία από μόνο του. Ε, και να κλείσω ε, λέγοντας και σχολιάζοντας λιγάκι για τις ΜΚΟ και εγώ, αρκετέ φορέ στο εσωτερικό τη χώρα. Νομίζω ότι και ο ίδιο Υπουργό Μεταναστευτική Πολιτική έχει αναφερθεί στη βοήθεια που έχουν προσφέρει, αλλά ταυτόχρονα και στην ανάγκη που υπάρχει για ένα προγραμματισμό και μια οργάνωσή του, έτσι ώστε να μην υπάρχει ε, αρκετό ανθρώπινο δυναμικό που θέλει να προσφέρει βοήθεια και να μην μπορεί να προσφέρει κατευθυνόμενο. Ε, θα μπορούσα να πω και άλλα, αλλά ο χρόνο μου. Thank you. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Σέμπρι. αν θέλετε, έχετε τρία λεπτά. Θα προσπαθήσω λοιπόν να απαντήσω σε ορισμένε από τι ε, ερωτήσει. Ε, κύριε Χολμάιερ, καταρχά σχετικά με τι ανάγκε που έχουμε σε προσωπικό αυτή τη στιγμή. Όταν λειτουργήσουν όλα τα hot spot, υπολογίζουμε σε 60 ε, ανθρώπους να είναι στην Ελλάδα, full time. Τώρα, σε σχέση με το σχεδιασμό πρέπει να είμαστε αρκετά ευέλικτοι σε σχέση με το πού θα πάει ο καθένας. Τώρα, ε, όσο για τις προκλήσεις, αυτό που ανέφερε η κυρία Μετσόλα, καταρχάς πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε σε όλες τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ίσως κάτι άλλο που θα παει ο καθενας τωρα οσο για τις προκλησεις αυτο που ανεφερε η κυρια μετσολα καταρχας πιστευω πως η ευρωπαικη επιτροπη αναφερθηκε σε ολες τις προκλησεις που εχουμε να αντιμετωπισουμε ισως κατι αλλο που θα μπορουσα να πω είναι τα σημεία πληροφόρησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να ενισχύσουμε τις ε, μεθόδους για πληροφόρηση που έχουμε στα ε, hotspot, να βοηθήσουμε ε, σχετικά με την ζήτηση, να υπάρχει μεγαλύτερη απορρόφηση ανθρώπων στα πλαίσια της μεταγκατάστασης και πιστεύω επίσης πως στην ερώτηση για το πώς προσπαθούμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη να ε, μας διαθέσουν περισσότερους εμπειρογνώμονες, να σας πω πως επικοινωνούμε με το Διοικητικό μας Συμβούλιο και έχουμε κάνει μια έκκληση στο Συμβούλιο την περασμένη Παρασκευή, όπου ζητήσαμε περισσότερους εμπειρογνώμονες. Να γνωρίζετε όμως ότι αυτή τη στιγμή το θέμα αυτό δεν είναι τόσο επίγον, διότι δεν λειτουργούν πλήρως τα hotspot. Μόλις λειτουργήσουν, τότε ναι, θα χρειαστούμε περισσότερη βοήθεια. Ο κύριος Ρόσλερ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, θα εστιάσω σε τρία-τέσσερα σημεία και θα προσπαθήσω να συνοψίσω. Καταρχάς, ε, να πω ότι η Frontex στηρίζει τις αρχές ε, στο screening, στη διάγνωση, στον εντοπισμό της εθνικότητας, έπειτα, δακτυλικά αποτυπώματα. Υπάρχει ένα σύστημα που προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ταυτοποιήσουμε τους ανθρώπους. Επίσης προσπαθούμε να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με, ποινικές, ε, με ποινικό μητρό. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ε, δημιουργία ε, αιτήσεων ασύλου, δεν είμαστε υπεύθυνοι, δεν χορηγούμε άσυλο, παραπέμπουμε στις αρμόδιες ε, αρχές και επίσης δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ε, διαδικασία επιστροφής. Αυτό είναι αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Έπειτα, οι πόροι που διαθέτουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 260 ε, υπαλλήλους που στηρίζουν τα πέντε hot spots, τα πέντε νησιά και ενδεχομένως χρειαστεί και ο ίδιος αριθμός για την ε, στήριξη και επιτάχυνση της ε, διαδικασίας σε βάρδιες από τη στιγμή που λειτουργήσουν τα hot spots στα υπόλοιπα νησιά. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί και από την δυνατότητα φιλοξενίας των αρμόδιων εθνικών αρχών. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τις ε, εθνικές αρχές και δεν μπορούμε να είμαστε πάνω από το 25% των διαθέσιμων πόρων για την ε, διαδικασία ε, αυτή. Η Frontex δεν είναι η αρμόδια αρχή επίσης για να διατηρήσει μία εύρυθμη κατάσταση στα σημεία αυτά ή για να μεταφέρει τους ε, πρόσφυγες από τα νησιά αλλού. Αυτό είναι αρμοδιότητα εθνική. Και τέλος, από ό,τι καταλαβαίνουμε, υπάρχει ανάγκη για περισσότερη πληροφόρηση των ε, μεταναστών σχετικά με τις ε, διαδικασίες ασύλου για να αποτρέψουμε, για παράδειγμα, συμπλοκές ή διάφορες άλλες τέτοιες δυσάρεστες ε, συνθήκες. Στα τέλη Οκτωβρίου έγινε μια ε, συνάντηση για τα Δυτικά Βαλκάνια και αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί ε, στα ελληνικά σύνορα με την Πουγουδουμού ένα σύστημα καταγραφής έτσι ώστε να στηρίζονται οι προσπάθειες καταγραφής και ταυτοποίησης μέσω της ε, Eurodac όσων δεν έχουν ήδη καταγραφεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε επισκεφτεί αυτές ε, τις ε, τοποθεσίες έτσι ώστε να διαπιστώσουμε τι ακριβώς θα χρειαστούμε. Βρισκόμαστε λοιπόν σε στάδιο σχεδιασμού μέχρι να οδηγηθούμε στην συμφωνία με τις ελληνικές αρχές και σε σχέση με την δευτερογενή μετακίνηση στα σύνορα Κροατίας και Σλοβενίας. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ενισχύσουμε την παρουσία μας εκεί και να στηρίξουμε τις εθνικές αρχές. Δεν υπάρχει ακόμα η σύμφωνη γνώμη των αρχών της Κροατίας για την εφαρμογή περισσότερων ε, δράσεων παρακολούθησης στα σύνορα με την Σερβία. Ευχαριστώ. Η κυρία Φορτιά έχει το λόγο. Η πρώτη ερώτηση ήταν σε σχέση με το τι μπορεί να γίνει. Είχαμε μια θετική σχέση με τις ελληνικές αρχές. Αυτό που λείπει όμως είναι η δυνατότητα λήψης αποφάσεων στο αναγκαίο ε, επίπεδο στο οποίο πρέπει να λαμβάνονται άμεσα, καθώς επίσης και με έναν ηγετικό ρόλο όσον αφορά το συντονισμό. Αναμένουμε να αναλάβει περισσότερο ηγετικό ρόλο η Ελλάδα και στην στο να συμμεριζόμαστε τις πληροφορίες μέχρι την, το τελικό επίπεδο λήψης απόφασης, λήψης αποφάσεων, ώστε να μπορούν οι υπηρεσίες να παρέχονται σε όσους έχουν ανάγκη αυτές, αυτές τις υπηρεσίες. Σε σχέση τώρα με την ε, βίαιη αντίδραση όταν υπάρχουν στενοποί, δεν είναι θέμα του να μην υπάρχουν επαρκή στελέχη επιτόπου, είναι το να μην υπάρχουν προβλήματα τα οποία θα οδηγούν σε τέτοιες ε, εντάσεις. Θα πρέπει λοιπόν και πάλι εδώ με το αυξημένο δυναμικό από πλευράς ελληνικών αρχών να μπορούμε με την διάχυση πληροφοριών να γνωρίζουμε αμέσως το τι συμβαίνει. Υπάρχει αυτή η πίεση λοιπόν που πρέπει να μπορεί έτσι άμεσα να αντιμετωπίζεται. Και το δεύτερο ε, σκέλος της ερώτησης όταν ε, υπάρχει ένταση μεταξύ διαφορετικών εθνοτήτων ή ε, εθνικοτήτων και πρέπει εδώ να δούμε λοιπόν ε, το πρόβλημα αυτό να έχουμε, να διασφαλίζουμε ότι όλοι θα έχουν πρόσβαση, να υπάρχει προσπελασιμότητα στην ίδια ταχύτητα και ρυθμούς καταγραφής και διεκπαιρέωσης. Και από πλευράς επιμελητίας μπορούμε να πούμε ότι τα πράγματα όταν μπορούν να λειτουργήσουν ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των όσων φτάνουν στην Ελλάδα γιατί διαφορετικά η κατάσταση θα είναι αφόρητη επίσης ε, για τις γυναίκες, τα παιδιά και τα μη συνοδευόμενα ανήλικα κάνουμε μια επισκόπηση αποκινούμε την UNICEF δεν έχω τις λεπτομέρειες αλλά μπορώ να ε, επανέλθω στο θέμα αυτό και να σας διαθέσω τα στοιχεία ιστερότερα για τους μηχανισμούς από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή υποστήριξης αντιμετώπισης της κρίσης, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε με τα βιώματά μας και την πείρα που συλλέγουμε στα σύνορα και με τους μηχανισμούς που θα έπρεπε να μπορούν να λειτουργήσουν για τη χρηματοδότηση, για την ανθρωπιστική βοήθεια, ΕΚΟ και τον συντονισμό. Υπάρχει βραδύς ρυθμός ε, ε, αντιμετώπισης. Ε, αντιμετωπίζουμε θέματα τα οποία πρέπει να μπορούν να είναι αποτελεσματικά στα σύνορα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ιδιαίτερη λοιπόν ικανοποίηση όταν θα υπάρξουν αυτές οι δυνατότητες να υπάρχει ευελιξία και να μην είναι μια κατάσταση η οποία θα αντιμετωπίζεται απλά και μόνο με την σύνδρομη μηχανισμών του, της ΕΚΟ, ε, του Μηχανισμού Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Πρέπει να εξευρεθούν δυνατότητες άμεσης αντίδρασης, πιο γοργής αντίδρασης στο μέλλον. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους και όλους όσους παρενέβησαν για σε αυτή τη σημαντική συζήτηση. Και θα περάσουμε τώρα στο θέμα των hot spots στην Ιταλία και είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ να μπορέσουμε να επικεντρωθούμε επίσης ε, στα θέματα των hotspots ε, των κομμικών αυτών κέντρων στην Ιταλία για να συμπληρωθεί η συζήτηση με αυτό το σκέλος. Να μείνετε στις θέσεις σας, ε, θα αλλάξουν κάποιοι από τους συμμετέχοντες στο πάνελ εδώ γιατί θα υπάρξει αλλαγή ομιλητών και θα έχουμε μια βιντεοσκοπημένη διάσκεψη, ένα τμήμα βιντεοσκόπησης όπου παρα, παρα, παρακαλώ να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Daniela. Alors, on ne vous voit pas. On ne voit rien du tout.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 ε, Miss Viviana Balastro. Είναι η κυρία Βιβιάνο Παλάστρο. Με ακούτε? You can, yeah. Ναι, μπορείτε να ξεκινήσετε. Ε, μάλλον όχι. At your end and then we can begin the, the next session. Is that okay? Ε, ε, θα πρέπει να μην μιλήσετε για λίγο από τη δική σας πλευρά για να σας πω πότε θα ξεκινήσουμε. Okay. Uh, to a, quick start now because we we've lost some time. Πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν άμεσα γιατί έχουμε χάσει λίγο χρόνο και δεν είναι σωστό να μην έχουμε αρκετό χρόνο για το δεύτερο τμήμα όσο είχαμε τουλάχιστον και για το πρώτο. Θα δώσω αμέσως το λόγο ε, στην ανάλυση της ε, κατάστασης στα hot spot της ε, Ιταλίας. Παρακαλώ συνάδελφοι ησυχία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους που παρέμειναν. Ξέρω ότι γίνονται, είναι ένα πολύ έντονο απόγευμα. Θα αρχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, με παρουσιάσεις από τον εκπρόσωπο της DG Home. Ε, πέντε λεπτά θα μας μιλήσει για την κατάσταση. Thank you, Mr. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω να υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον για την Ιταλία όπως υπήρχε και για την Ελλάδα. Θα ήθελα να πω αρχικά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα θα δημοσιεύσει μία έκθεση για τα hot spot στην Ιταλία και την Ελλάδα. Στις 15 λοιπόν του μήνα θα έχετε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση στις δύο αυτές χώρες. Η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική στην Ιταλία σε σχέση με την Ελλάδα για πολλούς λόγους. Διότι τα νούμερα είναι διαφορετικά. Όπως γνωρίζετε, ο αριθμός των μεταναστών στην Ελλάδα είναι πολύ μικρότερος από ότι στην Ελλάδα. 150.000 έχουν φτάσει στην Ιταλία φέτος και οι Ιταλικές αρχές είχαν περισσότερο χρόνο να προετοιμαστούν, διότι δεν βρίσκονταν σε ε, κρίση όπως στην Ελλάδα και δεν είχαν ε, πίεση τα προηγούμενα έτη. Υπήρχαν σταθερές ερωές σε μεταναστών που έφταναν τα προηγούμενα έτη, γι' αυτό λοιπόν είχαν χρόνο να προετοιμάσουν τα hotspot. Όπως και στην Ελλάδα, έτσι και εδώ αναπτύξαμε μια ομάδα ε, τα, στο έδαφος της Ιταλίας και προσπαθήσαμε να συντονιστούμε με τις Ιταλικές αρχές. Ένα hot spot υπάρχει αυτή τη στιγμή που είναι πλήρως λειτουργικό στην Λαμπεντούσα. Σε σχέση λοιπόν με την Ελλάδα, εμείς έχουμε μόνο ένα hot spot στην Ιταλία που ε, λειτουργεί. Επισκεφθήκαμε πολλές φορές τις εγκαταστάσεις σε αυτό το hot spot και η Frontex και η EASO, αλλά ε, και διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις, η IOM και η Save the Children δραστηριοποιούνται εκεί. Ε, οι άνθρωποι ε, καταγράφονται, παίρνονται τα δακτυλικά αποτυπώματα, υποβάλλονται σε ιατρικά check-up και διαρευνούνται οι δυνατότητες μεταγκατάστασης για όσους την δικαιούνται. Επίσης, προσπαθούμε να συλλέξουμε πληροφορίες για τις ε, οδούς διακίνησης ανθρώπων και συνεργαζόμαστε με την ε, Europol γι' αυτό. Και να σας πω ότι την Παρασκευή που μας πέρασε η Europol με τη Frontex υπέγραψαν μια συμφωνία για ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις δύο υπηρεσίες που θα διευκολύνει την ε, δουλειά τους. Λοιπόν, το hotspot αυτό στη Λαμπεντούσα είναι πλήρως λειτουργικό. Ε, μας ανησυχεί η έλλειψη προόδου στα άλλα υπόλοιπα hot spot. Οι εγκαταστάσεις στο Ποτσάρο και στην ε, Λεσχανία θα μπορούσαν να είναι έτοιμες, όμως ακόμα περιμένουμε τις ε, πολιτικές αποφάσεις, την πολιτική έγκριση, έτσι ώστε να γίνουν και αυτά τα hot spot πλήρως λειτουργικά. Ελπίζω μέχρι το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός Ρέντσι να δώσει το OK για να γίνουν πλήρως λειτουργικά και τα υπόλοιπα δύο hotspot. Στην Αγκούστα, στο Ταράντο και στο Τράμπανι χρειάζεται να γίνουν πολλά ακόμα για τη δημιουργία των hotspot, όμως και εκεί βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά στην ε, τελική λειτουργία τους ε, και ελπίζουμε να υπάρχουν σύντομα αρκετά hotspot έτσι ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε τις μεταναστευτικές ροές επαρκώς. Αυτή τη στιγμή έχουμε 500 διαθέσιμες ε, μονάδες στην Ελαμπεντούσα, κάτι που δεν επαρκεί. Αν δείτε για παράδειγμα αυτό που έγινε την τελευταία εβδομάδα, όπου είχαμε πάνω από 5.000 μετανάστες που έφτασαν ταυτόχρονα στο νησί, καταλαβαίνουμε ότι οι εγκαταστάσει είναι ανεπαρκείς και ότι η Λαμπεντούσα δεν μπορεί μόνη της να ανταπεξέλθει. Αυτή είναι και η κυριότερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα, ε, πέρα από τα hot spots, σχετικά με το σύστημα μετεγκατάστασης, η Ιταλία έχει κάνει τους ε, κατάλληλους διακανονισμούς έτσι ώστε να προωθηθούν οι περιπτώσεις μετεγκατάστασης. και ε, δερμολογούνται διαδικασίες καταγραφής και αξιολόγησης. Να πω επίσης ότι πολλοί μετανάστες φτάνουν στην Ιταλία ε, οι οποίοι δεν ετούνται άσυλο, δεν μπορούν να αποφαληθούν του συστήματος αμετεγκατάστασης. Και ε, βλέπουμε ότι πρόσφατα έφτασαν πάρα πολλοί άνθρωποι από την Δυτική Αφρική, οι οποίοι χρειάζεται να επιστρέψουν τις ε, χώρες τους. Χρειάζεται λοιπόν η Ιταλία να εντείνει τις ε, προσπάθειες ε, επιστροφής και είναι κάτι αρκετά δύσκολο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ιταλία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις χώρες της Δυτικής Αφρικής έτσι ώστε να δρομολογηθεί η επιστροφή των μεταναστών. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ κύριε Μισελ. Ε, ο Μορκόνε έχει τώρα το λόγο, επικεφαλής της Ιταλικής ε, Αντιπροσωπείας Πολιτικών Ελευθεριών και Μετανάστευσης. Την τελευταία φορά που ήσασταν εδώ μας παρουσιάσατε με αρκετέ λεπτομέρειες την κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε ξανά σήμερα για να μας ενημερώσετε. Έχετε 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κυρίως γιατί μου δώσατε για μία ακόμα φορά την δυνατότητα να εξηγήσω αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στην Ιταλία. Ε, ενώ ήδη ακούσατε και από τον κύριο Μουσέλ ε, τα στοιχεία τα οποία έχουμε. Έχουμε παραπάνω από 300.000 ανθρώπους αυτή τη στιγμή, αλλά κυρίως μεγάλο αριθμό ε, ασυνόδευτων ανηλίκων, πρόβλημα ιδιαίτερα μεγάλο. Επίσης, ε, όσον αφορά τους ετούντες άσλο, τους πρόσφυγες, έχουμε τα, τις ΣΠΡΑΡ που είναι κέντρα που υποδέχονται χιλιάδες ε, ενήλικες και χίλιους ε, ανηλίκους. Ε, όλα αυτά βεβαίως τα κάνουμε σε συνεργασία με μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, με την Υπατιαρμοστία, με το IOM και το Save the Children και σε μερικές περιπτώσεις και με τον Ερυθρό Σταυρό. Ερχόμενος σε το κύριο πρόβλημα που είναι τα hot spots και η relocation, να σας εξηγήσω πώς έχουν τα πράγματα. Ο κύριος Μουσέλ ήδη έδωσε το πλαίσιο της ε, κατάστασης, αλλά <coughs> η άποψη της χώρας μου, της χώρας μου ε, προσπαθεί να εξισορροπήσει την ε, αλληλεγγύη με την υπευθυνότητα. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει ότι η ιδέα που έχουμε είναι ότι τα hot spots θα ανοίγουν σιγά σιγά όσο προχωράει και η relocation. Είναι αλήθεια ότι ε, η κατανομή είναι ακόμα πολύ μικρή γιατί ήταν λίγες οι αποβάσεις μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα. Γι' αυτό καταφέραμε 135, 130 ανθρώπους ε, να ε, τοποθετήσουμε, αλλά και ίσως λόγω του μεγάλου, ε, της μεγάλης ανησυχίας, του μεγάλου κλίματος ανησυχίας που προκλήθηκε μετά από τα αιματηρά γεγονότα στο Παρίσι όπου έχασαν τη ζωή τους τόσοι άνθρωποι. Αυτές οι 137, αυτοί οι 137 άνθρωποι που είμαστε έτοιμοι να με μεταφέρουμε στην Ισπανία αλλά και στη Γαλλία, στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην ουσία εδώ και με πολλές εβδομάδες δεν έχουν καταφέρει να μετακινηθούν. Αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης που λέει εμείς είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τουλάχιστον τέσσερα hot spots από τα έξι που, ε, υπάρχουν, που προβλέπονται στην Ούκμα. Ε, ήδη στην Λαμπεντούζα υπάρχει άλλο ένα ε, τα hot spot του Τάραντο και της Αγγούστα χρειάζονται ακόμα λίγο χρονικό διάστημα, μερικές εβδομάδες, αλλά οπωσδήποτε αυτή η κίνηση θα πρέπει να βρει σαν αντίβαρο την αλληλεγγύη ε, ε, που έχουν αναγγείλει οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή είναι η πολιτική βεβαίως επιλογή της χώρας μου. Ε, άλλωστε αυτό το θέμα το ε, ε, υποβάλαμε και σε το Συμβούλιο Τζάι της ΔΕΗ της Παρασκευής. Βεβαίως πρέπει να σημειώσουμε ότι έχουμε όλο και περισσότερους Αφγανούς και Πακιστανούς που φτάνουν από το Φρίουλι, από τα βόρειο-ανατολικά σύνορα μέσω Αυστρίας, Γερμανίας, Βένετο. μπορώ να καταλάβω την ε, προϋπόθεση, την κατάσταση των Παγκλαντεσιανών και των Πακιστανών, αλλά το θέμα των Αφγανών είναι ένα θέμα το οποίο εμείς έχουμε υποβάλει επισταμένως ε, εις ε, το ε, Συμβούλιο Δικαιοσύνης, ε, γιατί είναι ένα ειδικό θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί και στα πλαίσια της ε, relocation, γιατί έχει ξεκινήσει μια νέα διαδρομή από το Φρίουλι Βενέτσια Τζούλια, από τα βόρειο-ανατολικά μας σύνορα. Προηγουμένως έγινε λόγος στην δυσκολία που έχει προκύψει στα συνορα Ελλάδας Φύρομ. Ξέρω ότι η ε, Φύρομ ε, ε, σταματάει μεγάλους αριθμούς ανθρώπων που προσπαθούν να φτάσουν στην, στον χώρο Σέγγεν. είναι άνθρωποι οι οποίοι μέσω των Δυτικών Βαλκανίων θα προσπαθήσουν να φτάσουν μέχρι το Φρίουλι, μέχρι την Ιταλία. Υπάρχουν βεβαίως και κάποια στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τις αποφάσεις ε, του θεματολογίου ε, Γιούγκερ που εμείς έχουμε ενστερνιστεί ε, και που ενδεχομένως θα πρέπει να τους ξαναδούμε λίγο. Οι διαδικασίες είναι εξαιρετικά περίπλοκες και θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν πιο απλές και θα πρέπει να είναι και πιο γρήγορες οι απαντήσεις των χωρών που δέχονται την κατανομή των ε, προσφύγων, γιατί και εδώ είναι ένα θέμα το οποίο συχνά απαιτεί πολύ χρόνο. Είναι σαφές ότι ε, ας πούμε για, στους ε, προερχόμενους από την Ερυθρέα μπορώ να, δώσω, να τους δώσω μία διαδικασία έτσι ώστε να τους πείσω να περάσουν από τις διαδικασίες ταυτοποίησης, ταυτοποίησης της Eurodac ε, διαβεβαιώνοντάς τους ότι θα πάνε στην Ισπανία και μετά η Ισπανία και το λέω έτσι για παράδειγμα μετά η Ισπανία κάνει τρεις ή τέσσερις εβδομάδες μέχρι να απαντήσει οι άνθρωποι αυτοί δεν ε, θα πιστέψουν ότι εγώ λέω αλήθεια, θα πιστέψουν αντιθέτως ότι τους έχω κοροϊδέψει. Αυτό λοιπόν το θέμα της έγκαιρης ε, υποδοχής ε, είναι κάτι σημαντικό και θα ήθελα να παρακαλέσω εδώ όλους τους φίλους τους οποίους στέλνουμε τα αιτήματα, τα έντυπα, να απαντούν γρήγορα Ίσως υπάρχουν ε, κάποια ε, ευρωπαϊκά συστήματα τα οποία ε, βασίζονται σε μεγαλύτερο διάστημα αλλά φοβούμε ότι αυτά τα μεγάλα χρονικά διαστήματα θα δημιουργήσουν πρόβλημα εν τέλει. Και αυτά ήθελα να σας πω. Εάν θέλετε να υποβάλλετε ερωτήματα, είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μορκόνε από Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα επεξηγήσω τις κύριες λειτουργίες μας και το πώς εργαζόμαστε. Όσο, όπως προηγούμενα επεξήγησα, εργαζόμαστε με βάση ένα λειτουργικό πρόγραμμα του, των, για τα hotspots και συζητάμε για τις τελευταίες φάσεις ε, με την Ιταλική κυβέρνηση για την υπογραφή αυτού του λειτουργικού προγράμματος. Στο μεσοδιάστημα όμως εντωμεταξύ έχουμε τρεις κύριες λειτουργίες ε, Πρώτον, διάθεση πληροφοριών που πρέπει να διασφαλίσετε για την επαναγκατάσταση και για την χορήγηση ασύλου, καταγραφή, δεύτερον, καταχώρηση και για την ε, απόφαση που, παροχής προστασίας και την ε, ε, αντιστήχηση αντίστοιχων ε, χαρακτηριστικών ώστε να μπορέσουν τα προγράμματα των κρατών μελών να λειτουργήσουν. Στην Λαμπεντούζα υπάρχει το έργο αυτό που εκτιλήσεται. Έχουμε ε, στην Βίλα Σικάνια μια ομάδα ε, αξιωματούχων επαϊόντων που εργάζονται σε αυτή την καταγραφή και στην Κουεστούρα τέσσερις αξιωματούχοι και άλλοι τέσσερις σε άλλη μονάδα που ε, συνοδεύουν αυτό το έργο. Επίσης ε, με τη μονάδα ε, για την, τις διαδικασίες Δουβλίνου στη Ρώμη για την αντιστήχηση στοιχείων για να μπορέσουμε να δούμε πώς λειτουργούν όλα αυτά θα επενδύσουμε περισσότερο στην συνεργασία με ΜΚΟ, μη κυβερνητικέ οργανώσεις επιτόπου οι κύριες προκλήσεις στην Ιταλία όπως προαναφέρθηκε είναι ο αριθμός των ε, νεοαφικνούμενων ε, με την ε, υπηκότητα εκείνων που θα επιλέγονται για μετεγκατάσταση. Έχουμε όμως και κατά τις τελευταίες τρεις-τέσσερις ημέρες αυξημένο αριθμό. Πρέπει να επικεντρωθούμε στην χορήγηση συνδρομής ακόμα και εκτός hotspots με κινητές ομάδες, mobile teams και δραστηριότητες σε σχέση με μετανάστες στα ε, ε, κομβικά σημεία ε, διαμετακόμισης. Επίσης η ελαστικότητα, η ευληγησία πρέπει να είναι κάτι που θα τονίσουμε στη σπουδαιότητά του. Είναι ανάγκη λοιπόν να έχουμε ευλίγησες, ελαστικές προσεγγίσεις για αυτές τις ανάγκες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Εσείς από πλευράς Frontex έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ξεκινήσω κάπως ε, λέγοντας πώς έχει η κατάσταση επιτόπου. Οι συνολικές αφήξεις στην Ιταλία μειώθηκαν σε σχέση με πέρυσι κατά περίπου 10 ή 11% στην κεντρική διαδρομή της Μεσογείου. 144.000 συν 4.600 μη επιβεβαιωθέντες για την αποβίβασή τους. Frontex στην Λαμπεντούσα, 24 αξιωματούχοι στο Ποτσάλο, καθώς επίσης και σε άλλες τοποθεσίες, σε άλλα λιμάνια, όσον αφορά τις αποβιβάσεις, 28 αξιωματούχοι και εκτός hot spots επίσης και σε σχέση με το Κροτόνε, Σιρακούζα και Κατάνια έχουμε 15 ομάδες ε, καταγραφής και ανείχνευσης. Ε, σε σχέση με τη Λαμπεντούζα ε, προχθές ήδη είχαμε ε, νέες αφήξεις και στην Αυγούστα 394 που αφήχθησαν οι συνθήκες και όροι υποδοχή στην Αυγούστα και στο πόρτο εμπεντόκλε του Ακράγαντα και για την συστηματική καταγραφή και την δακτυλοσκόπηση και ταυτοποίηση των ατόμων αυτών. Οι προκλήσεις παραμένουν λοιπόν υπάρχει ανάγκη να έχουμε τα πρώτα κέντρα υποδοχής που θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. Είναι επιτακτική ανάγκη για την προσέγγιση hot spots αυτό και ελπίζουμε ότι γοργά θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Η ανείχνευση, η καταγραφή πρέπει καλύτερα να εντάσσεται στη σφαιρική αυτή διαδικασία συνολικά στα πρώτα κέντρα υποδοχής δεν επιτρέπουν οι όροι ε, υποδοχής αυτή την καταγραφή αυτή τη στιγμή όπως θα έπρεπε. Και ένα άλλο στοιχείο που εν μέρει είχε αναφερθεί, έχουμε τις ίδιες διαδικασίες, ίδιες διαργασίες για εκείνους που απολάβουν διεθνούς προστασίας και εκείνους ε, που πιθανόν ε, δεν θα μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτή την κατηγορία και εδώ πρέπει να υπάρξει διαφοροποιημένη αντιμετώπιση ώστε να είμαστε επαρκή, να, να επαρκέσουμε στις διαφορετικές ανάγκες και άμεση μεταφορά μεταναστών από το σημείο αποβίβασης ε, στις, στα κέντρα της καταγραφής και καταχώρησής τους. Πολλές φορές το χρονικό διάστημα από την αποβίβαση μέχρι τη μετάβασή τους εκεί δεν επαρκεί για αυτή την καταγραφή. Πρέπει να ενημερώνονται καλύτερα οι μετανάστες για όλες αυτές τις διεργασίες και τις δυνατότητες μετεγκατάστασής τους. Η Frontex όπως ε, εξήγησα προηγούμενα και ο ρόλος ε, που έχουμε για την συνδρομή και υποστήριξη των Ιταλικών αρχών είναι η καταχώρηση, η ε, ε, δακτυλοσκόπηση, η φωτογράφηση, η δημιουργία της European Regional Task Force στην Κατάνια και οι Frontex και οι άλλες υπηρεσίες δρούν συνεργαζόμενες ε, στενότατα μεταξύ τους συντονίζοντας το έργο συνδρομής τους, ανταλλάσσοντας πληροφορίες, συμπεριλαμβάνοντας και στην ανταλλαγή αυτή πληροφοριών και την Euronav Σοφία ε, το πλαίσιο αυτό δράσης δηλαδή όσον αφορά και την καταπολέμηση των εγκληματικών δικτύων και των ε, διακινητών ε, ε, μεταναστών ε, και προσφύγων. Έτσι συνεχίζουμε με έντονο ρυθμό το έργο μας ως Frontex στις κοινέ αυτές δράσεις <clears throat> και θα συνεχίσουμε κατά τους επόμενους μήνες και κατά το 2016. Ευχαριστώ. Τώρα έχουμε την κυρία Διδιάνα Βαλάστρο που εκπροσωπεί το Save the Children της Ιταλίας για πέντε λεπτά. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ εξ ονόματος του Save the Children και θα ήθελα να σας, πω δύο λόγια σχετικά με τα όσα κάνουμε στην Λαμπεντούζα, στο κέντρο υποδοχής της Λαμπεντούζα. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο μας και βοηθούμε στην ταυτοποίηση των ανηλίκων, κυρίως ε, των ε, ανηλίκων των ασυνόδευτων και προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες της υποδοχής ε, θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό να μας δοθεί, που μας δόθηκε η δυνατότητα ε, να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε και να υποδεχόμαστε τους ε, νέους, τα παιδιά τα οποία βρίσκονται σε αυτό το κέντρο. ε, αμέσως μετά την άφηξή τους ε, οι μετανάστες ε, μοιράζονται σύμφωνα με την εθνικότητά τους ε, και σε, με συγκεκριμένο τρόπο γίνεται προσπάθεια να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να ενταχθούν στη διαδικασία της relocation. Επίσης, ελέγχουμε τις ε, αποφάσεις ε, επαναπροώθησης ε, που αφορούν όσους έχουν φτάσει στο νησί. Εμείς ε, υπάρχουν δυσκολίες τις οποίες ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να ε, ε, περάσουμε. Βεβαίως εμείς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και τις εντάσεις που δημιουργούνται μεταξύ κυρίως των Σομαλών και των Ερυθρέων γιατί οι προερχόμενοι από την Σομαλία δεν, ε, είναι, δεν εντάσσονται στη διαδικασία relocation. Και μέχρι τώρα αυτό έχει δημιουργήσει εντάσεις και τριβές, κυρίως ανάμεσα σε αυτές τις δύο εθνικότητες. Ε, ε, εκτός από τις δυσκολίες λοιπόν αυτής της διαδικασίας, ε, έχουμε και την δυσκολία ότι δεν έχουμε αρκετούς ενδιάμεσους ε, έτσι ώστε να δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες ε, στους μετανάστες και έχουμε και μετανάστες από την Νιγηρία Ε, και χρειαζόμαστε τους ενδιάμεσους έτσι ώστε να καταλάβουμε ποια είναι τα άτομα ε, τα οποία προερχόνται από την Ιγυρία και που έχουν μεγαλύτερα και που είναι πιο ε, πιθανόν να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, ε, σε πολλές περιπτώσεις ε, να έχουμε ικανοποιητικές και σε βάθος προσωπικές συνεντεύξεις στα πλαίσια του Υπουργείου Εσωτερικών διαπιστώνουμε επίσης κάποιες ελλείψεις όσον αφορά μια διαδικασία η οποία να συμπεριλαμβάνει στη διαδικασία relocation και τους ανηλίκους γιατί πολύ συχνά υποχρεώνονται οι ε, ανήλικοι να συνοδεύονται από ενηλίκους που δεν είναι όμως η φυσική τους ε, ε, συνοδη. Θα πρέπει να υπάρξει ε, ε, προσωπικό που να γνωρίζει και να είναι εξειδικευμένο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και σας όπως και τους υπόλοιπους ομιλητές. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε πάρα πολύ μακρύ κατάλογο ομιλητών. Παρακαλώ να μην ξεπεράσετε τα δύο λεπτά. Θα ξεκινήσω από την Μπάρμπαρα Κοντζίκα του ΕΛΚ. Μπάρμπαρα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την περιεκτική παρουσίαση. Ουσιαστικά δύο ερωτήσεις θα είχα. Η πρώτη ερώτηση προς τους εκπροσώπους από πλευράς της ε, Ιταλίας. Τι συμβαίνει ακριβώς, πώς έχει η δομή σε σχέση με τους πρόσφυγες, Ποιοι, τι άνθρωποι είναι αυτοί, πρόκειται για νέους ανθρώπους είναι κυρίως γυναίκες και παιδιά μεταξύ αυτών. Έχετε κάποια ποσοστά να μας δώσετε πόσα είναι τα παιδιά, πόσα, πόσες είναι οι οικογένειες, πόσες είναι και οι γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες τους και με παιδιά ίσως. Δεύτερη ερώτησή μου έχει ως εξή. Η Ιταλική κυβέρνηση στην αρχή είχε αναφέρει ότι υψηλός αριθμός συνοριοφυλάκων θα θα ασχολούντουσαν με την, ε, τα θέματα της μεταναστευτικής κρίσης ε, και θα μετετίθεντο. Αυτό ακούσαμε και από τους εκπροσώπους της Frontex. Τώρα θα θέλαμε να γνωρίζουμε αν ο αριθμός των συνοριοφυλάκων από πλευράς Ιταλίας που τώρα εμπλέκονται σε αυτή την κατάσταση ανταποκρίνονται στα όσα υποσχέθηκε ή είχε αναφέρει ότι θα έκανε η Ιταλική κυβέρνηση. Είναι λιγότεροι, όχι και γιατί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα αυτά τα οποία οι Ιταλοί εκπρόσωποι εδώ ανέφεραν και φυσικά ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο βέβαια σίγουρα. Σε σχέση τώρα με μια πτυχή της κατάστασης εδώ που έχει τεράστια σπουδαιότητα για πολλούς από εμά ευρωβουλευτές εδώ στην Ευρωβουλή όταν έρχεται η ώρα του να υπάρχει η κοινοποίηση αυτών των αντιδράσεων και δράσεων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων εν ώψη της προσφυγικής κρίσης όπως την αποκαλούμε. Έχουμε εδώ ένα νέο τεράστιο πρόβλημα επικοινωνίας. Τα hot spots τα αντιμετωπίζουν πολύ γύρω μας ως ένα είδος αντίδρασης που κυρίως στοχεύει στην προσέγγιση της διασφάλισης της ψυχής της ασφάλειας, των θεμάτων ασφάλειας κυρίως. Θα ήθελα ως προς αυτό να έχω λεπτομερείς πληροφορίες για τα πρωτόκολλα τα οποία υπεγράφησαν από τις Ιταλικές αρχές για την χρήση βίας. Πώς ε, οι αρχές, ε, οι δυνάμεις ασφαλείας εμπλέκονται και με ποιο τρόπο στα hot spots. Πώς ε, μπορούν, πώς η βία, η, η κρατική βία δρά σε σχέση με απειλούμενες καταστάσεις ή απειλές που διαμορφώνονται. Και δεύτερον, πώς υπάρχει, έχει συμφωνηθεί να λειτουργεί η συνεισφορά ή η συμμετοχή με άλλα λόγια των ΜΚΟ, των μη κυβερνητικών οργανώσεων ιδιαίτερα όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων εκείνων που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι και την προστασία των δικαιωμάτων τους. Ακούσαμε από αρμόδιες μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις σε σχέση με τα παιδιά και τα ανήλικα ότι τα παιδιά ακριβώς είναι η πιο ευάλωτη ομάδα, η πιο ο πιο ευάλωτος στόχος, η πιο ευάλωτη ομάδα πληθυσμιακά και πρέπει ξεχωριστά να μπορούν να αντιμετωπίζονται μέσα στο πλαίσιο των hot spots, μέσα σε αυτή την διοργάνωση εντό εισαγωγικών. Θα ήθελα να ξέρω πώς έχει η συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων που εμπλέκονται για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων που είναι τα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ για τους ε, συντηρητικούς, κυρία Στίβενς. Ο κύριος Στίβεν, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω και εγώ μια παρόμοια ερώτηση που είχα και για την ε, κατάσταση στην Ελλάδα. Αν και γνωρίζω πως υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε Ιταλία και σε Ελλάδα. Η Σαρδινία είναι ένα ε, νησία από τα οποία μπορούν πιο εύκολα να πάνε ε, στην ε, κυρίως Ιταλία. Υπάρχουν και πιο μακρινά νησιά. Θα ήθελα λοιπόν να επαναλάβω την ερώτηση που έκανα και πιο πριν. Η κατάσταση στην Ιταλία έχει ως εξής. Οι περισσότεροι που καταγράφονται έχουν γίνει κατάλληλες Έρευνε για να διαπιστωθεί αν προέρχονται από τη Συρία, από το Ιράκ, το Αφγανιστάν ή από κάποια άλλη χώρα. Υπάρχει ε, κάποια διαδικασία για να ε, διαπιστωθεί αν πρόκειται για πρόσφυγες ή για μετανάστες. Η διαδικασία καταγραφής έχουμε δει πως εφαρμόζεται και σε γενικές γραμμές λειτουργεί. Όμως αυτές οι έρευνες, αυτά τα screening που γίνονται πρέπει να έχουν και αποτέλεσμα, διότι διαφορετικά πιστεύω πως δεν υπάρχει νόημα σε αυτών των hot spot από τη στιγμή δηλαδή που καταγράφονται τι γίνεται μετά. Μπορούν να φύγουν, να συνεχίσουν μέχρι να φτάσουν εκεί που θέλουν, τι γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Αντζέλικα, μια για τους ε, φιλελεύθερους. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και την εκπρόσωπο του Save the Children που είναι εδώ ε, στο βιντεοδιάσκεψη. Στην συνάντηση στη Λαμπεντούσα και με εντυπωσίασε πάρα πολύ η δουλειά της. Η ερώτηση που έχω εγώ προς ε, εσάς έχει να κάνει με την κράτηση των ε, τον άσυλο. Μπορώ να σας πω ότι από την οπτική γωνία της Αυστρίας υπάρχει η δυνατότητα κράτησης των ανθρώπων μέχρι 48 ώρες. Μίλησα με τις αστυνομικές αρχές και μου είπαν ότι δεν ε, θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο διότι η αίτηση ασύλου δεν, ε, δεν αποτελεί έγκλημα και μάλιστα η κράτηση αποτελεί τεράστιο πρόβλημα διοικητικό, ε, οικονομικό και οι αστυνομικές αρχές δεν βλέπουν την ανάγκη κράτησης ανθρώπων οι οποίοι απλά ζητούν άσυλο. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω την άποψή σας γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Η Μαρή Κριστίν Βερζιά έχει το λόγο για την ΚΟΕ. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Συμφωνούμε όλοι ότι η Ιταλία δεν βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με την Ελλάδα. Δεν είναι ούτε στην ίδια κατάσταση σε σχέση με το ε, καλέ, αλλά πάντως ε, ε, βρίσκεται πάντα υποπίεση και βεβαίως έχει και σχετική εμπειρία γιατί εδώ και πολύ καιρό αντιμετωπίζει αυτήν την αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Πώς αναλύεται λοιπόν την εξέλιξη των ροών κυρίως σε σχέση με την αύξηση των παιδιών και των ανηλίκων ε, που έχετε ε, που έχει τευτοποιηθεί και σημειώνεται από τις περισσότερες ε, ΜΚΟ το θέμα αυτών των, ε, της, του χειρισμού, επιτρέψτε μου την έκφραση, των ε, ανηλίκων, ε, γιατί πολλές ΜΚΟ μας λένε ότι αυτοί οι ανηλικοί ταυτοποιούνται ως ενήλικες και δεν ακολουθούνται ας πούμε οι διαδικασίες όλες για τον καθορισμό της υγείας, της ηλικίας συγγνώμη ε, εμείς έχουμε μια παρακρά παράδοση με αυτές ε, τις ε, ταυτοποιήσεις στη Γαλλία. Πεςτε μου λοιπόν τι γίνεται στην Ιταλία. Επίσης, γενικά για την ταυτοποίηση, αυτό το ζήτημα της διαλογής ανάμεσα στους καλούς μετανάστες που συνήθως είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν ε, να ε, ε, πάνε σε ένα σύστημα relocation, αλλά τι γίνεται με τους άλλους, με ποιο τρόπο μπορούν να υποβάλουν το αίτημα, αυτοί που δεν εμπίπτουν σε αυτούς που κατά 75% γίνονται δεκτοί, εμπίπτουν στα κριτήρια όλων των χωρών. Επίσης λέτε ότι δεν είναι γρήγοροι ε, η ε, ε, ανταπόκριση και βεβαίως η ανταπόκριση οποιαδήποτε θα γίνει μετά από την πρώτη διαλογή από την αστυνομία αυτό μας προβληματίζει λίγο και επίσης όσον αφορά τις επιστροφές θα ήθελα εδώ να το υπογραμμίσω γιατί μας ανεφέρθη η περίπτωση μιας γυναίκας από την Ιγυρία η οποία φαίνεται ότι ε, ε, εστάλει ξανά στην Νιγηρία ενώ ήταν, είχε υποστεί τράφικινγκ και σε μερικές μέρες ε, την ξαναστήλατε στην Νιγηρία. Αυτό δεν μου φαίνεται πολύ ικανοποιητικό όσον αφορά την αναπερίπτωση αντιμετώπιση. θα πρέπει ε, όσο γίνονται στην Ιταλία να συνδυάζονται ε, με το ευρωπαϊκό δίκαιο και βεβαίως ε, με τις διαδικασίες για τους πρόσφυγες και θα πρέπει και οι περιπτώσεις των προσφύγων να αντιμετωπίζονται ανά περίπτωση όπως λέει η νομοθεσία και όχι ανά εθνικότητα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους σας και ευχαριστώ όλους όσοι πήραν το λόγο. Όσον αφορά τις διαδικασίες ταυτοποίησης, ε, οι άλλες χώρες εξακολουθούν να μας ε, ψέγουν ε, γιατί δεν κάνουμε καλά την καταγραφή και την ταυτοποίηση των μεταναστών. Μίλησα με στονούς βουλευτές που εξακολουθούσαν να θεωρούν την Ιταλία σαν ε, μια χώρα γεμάτου, γεμάτη πονηρούλιδες οι οποίοι δεν καταγράφουν καλά τους πρόσφυγες και τους αφήνουν να φύγουν προς τη Γερμανία. Θα ήθελα λοιπόν να καταλάβω εάν με τη δημιουργία αυτών των hot spots βελτιώνεται πραγματικά η κατάσταση. Αναφέρομαι πρωτίστως στο εξή. Ε, στη Ρέτζο Καλάμπρια ε, κατέβηκαν 990 πρόσφυγες από την Βόρεια Αφρική. Δεν ξέρω μεταξύ αυτών πόσοι ήταν οι ανήλικοι, αλλά αυτοί ε, οι 905 πώς ε, φτάνουν, ε, ε, πώς γίνεται ακόμα και σε περιόδους όπως τώρα που, το, που είναι χειμώνας και που θα έπρεπε κανονικά να έχει καμφθεί αυτή η μεγάλη, αυτός ο μεγάλος αριθμός αφήξεων ε, τι, τι γίνεται, γίνονται άμεσα οι ταυτοποιήσεις ε, με φωτογραφίες, ε, με λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, γιατί μας έχει αναφερθεί ότι ακόμα και στις μεταφορές φαίνεται ότι εξαφανίζονται κάποιοι, φεύγουν κάποιοι και κυρίως μας απασχολεί όσον αφορά τους ασυνόδευτους ανηλίκους στην Ιταλία έχουμε ένα πάρα πολύ σωστό ασυνόδευτο των που εξαφανίζονται. Θα ήθελα λοιπόν να καταλάβω ποια είναι η στρατηγική κυδαιμονίας και προστασία την οποία έχετε σκεφτεί κυρίως όσον αφορά αυτήν την ιδιαίτερη κατηγορία ιδιαίτερα τροτών ε, ε, πολιτών. Θα ήθελα επίσης ε, να κάνω άλλη μία ερώτηση. Έγινε λόγο στο πρόγραμμα Presidium. Θα ήθελα να μου πείτε ε, οι σηματοδοτήσεις που στέλνονται, οι σημάνσεις μάλλον που στέλνονται στο Υπουργείο Ιστορικών, ε, ποια συνέχεια δίνονται ε, αυτές οι σημάνσεις μετά από επισκέψεις στα κέντρα. Έχουν παραμείνει κενό γράμμα ή έχει υπάρξει μια συνέχεια που έχει δοθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα να καταλάβω λίγο καλύτερα από τον ε, κύριο Μορκόνε τι γίνεται μετά από την καταχώρηση στα hot spot τα οποία ε, είτε υπάρχουν είτε πρόκειται ε, να δημιουργηθούν. Πήγα λοιπόν εγώ στο τσία του Πόντε Γκαλέβια ε, εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί Νιγηριανοί. Είδαμε λοιπόν ότι όταν φτάνουν τα άτομα αυτά δεν έχουν πληροφόρηση σωστή για τα δικαιώματά τους ε, μεταξύ των οποίων και το δικαίωμα αιτήματο ε, διεθνούς προστασίας. Ε, δηλαδή γίνεται ένα μπέρδεμα ανάμεσα στην κατηγορία 2 που είναι η παράνομη ε, με την κατηγορία των, των ε, υποκείμενων σε relocation. Ξεχνάμε όμως ότι το το δικαίωμα στο άσυλο είναι ένα δικαίωμα γενικό, δεν είναι ένα ε, ε, ε, δεν είναι κάτι το οποίο υπόκειται στις διάφορες εθνικότητες. Στο Πόντε Γκαλέρια είδαμε και νέους, μικρά ανθρώπους που δεν είναι συνοδευόμενοι και μάλιστα και βάσει της νομοθεσίας και συγκεκριμένα του νόμου 142 του Σεπτεμβρίου του 9 μπορούν να, διατηρη... να κρατηθούν μονάχα για 90 ημέρες ε, και μάλιστα καταλαβαίνετε ότι σε αυτά τα κέντρα τώρα που είναι χειμώνας τα κέντρα αυτά δεν έχουν ζεστό νερό δεν ε, ε, οι χώροι δεν είναι καλοί, σπασμένα μπάνια κτλ. δεν είναι δυνατόν οι ανήλικοι να μένουν σε τέτοιες συνθήκες. Ο υπολογισμός της ηλικία φαίνεται ότι δεν γίνεται με το σωστό τρόπο και διακινδυνεύουμε να υπάρχουν νέοι ανήλικοι οι οποίοι να μένουν σε αυτές τις δομές. Αλλά εν πάση περιπτώσει και σε αυτές τις δομές δεν είναι δυνατόν όλοι να έχουν τον ίδιο δικηγόρο ο οποίος ε, εξ οφίτσιο ε, ορίζεται. Τέλος, ε, ήθελα να πω ότι συμφωνώ ότι αυτά, αυτές οι προϋποθέσεις είναι παράλογες. Το πρόγραμμα της relocation θα έπρεπε να έχει ήδη ξεκινήσει χωρίς αυτές τις ε, προϋποθέσεις που βαραίνουν την Ιταλία αλλά και την Ελλάδα, δηλαδή πρώτα να φύγουν από τα hot spots αυτοί που είναι του 75% και μετά. Ε, ή μιλάμε για ελληνική ευρωπαϊκή ή δεν μιλάμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη γιατί δεν ήμουν παρούσα από την αρχή, ζητώ συγγνώμη από τους εισηγητές, αλλά δυστυχώς Ταυτόχρονα ε, είχα και μια άλλη επιτροπή. Ε, ευχαριστώ πολύ γιατί ξέρω ότι κάνατε μία πολύ σε βάθος σκέψη και από διάφορες οπτικές γωνίες ε, του θέματος της μετανάστευσης. Πολύ σύντομα θα ήθελα να κάνω δύο-τρεις ερωτήσεις. Ε, ξέρουμε ότι συνεχίζει η μεταναστευτική ροή και γνωρίζουμε και ξέρω για την Ιταλία ότι την προηγούμενη εβδομάδα, τις τελευταίες μέρες, 4.000 ε, άνθρωποι φτάσανε στις ακτές μας και φυσικά δεν έχουμε κανένα σημάδι που να μας λέει ότι στο μέλλον θα αλλάξει η ροή, θα μειωθεί η ροή στο εγγύς μέλλον. Ήθελα λοιπόν να υποβάλω ένα πρώτο γενικό ε, ε, ερώτημα προς την Κομισιόν. Μπορούμε να σκεφτούμε τώρα υπό το φως των αποτελεσμάτων της εργασίας που έγινε τους τελευταίους μήνες, μπορούμε λέω να θεωρήσουμε ότι γνωρίζουμε καλά την ε, πραγματικότητα του φαινομένου της μετανάστευσης, διαστάσεις που έχει το φαινόμενο αυτό ε, έχουμε την εντύπωση ότι έχει υπάρξει σωστή ευαισθησία ε, από όλες τις χώρες και ότι ελήφθησαν όλα τα πλέον δόκιμα μέτρα έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό και τι ακόμα μπορούμε να σκεφτούμε ε, να εφαρμόσουμε. Ε, ε, έχοντας σαν πρότυπο βεβαίως ε, τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Αυτή ήταν η μία ερώτηση. Ερώτηση για την συνεργασία, την πλήρη συνεργασία των υπηρεσιών, κυρίως συνεργασία μεταξύ της Europol και της Frontex. πού ακριβώς θα επικεντρωθεί αυτή η συνεργασία. Και η Eurojust ζήτησε να ενταχθεί στο θεματολόγιο της ε, μετανάστευσης έτσι ώστε να συμβάλλει στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα, το, τον αντίκτυπο που αυτές οι ροές έχουν. Πώς θα γίνει αυτή η συνεργασία μεταξύ Frontex, Eurojust και τέλος ένα άλλο θέμα το οποίο μου είναι ιδιαίτερος προσφυλές και που αφορά, αφορά τους ε, ανηλίκους. Ε, ξέρουμε ότι ένα τέταρτο των μεταναστών είναι ε, ανήλικοι. Ξέρουμε ότι αυξάνεται ο αριθμός των συνόδευτων ανηλίκων και ε, μονάχα στην ε, Σουηδία μέχρι τώρα έχουν διπλασιαστεί ε, οι αιτήσει ασύλου μέχρι τώρα δηλαδή έχουν διπλασιαστεί οι αιτήσει σε σχέση με ολόκληρη τη χρονιά του 2014. Τι γίνεται λοιπόν στα hot spots για να στηριχτούν οι ανήλικοι, οι ασυνόδευτοι, αλλά ε, και κάτι άλλο το οποίο γνωρίζει πολύ καλά η οργάνωση Save the Children, δηλαδή αυτή η αόρατη ανήλικη. αυτοί για τους οποίους δεν γνωρίζουμε τίποτα, δεν ξέρουμε που βρίσκεται και που ε, πραγματικά διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο και είναι αντιμέτωποι με δραματικές καταστάσεις δυστυχώς. Ε, η Save the Children και αναρωτιέμαι αν κάτι τέτοιο είναι δυνατόν, είχε σκεφτεί ε, να δοθεί ένα ποσοστό της relocation σε αυτούς ε, τους ε, ε, τους ανήλικους. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα και τέτοια πιθανότητα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Άννα Γκόμες παρακαλώ τελευταία. Τουλάχιστον 1,5 hot spot φαίνεται ότι έχουμε. Ένα στην Λαμπεντούζα και μισό κοντά εκεί. Ωστόσο λειτουργεί αυτό στη Λαμπεντούζα και μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία επανεγκατάστασης ε, προσφύγων διότι και πάλι έχουμε το πρόβλημα στην Πορτογαλία εδώ με το παράπονο ότι δεν φτάνουν λέει οι μετανάστες οι πρόσφυγες ε, όπως θα έπρεπε από την ε, χώρα εκείνη που θα έπρεπε να προέλθουν. Τώρα στην περίπτωση των παιδιών και των ασυνόδευτων ανηλίκων θα ήθελα να γνωρίζω ιδιαίτερα αν η UNICEF το Save the, Save the Children ή άλλος οργανισμός έχουν κάποιο σύστημα αρρωγής για να παρακολουθούν τα παιδιά που μετεγκαθίστανται, ώστε να μην εξαφανίζονται αυτά τα παιδιά, να διασφαλίζουμε ότι θα τα παρακολουθούν όταν κάπου μετεγκαθίστανται. Και τέλος όσον αφορά την διαδικασία επεξεργασίας, την εξέταση δηλαδή των ετοιμάτων χορήγησης ασύλου. Σε ποιο βαθμό αυτό αποτελεί και ένα βάση της, με εθνικότητα ώστε να μην εγκρίνονται κάποια αιτήματα διότι στην Βαλέτα στη Σύνοδο Κορυφής ακούστηκαν πολλά και διάφορα. Γνωρίζουμε όμως ότι εκείνοι που προέρχονται από την Ερυθρέα και την Αιθιοπία ουσιαστικά ξε, προσπαθούν να ξεφύγουν από ένα κατασταλτικό καταπιεστικό καθεστώς. Αυτό τώρα τι θα σημαίνει. Δεν θα έχουν δικαίωμα να τύχουν έγκριση οι αιτήσει τους ε, από την Αιθιοπία ή την Ερυθρέα όταν ζητούν άσυλο. Και μετά την καταπολέμηση των δικτύων μαζί με την Euronavforce ε, Σοφία Ποια είναι η αξιολόγηση ώστε να μπορούν οι ε, διακινητές πραγματικά να καταπολεμηθούν ο σωστός τρόπος δεν θα ήταν να υπάρχουν ε, ασφαλείς διάβλοι και ασφαλείς λεωφόροι και διαδρομές για τους μετανάστες και πρόσφυγες ώστε να βρίσκονται σε ένα καθεστώς ασφάλειας και να μην τους αφήνουμε σε ένα ελάχιστο επίπεδο όσον αφορά την αντιμετώπιση των διακινητών και των δουλεμπόρων όταν βλέπουμε ότι το κέρδος είναι εκείνο το οποίο διατηρεί αυτό το εμπόριο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακέ οι ερωτήσεις. Και τώρα έχετε το δύσκολο έργο εσείς ε, να μπορέσετε να τοποθετηθείτε και να απαντήσετε και στα θέματα εμπορίας και στα θέματα ανηλίκων και ασυνόδευτων παιδιών και σε σχέση με την κατεπίγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των θεμάτων εμπορίας, εμπορίας γυναικών και ανθρώπων. Και εδώ ίσως θα μπορούσατε να προσπαθήσετε να απαντήσετε με, υπό τους όρους αριθμών πώς αυτό έχει επίπτωση στο έργο hotspots και αυτό το πολύ επιθετικό πλαίσιο των εμπόρων και διακινητών των μεταναστών και προσφύγων ιδιαίτερα όσον αφορά τα ανήλικα παιδιά διότι πραγματικά αυτό είναι μια κατάσταση κατεπίγουσα, κατεπίγουσας ανάγκης που πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα οπωσδήποτε. Λοιπόν, ξεκινούμε με τον Λόρα Μισελ, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μια που αρχίσατε αναφέροντας τους ανήλικους, θα σας δώσω μερικά δεδομένα και στατιστικά στοιχεία από τον Ιανουάριο μέχρι τέλειο Οκτωβρίου. Είχαμε λοιπόν έξι σχεδόν 20.900 γυναίκες, 60.000 άντρες, 40.000 ανήλικους. «15.000 ήταν οι ανήλικοι, μάλλον από τον Ιάριο μέχρι τον Οκτώβριο. Είναι λοιπόν αρκετά σοβαρό το πρόβλημα και νομίζω πως ε, θα μπορούσε να τοποθετηθεί και η εκπρόσωπος του Save the Children γι' αυτό. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες μόνο για τους αθηνόδευτους ανήλικους. Στη Λαμπεντούσα όμως ε, όντως υπάρχει πρόβλημα χωρητικότητας. Σχετικά με την ε, χρηματοδότηση, την έκτακτη χρηματοδότηση, υπάρχουν κονδύλια στην Ιταλία που προορίζονται συγκεκριμένα για τους ασυνόδευτους ανήλικους. Ε, Τώρα, ποιες είναι οι διαφορές ε, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία και αν υπάρχουν. Υπάρχουν διαφορές. Βλέπουμε αρκετούς ασυνόδευτους ανήλικου από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν που πηγαίνουν στα ελληνικά νησιά. Είναι δηλαδή ένα κοινό πρόβλημα στην Ελλάδα και στην Ιταλία αυτό. Ε, κυρία Βερζιά, μιλήσατε για την εξέλιξη των ε, μεταναστευτικών ροών εάν συγκρίνουμε αυτή τη χρονιά με την προηγούμενη, η μεγάλη ε, αλλαγή είναι η αλλαγή των ενηλίκων. Ε, είμαστε στις 160.000 ενώ τώρα βρισκόμαστε ήδη στις 150.000. Ε, την Προηγούμενη χρονιά είχαμε πολλούς από την ε, Ερυθρέα, ενώ τώρα έχουμε περισσότερους από τη Δυτική Αφρική, έχουμε από τη Γάμπια, από την ε, ε, Σενεγάλη, από την Νιγηρία, καθώς επίσης και από την ακτή του Ελεφαντοστού. Ε, η διαφορά είναι, συγγνώμη, ότι δεν έχουμε τόσους ε, σύρους. Ε, ενώ στην Ελλάδα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Επίσης, εάν κλείσουν τα σύνορα ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Φύρωμα, τη Φύρωμα και τη Σερβία κτλ, η διαδρομή γίνεται πιο, πολύ πιο δύσκολη. Ίσως τότε μπορούμε να προβλέψουμε ότι κάποιοι σύροι θα φτάσουν στην ε, ε, Ιταλία είτε άμεσα από την Λιβύη είτε περνώντας από την Ελλάδα στην Αλβανία και από εκεί στην Ιταλία. Ένα σημείο σημαντικό είναι ότι συγχαίρεται το θέμα του ασύλου με το θέμα της ε, υπηκότητας δεν υπάρχουν κριτήρια ε, για την χορηγήση ασύλου. Υπάρχουν εθνικά κριτήρια, ε, κριτήρια μάλλον υπηκότητας για την ε, μετακατάσταση. Υπάρχουν κάποιες ε, χώρες, Ιράκ, Ερυθρέα, Συρία, οι οποίες είναι χώρες όπου στους πολίτες των οποίων χορηγείται άσυλο. Τώρα, αν προέρχεσαι από την Κάνα και ζητήσεις άσυλο, η περίπτωση αυτή θα εξεταστεί υπό άλλο νομικό πλαίσιο. Τώρα, αν θέλει κάποιος να κάνει αίτηση για το πρόγραμμα κατάσταση, αυτό είναι τελείως διαφορετική υπόθεση. Εμείς δεν αποφασίζουμε βασιζόμενοι μόνο ε, στην ε, εθνικότητα. Αν προέρχεται κάποιος από μια ασφαλή χώρα, τότε φυσικά και έχει αυτό ε, επιπτώσει στην απόφαση. Στην ε, Ιταλία όμως υπάρχουν εμπειρογνώμονες από την ΕΑΣΟ οι οποίοι αξιολογούν τις, την κάθε περίπτωση. σχετικά με την ερώτηση της κυρία Φερέρα για την Καλαβρία. Στην Καλαβρία δεν υπάρχει hot spot και είναι και μία από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτό έχουμε ζητήσει από την Ιταλία να δημιουργήσει περισσότερα τέτοια ε, hot spot και να μην περιοριστεί στην Λαμπεντούσα που έχει χωρητικότητα μόνο 500 ατόμων. Όταν ε, κάθε μέρα καταφτάνουν πολύ περισσότεροι δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό η Ιταλία. Χρειάζεται λοιπόν ε, άμεσα να δημιουργηθούν περισσότερα hotspot. Σας ευχαριστώ. Η εκπρόσωπος του Save the Children θα ε, πρέπει να φύγει πολύ σύντομα. Γι' αυτό λοιπόν κυρία Βελάστρο, αν δεν έχετε πρόβλημα και αν θέλετε να δοθούν απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, θα ε, χρειαστεί να περιμένετε μέχρι 5 λεπτά για να απαντήσει η εκπρόσωπος του Save the Children. Σας ευχαριστώ. Τρία σημεία. Πρώτον, τα στοιχεία τα οποία ο Δ. Μορκόνε μπορεί να ε, πει με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Τρί, δεύτερον, ε, η ταυτοποίηση. Τρίτον, ε, η απομάκρυνση ή εξαφάνιση των ε, ε, ανηλίκων. 15.000 περίπου είναι οι ανήλικοι που έφτασαν εδώ. Ε, το 1 τρίτο έφτασε με έναν ή δύο γονείς, ενώ τα δύο τρίτα μόνα τους. Μεταξύ των ε, ανσυνόδευτων οι περισσότεροι είναι από την ε, Ερυθρέα, 3.000, 1.000 από την Σομαλία και 1.700 από την Αίγυπτο οι προερχόμενοι από την Σομαλία και την Ερυθρέα θέλουν να πάνε σε άλλες χώρες και είναι ε, οι περισσότεροι από αυτούς τους νέους ε, αυτοί που εξαφανίζονται. Δηλαδή εξαφανίζονται με την έννοια ότι ε, πηγαίνουν να ζήσουν με φίλους και γνωστούς. Για να προβλέψουμε λοιπόν και να προλάβουμε αυτήν, αυτό το φαινόμενο ε, της ε, απομάκρυνσης και εξαφάνισης των νέων, ε, θα πρέπει τουλάχιστον τους νέους από την Ερυθρέα να τους ταυτοποιήσουμε άμεσα ε, για τους οποίους ε, να εφαρμοστεί άμεσα ο κανονισμός του Δουβλίνου. Ε, στην ουσία ένας χρόνος χρειάζεται βάση του Δουβλίνου έτσι ώστε ένας καθόλου επιλέξιμος νέος να ολοκληρώσει τις διαδικασίες και να πάνε προς μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι διατεθειμένοι να περιμένουν αυτό το χρόνο οι ανήλικοι και εξαφανίζονται λοιπόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σημαντικό και θεμελιώδους σημασία, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα ένα, κάποιο πρωτόκολλο που να λέει ακριβώς ποια είναι τα βήματα τα οποία θα πρέπει να αναλυθούν έτσι ώστε ε, να καταλάβουμε την πραγματική ηλικία ενός ε, νέου που δηλώνει ότι είναι ανήλικος. Υπάρχει στην Ιταλία ένα κείμενο το οποίο, ε, με το οποίο συμφωνούν και οι οργανώσεις αλλά και οι περιφέρειες. Αυτό το κείμενο θα πρέπει να εγκριθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα γιατί διαφορετικά θα συνεχιστεί αυτό που συμβαίνει τώρα στην Λαμπεντούζα και όπως ε, υπόθηκε άλλωστε δεν είναι σε θέση ε, η ε, πολιτεία να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία όσον αφορά το που βρίσκονται αυτοί οι νέοι, όσον αφορά τα θύματα του τράφικινγκ. Λείπουν θέσεις υποδοχής. Προσπαθούμε να ε, ε, βγάλουμε τα παιδιά αυτά από κυκλώματα σεξουαλικής κυρίως εκμετάλλευσης. Ωστόσο ε, δεν έχουμε μια ειδική αντιμετώπιση. Γι' αυτό ζητούμε και από την Πολιτεία και από την Ένωση μεγαλύτερη, σωστότερη αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Ευχαριστώ κύριος Μορκόνε. Ευχαριστώ. Αποσαφηνίζω κάτι για την ε, συνάδελφο που είπε για την εξαφάνιση των νέων. Ναι, συμφωνώ για, τους, για αυτά που είπε για τους ασυνόδευτους, αλλά ε, λυπούμε κάποιος που δουλεύει ε, ήδη από το 2007-2008 μαζί μας ε, να μιλάει για επαναπροωθήσεις. Δεν υπάρχουν επαναπροωθήσεις ε, ναι, υπάρχουν διατάξεις οι οποίες σε μερικές περιπτώσεις ε, ορίζουν ότι σε 7 ημέρες θα πρέπει να ε, εγκαταλείψει ο ενδιαφερόμενος το έδαφος της επικράτειας της χώρας. Αλλά δεν είναι όμως επαναπροωθήσεις αυτές. Ε, κοιτάξτε, εμείς συνεργαζόμαστε με την ύπατη ε, αρμοστία ε, των ε, προσφύγων και διασφαλίζονται πλήρως οι διαδικασίες όσον αφορά τους ετούντες άσυλο. Ε, ναι, θέλουμε να αλλάξει το σύστημα ε, του ασύλου, αλλά φυσικά οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι συνολικές, γιατί με αυτόν τον τρόπο, κατά τη δικιά μας άποψη, υπάρχει η ασφάλεια και η ισορροπία όσον αφορά τη διαδικασία ε, αιτήσεως ασύλου. Ε, επίσης, ε, μελλοντικά θα μπορούν να γίνονται οι ταυτοποιήσεις ε, με καταγραφή ταυτόχρονη σε, ε, σε δισκέτα και έτσι θα είναι μεγαλύτερη η διαφάνεια όσον αφορά τα σύνορα με τη Σλοβενία και την κατάσταση. ξέρω ότι οι σχέσεις μεταξύ αστυνομικών αρχών είναι πολύ καλές, αλλά δεν μπορούν από μόνες τους να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Κύριε Αγκουγιάρο. στην ε, Ιταλία εμείς πάντα προσέχουμε ε, τα δικαιώματα. Η χρήση της ε, βίας είναι πάντα αναλογική. Όντως υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις και σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις εμείς καταγράφουμε τα πάντα σε βίντεο έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαστής θα κληθεί ε, να ε, ε, ελέγξει την κατάσταση και το κατά πόσον οι αστυνομικές αρχές έχουν φερθεί σωστά να υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Από το 2006 δουλεύουμε με όλες τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες ούτως ή άλλως έχουν πρόσβαση σε όλα. Έχουμε εφαρμόσει πολιτική ανοιχτών θυρών. Αυτά. Ε, κυρία Στίβενς, ήρθα στις Βρυξέλλες για να σας συναντήσω σήμερα και είναι μεγάλη τιμή για μένα και σας ευχαριστώ. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι αντίθετα από το τι συμβαίνει σε διάφορες χώρες ή τι θεωρούν ε, χωρίς ε, λόγο άλλες χώρες, στην Ιταλία γίνεται καταγραφή των δακτυλικών αποτυπωμάτων όλων όσων φτάνουν στις ακτές μας. Ε, και ο Γενικός Γραμματέας ε, της, και ο υπεύθυνο της Γενικής Διεύθυνσης Home ξέρει πάρα πολύ καλά ότι όλα τα στοιχεία καταγράφονται στη Eurodac ε, πέρα από τους μύθους που ενδεχομένως ακούγονται για τη χώρα μου χώρα η οποία κάνει μια τεράστια προσπάθεια και αυτό απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη οργανωτική προσπάθεια. Κοιτάξτε, στην Ιταλία δεν υπάρχει ε, κράτηση για τους ετούντες άσυλο. Ε, εμείς δεν κρατούμε αυτούς τους ανθρώπους, τους βάζουμε απλώς σε μία αναμονή της ρύθμισής τους ε, σε κάποιο κέντρο. Ούτε καν μας περνάει από το μυαλό να θέσουμε σε συνθήκες περιοριστικής κράτησης τους ετούντες άσυλο. Απλώς καταχωρίζουμε τους ε, ξεχωρίζουμε μάλλον αυτούς που ενδεχομένως θα χρειαστεί να ε, ε, επιστρέψουμε στις χώρες τους. Όπως είπα κυρία Βλεβιά, είναι πολλοί νέοι από την Αίγυπτο που τους στέλνουν οι γονείς τους στην Ιταλία ε, γιατί τους στέλνουν οι ίδιοι οι γονείς, ε, τους νέους τους, τα παιδιά τους, γιατί θεωρούν ότι μόνο έτσι μπορεί λίγο το μέλλον τους ε, να βελτιωθεί. Είμαστε φίλες χώρες και επαναλαμβάνω ότι εμείς δεν στέλνουμε πουθενά, ποτέ αυτής της, αυτούς τους νέους. Ποτέ εμείς δεν κάνουμε ε, δεν, δεν ενδιαφερόμαστε παρά μόνο για το κυρίαρχο δικαίωμα των παιδιών ε, και μονάχα Προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε τα, τους ε, ε, νέους από τους οικογένειες και από τους ενήλικες ενώ εμείς, γιατί έχω δει να γίνεται αυτό το ανακάτεμα σε πολλές χώρες, εμείς στην Ιταλία τους ξεχωρίζουμε. Κυρία Φεράρα. Ε, πάλι αυτή όλη η ιστορία για τις ε, ταυτοποίησεις. Ε, εμείς έχουμε, τους ταυτοποιούμε όλους, τα ονόματα είναι εκεί, μπορείτε να τους ελέγξετε. Ακόμα και αυτή τη στιγμή στα στα σημεία απόβασης ε, ε, κάνουμε την ταυτοποίηση, όχι μονάχα στο περίφημο hot spot της Λαμπεντούζα που είναι πραγματικά ε, με πάρα πολύ μεγάλο βάρος, αλλά και σε όλα τα άλλα σημεία απόβασης η ταυτοποίηση γίνεται κανονικά. και ε, εμείς ε, το OEM, το Save the Children, ο Ερυθρός Σταυρός, ε, η ύπατη αρνημοστία, πάντα ήταν συνοδοιπόροι μας αυτό το δύσκολο δρόμο. Κυρία Σάιμ, το είπα και λίγο πριν και το ξαναλέω. Εμείς δουλεύουμε με την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των των μεταναστών. Κοιτάξτε, σας είπα ότι δεν υπάρχει επαναπροώθηση. Ε, εγώ, τουλάχιστον από όταν εγώ έχω αναλάβει την θέση του Διευθυντού, ε, υπάρχουν αποφάσεις απομάκρυνσης από την εθνική επικράτεια. Αυτό είναι διαφορετικό. Η συνεργασία με τις διάφορες υπηρεσίες είναι εξαιρετική. Με την ΕΑΣΟ δουλεύουμε και κατανοούμε ο ένας τον άλλον πολύ καλά. Δουλεύουμε χέρι με χέρι όσον αφορά ε, την Πορτογαλία, ναι, είχαμε κάποιες εγκρίσεις, αλλά η, πρώτη αποστολή θα γίνει στην Πορτογαλία. Ξέρω ότι οι Πορτογάλοι έχουν κάνει πάρα πολύ καλά δουλειά, έχουν, ε, καλή δουλειά, έχουν ετοιμάσει ε, ήδη κέντρα υποδοχής. Όσον αφορά τώρα το τράφικινγκ γυναικών από την Ιγυρία, είναι ένα περίπλοκο ζήτημα, το οποίο δεν μπορεί να λυθεί έτσι στο πόδι. Δουλεύουμε πάρα πολύ για το θέμα αυτό. δεν είναι ένα πρόβλημα των ε, ε, δομών υποδοχής. Ε, είναι ένα πολύ πιο περίπλοκο ζήτημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ε, βγάλουμε τις, τους, τα άτομα αυτά από το περιβάλλον στο οποίο έρχονται. κοιτάξτε, εμείς το άρθρο 18 το έχουμε δημιουργήσει εμείς και το ακολούθησε μετά η Ιταλία. Βεβαίως μπορεί και πρέπει να γίνει κάτι περισσότερο έτσι ώστε να καταφέρουμε να βγάλουμε αυτές τις γυναίκες, αυτές τις κοπέλες από τις συνθήκες υποτέλειας στις οποίες ε, σκλαβιά στην οποία ζουν. Δεν είναι εύκολο. Δουλεύουμε με μη κυβερνητικέ οργανώσεις, δουλεύουμε με κάθε δυνατό τρόπο. Δεν είναι αλήθεια ότι όλες αυτές οι γυναίκες ξαναστάλθηκαν στην Ιγυρία. Όχι. Πολλές έχουν σταλεί σε δομές στην κεντρική και βόρεια Ιταλία. Ορισμένες όντως επέστρεψαν στην αλλά αυτό μόνο όταν ο δικαστής ε, υπέγραψε μια σχετική απόφαση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ήδη υπερβεί ε, τα όρια αυτής της ε, συνεδρίασης. Δυστυχώς δεν μπορώ να δεχτώ άλλες ερωτήσεις, δεν μπορώ να δώσω σε κάποιον άλλο το λόγο. Ναι, αν μιλήσετε μόνο για 10 δευτερόλεπτα, εντάξει. Αλλά διαφορετικά δυστυχώ όχι. Έχετε 10 δευτερόλεπτα. Τώρα μιλήστε παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Λακωνικά. Ζητώ συγγνώμη γιατί έφτασα αργοπορημένα, γιατί ε, ε, έφτασε αργά το πλάνο μου. Ε, πόσες είναι οι, δι, οι συμφωνίες που έχει υπογράψει η Ιταλία, τέσσερις από ό,τι φαίνεται όσον αφορά τους επαναπατρισμούς. Ε, μήπως όμως αυτό είναι μια ανομαλία του συστήματος έτσι ώστε ε, να ε, επιτρέψει αυτές τις ε, Αίγυπτος, Μαρόκο, την Ισία και Νιγηρία. Αυτές είναι οι συμφωνίες επαναπροώθησης που έχουμε υπογράψει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουμε ζητήσει από την Κομισιόν ακριβώς να ε, βοηθήσει παρεμβάσεις επαναπροώθησης ε, που αφορούν όλες τις ε, χώρες έτσι ώστε να γίνονται επαναπροωθήσεις και μέσω της, με τη βοήθεια της Frontex. Μάλιστα. Θα ήθελα να πω στον κύριο Σέμπρη και κύριο Ρόσλερ ή θέλετε να προσθέσετε κάτι. Κύριε Ρόσλερ πολύ σύντομα. Ξέρω πώς θα τα καταφέρετε. Σας ευχαριστώ. Σχετικά με την συνεργασία ανάμεσα σε γύρω πολλέ και Frontex, υπάρχει ένα στρατηγικός διακανονισμός συνεργασίας, ο οποίος υπεγράφεται την περασμένη Παρασκευή και διευρύνει το ε, πεδίο εφαρμογής ε, Τη συνεργασία και διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών για προσωπικά δεδομένα. Αυτό είναι κάτι καινούριο. Είναι δεδομένα τα οποία μπορεί να επεξεργαστεί η Frontex και να αποστείλει στην Europol. Ε, στα πλαίσια αυτή της διευρυμένης συνεργασίας είναι επίσης και η πρόσκληση της ε, Ευρωπόλ να συνεργαστεί σε κοινέ επιχειρήσεις με την Frontex ε, στα πλαίσια συνεργασίας και με την ε, Eurosur έτσι ώστε να παρέχει περισσότερο αναλυτικές πληροφορίες και να συνεργαστεί για την ανάπτυξη του ετήσιου κοινού προγράμματος εργασίας. Αυτό είναι το πεδίο εφαρμογής. Κύριε Σέμπρη, κλείστε παρακαλώ. Ναι, σχετικά με τους ε, ασυνόδευτους ανήλικους και το αν ε, έχουν προτεραιότητα οι αιτήσει τους. Καταρχάς πρέπει να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στην πρώτη καταγραφή και εκείνη που γίνεται στην διαδικασία αίτησης ασύλου. Υπήρχε και μία ερώτηση, αν δεν κάνω λάθος, για το ποιος ελέγχει την κατάσταση. Ναι, υπάρχει έλεγχος της κατάστασης του ασύλου, γι' αυτό έχουμε και έναν μηχανισμό ετοιμότητας, σε λειτουργία, όμως δεν έχουμε κάποια μαγική σφαίρα ε, στην οποία μπορούμε να δούμε τα πάντα. Δεν μπορούμε να ε, σας πούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους συμμετέχοντες ε, για τα δύο πάνελ και το επιτελείο τους και να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη της Επιστροπής που έκαναν πολύ ενδιαφέρουσες και κέρυες ερωτήσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ για το ότι εσείς οι ευρωβουλευτές ζητήσατε να γίνει μια έκτακτη συνεδρίαση. Πιστεύω πως ήταν το κατάλληλο ε, το καταλληλότερο που μπορούσαμε να κάνουμε και σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και την εκπρόσωπο του Save the Children. Είστε ελεύθεροι, μπορείτε να φύγετε.